Ja, liebe Kolleginnen Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία ξεκίνησε χτες, όλο ε, ημερή συνεδρίαση χτες ε, και συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα. Χαίρομαι ιδιαίτερως που σήμερα έχουμε έτσι νωρίς νωρίς μαζί μας ε, και μάλιστα στην πρώτη συνεδρίαση του έτους τον Επιτροπό Γεωργίας. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην Επιτροπή Γεωργίας. Και προφανώς ανυπομονούμε να ακούσουμε τις απόψεις σας για τις μεγάλες αυτές ε, αποφάσεις τις οποίες καλούμαστε να λάβουμε φέτος και σε χρηματοοικονομικό επίπεδο που είμαστε στην πλευρά σα. Είναι σαφέ και θέλουμε να είναι εκτενή ο προπολογισμό για τη γεωργία, να μην γίνουν περικοπέ και σε ό,τι αφορά την ήδη σε φάση μεταρρύθμιση σε πολιτική γεωργία, προκειμένου να καταλήξουμε τελικά σε καλέ αποφάσει, σε ένα καλό και εύλογο συμβασμό. Γι' αυτό λοιπόν θα χρειαστεί εντατική συνεργασία μεταξύ ημών και ημών και διαρκεί επαφή προ την κατεύθυνση αυτή για να ανταλλάσσουμε απόψει. Χαιρόμαστε λοιπόν που σε τέτοιο ε, έγκυρο σημείο έρχεστε στην Επιτροπή μας. Χθες έγινε ήδη μια ανταλλαγή απόψεων. Έχουμε και την στρατηγική Farm to Fork από το αγρόκτημα στο πιάτο. Και φυσικά οι αγρότες ε, έχουν ε, παρακολουθούν το θέμα αυτό με ε, μεγάλο ενδιαφέρον και φυσικά θα και το θέμα του ποιε θα είναι οι συνέπειε τη ε, μεταρρύθμιση αυτή στην γεωργική πολιτική και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Μα ενδιαφέρουν λοιπόν όλα αυτά τα σημεία. Γι' αυτό λοιπόν θα σα δώσω πάρα αυτά το λόγο για 15 λεπτά να κάνετε μία εισαγωγή και μετά θα κάνουμε ένα γύρο των συντονιστών. Ο καθένα θα έχει το λόγο για δύο λεπτά και στη συνέχεια θα ακούσουμε και του άλλου συναδέλφου για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι εδώ τόσο σύντομα στην Επιτροπή σας. Οι επαφές αυτές, αυτές οι συναντήσεις ε, και αυτή η μόνιμη επαφή με την Επιτροπή σας ε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Συνήθως ε, η πρώτη έκθεση γίνεται μετά από 100 ημέρες. Εγώ ε, έχω 15, 50 ημέρες συγγνώμη, που έχω αναλάβει καθήκοντα. Υπάρχουν κάποια σημαντικά ζητήματα και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να τα συζητήσουμε ήδη από τώρα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γνωρίζουμε, διότι το Κοινοβούλιο ασχολήθηκε με το θέμα αυτό ήδη από τις πρώτες εβδομάδες που ανέλαβε καθήκοντα η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα είναι το Green Deal. Υπήρξε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, υπάρχει ένα πάρα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα για προκλήσεις, ε, στόχους και κλιματική ουδετερότητα και υπάρχει και μεγάλη ε, σειρά δεσμεύσεων που απορρέουν από την συμφωνία. Ε, αυτή είναι και ε, η πλευρά που αφορά τη γεωργία. Η γεωργία είναι απόσπαστο τμήμα ε, όλου του Green Deal. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις που περιμένουν την ευρωπαϊκή γεωργία και αυτό δημιουργεί φυσικά και ε, λόγους ανησυχίας. Είχα και μια σειρά συναντήσεων διότι η κυρία Φοντερ μου ζήτησε να συναντηθώ με όλα τα κράτη-μέλη ήδη μέχρι το μέσον ε, της θητείας μου. Έχω ήδη επισκεφθεί τέσσερις χώρες, μπορεί λοιπόν να τα έχω καταφέρει και νωρίτερα ε, από το μέσο της θητείας. Πήγα στην Κροατία, αυτό έχει σχέση και με το γεγονός ότι έχει την Προεδρία αυτή τη στιγμή, αλλά συναντήθηκα και με γεωργούς και επιχειρηματίες ε, και παραγωγούς με τον Πρωθυπουργό. Μετά επισκέφθηκα τη Γερμανία και Υπήρξαν και πολλές ε, διμερείς συναντήσεις με την Επιτροπή Γεωργίας, ε, πήγα και στο Bundestag, αντίστοιχη επίσκεψη έκανα και στην Αυστρία. Ε, στην Αυστρία υπήρχε η γεωργική έκθεση, επισκέφτηκα επίσης και μία εκμετάλλευση στην οποία γίνεται βιολογική καλλιέργεια. Είχα συναντήσεις με γεωργούς, προσώπους οργανώσεων παραγωγών και αυτές ε, οι συναντήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και χάρη σε αυτό έχω και μία ευρύτερη εικόνα του τι συμβαίνει στη Γεωργία. Και είχα και κάποιες συναντήσεις και στην Πολωνία, στη χώρα μου. Οι Γεωργοί υποστηρίζουν ε, την πράσινη συμφωνία, το Green Deal. Ε, βλέπουν ότι υπάρχει κάποιο όφελος, αντιλαμβάνονται ότι η γεωργία πρέπει να γίνει και πιο φιλική προς το περιβάλλον, γνωρίζουν ότι πρέπει να αναβαθμίσουν ε, την παραγωγή τους και να κάνουν και την παραγωγή τους πιο βιώσιμη. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Ε, ωστόσο υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, υπάρχουν ε, νέες απαιτήσει οι οποίες δεν υποστηρίζονται και από αντίστοιχη χρηματοδότηση. Υπάρχει λοιπόν το όλο θέμα της χρηματοδότησης και του προϋπολογισμού της κοινή γεωργικής πολιτικής και όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν. Η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι ο προϋπολογισμός ο οποίος έχει προβλεφθεί το 2018 είναι η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καθήκον μου είναι να υπερασπιστώ την πρόταση του προϋπολογισμού από το 2018 και είχα δηλώσει δημοσίως ότι θα υπερασπιστώ τη διατήρηση αυτού του προπολογισμού. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις για περικοπές και για μείωση του προπολογισμού, αλλά εγώ ε, θα ήθελα να παραμείνει ο προϋπολογισμός αυτός. Επίσης θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να προλάβουμε και κάποιες ε, προτάσεις ε, για αύξηση. Ε, θέλουμε να ενισχύσουμε και να ενδυναμώσουμε τον προπολογισμό και βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίω, οι Υπουργοί Γεωργία δεν είναι οι μόνοι που ενδιαφέρονται και λαμβάνουν αποφάσει. Ε, βλέπω όμω ότι υπάρχει μια κάποια προθυμία. Ε, φαίνεται να είναι έτοιμοι κάποιοι και ο κόσμο θέλει να ενισχύσει κάπω τον προπολογισμό. Ε, είναι θετικό λοιπόν αυτό το μήνυμα. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση τη Γαλλία, Γερμανία και τη Ισπανία των αρμοδίων υπουργών και οι υπουργοί αναφέρονται στην ενίσχυση του προπολογισμού τη ΚΑΠ και φυσικά αυτό είναι θετικό μήνυμα. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι στην επόμενη συνάντησή μας θα μπορέσω να σας πω ίσως κάποια περισσότερα πράγματα, διότι αυτή τη στιγμή είμαι στο στάδιο της ανάλυσης ε, και αξιολόγησης, κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο ιδίω ε, όταν θα συζητήσουμε τον αντίκτυπο του Green Deal και τι αντίκτυπο είχε στην ΚΑΠ. Ακόμα λοιπόν είμαστε στη διαδικασία της ανάλυσης και ε, βεβαίως γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο πέρασε και σχετικό ψήφισμα στο οποίο έκανε έκκληση ε, για τον ίδιο λόγο και επίσης ζητήσατε να γίνει και αξιολόγηση της συμφωνίας με στόχο φυσικά να δούμε και τη γεωργία. Και αυτό κάνει αυτή τη στιγμή η Επιτροπή και θα παρουσιάσουμε την άποψή μας στην επόμενη συνάντησή μας. Υπάρχει, όπως σας είπα, λοιπόν, το θέμα του προπολογισμού. Και αν ε, θεμέλιο της περαιτέρω συζήτηση για τον προπολογισμό είναι το Green Deal και ε, διαπιστωθεί ότι χρειαζόμαστε αύξηση του προπολογισμού για να εφαρμοστεί, τότε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και μια πολιτική συμφωνία. Ε, έτσι αξιολογώ εγώ την κατάσταση. Ε, πρέπει επίσης να δούμε και το δεύτερο πυλώνα, τα οικολογικά σχέδια, τα eco schemes και το πρώτο πυλώνα και τι χρηματοδότηση χρειάζεται εκεί και νομίζω ότι αν υπάρξει κατάλληλη συνεννόηση θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία είχαμε συζητήσει και στην ακρόασή μου. Ε, συζητήθηκαν τα οίκο schemes, υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένε προσδοκίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε να υποβάλει ένα κατάλογο και τα κράτη-μέλη να ε, επιλέγουν τα οίκο που προτιμούν. Πρέπει να σας πω ότι εμείς καταρτίζουμε τώρα ε, τον προϋπολογισμό, το εξετάζουμε και αν υπάρχει κάποια πρωτοβουλία από πλευρά σας, τότε ε, θα πρέπει να συζητηθεί γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν έχει κάποια πρωτοβουλία, αλλά αν υπάρχει αντίστοιχη πρωτοβουλία από πλευρά σα, θα μπορέσουμε ίσω να έχουμε ε, ένα σχέδιο καταλόγου για να καταλήξουμε σε συμβιβασμό, αν υπάρχει πολιτική διάθεση βεβαίω να αλλάξουν τα προγράμματα αυτά. Για την ε, βιολογική γεωργία. Είμαστε στη διαδικασία προετοιμασίας του σχεδίου δράσης. Οριστικοποιείται το σχέδιο κειμένου για την ανάπτυξη βιολογικών εκμεταλλεύσεων Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Είναι πολύ διαφοροποιημένο το επίπεδο εξέλιξης αυτής της μορφής γεωργίας και το συζήτησα το θέμα και όταν ήμουν στην Αυστρία. Και συζητήθηκε το εξής. Κάποιες εκμεταλλεύσεις μπορεί να χάσουν ε, τη σφραγίδα της βιολογικής εκμετάλλευσης διότι ε, δεν μπορούν να επιτύχουν το επίπεδο των προσδοκιών. Ε, είναι θέμα κτηνοτροφίας, πρόσβαση σε βοσκοτόπους, ε, που βρίσκονται σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν, για παράδειγμα, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες ε, δεν είναι ενιαίες, είναι διάσπαρτες και δεν υπάρχει δυνατότητα τα ζώα να έχουν πρόσβαση σε βιολογικούς βοσκοτόπους. Επισκέφτηκα μια τέτοια εκμετάλλευση Υπάρχουν κάποια ε, πρότυπα τα οποία τηρούνται, για παράδειγμα είναι ελευθέρας βοσκής, ε, τα ζώα, αλλά υπάρχει ένα θέμα ε, που αφορά την πρόσβαση σε βοσκοτόπους και αυτό φυσικά μπορεί να αποτελήσει και τραγωδία για περίπου 2.000 εκμεταλλεύσεις που μπορεί να χάσουν τη σφραγίδα της βιολογικής καλλιέργειας και κτηνοτροφίας παρά το γεγονός ότι ασχολούνται με τέτοιες ε, Μορφέ καλλιέργεια εδώ και χρόνια. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση ώστε να υπάρχει και μια πιο δίκαιη ε, συμφωνία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και ότι οι περιπτώσεις αυτές ε, είναι ιδιαίτερες. Συζητήθηκε επίσης και το θέμα της συγκέντρωσης ε, της γης και νομίζω ότι υπήρχε και ένα σχετικό ψήφισμα. Η κυρία Μίλλερ ήταν ε, αρμόδια, αν δεν κάνω λάθος, ε, τη συγκέντρωση της των γεωργικών γεών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα. εμείς δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τα θέματα ιδιοκτησία και κατοχής των γεωργικών γεών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά Γίνεται αυτή τη στιγμή μια αναθεώρηση διαφόρων κανονισμών που ισχύουν στα κράτη-μέλη, κανονισμοί οι οποίοι προστατεύουν ε, τις ΓΕΕΣ ε, από τη συγκέντρωση ε, γεωργικών γεών, υπάρχουν κάποιες καλές πρακτικές, ε, υπάρχει νομοθεσία στα κράτη-μέλη, θα πρέπει να τα εξετάσουμε όλα αυτά και πράγματι πρέπει να αναλάβουμε δράση, διότι το 3% των ιδιοκτικών είναι κάτοχοι του 50% της γεωργικής γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά αυτό δεν είναι προς όφελος κανενός. Υπάρχει ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα, το οποίο θα αποτελεί και μία από τις προτεραιότητές μου. Το συζητώ με την Επίτροπο Φερέιρα, η οποία είναι αρμόδια με θέματα ε, περιφερειακής πολιτικής. Θα θέλαμε η αγροτική πολιτική να αποτελέσει ένα από τα πολλά εργαλεία για την ανάπτυξη των περιοχών της Υπέθρου. Υπάρχει πολιτική συνοχής, και όπως ε, διαπιστώνουμε η πολιτική συνοχής δεν ε, συνεισφέρει και πάρα πολύ στην ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου. Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν σε περιοχές της υπαίθρου και δεν είναι γεωργοί και αυτό είναι φυσικά απόλυτα φυσιολογικό. Θεωρούμε λοιπόν ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει επίσης να συμβάλλει και στην ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου πρέπει να υπάρχει συνέργεια μεταξύ των δύο πολιτικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτή η ιδέα είναι αρκετά δημοφιλής. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρξουν αυτές οι συνέργειες και θα πρέπει να υποστηρίξουμε καταλήλως και τις περιοχές της υπαίθρου χρησιμοποιώντας τα ταμεία συνοχής. Αυτό Αυτά είναι λοιπόν τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία μας απασχολούν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας για συζήτηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επίτροπε για αυτή την εισαγωγή και ε, είδα ότι δεν διαβάζετε μόνο το έγγραφο που σας έχουν προετοιμάσει, αλλά μας αναφέρατε και τις εμπειρίες σας ε, τις πρώτες εβδομάδες, το χάρη δύο καλλιέργειες στην Αυστρία, εκεί δηλαδή όπου υπάρχει πρόβλημα, όπου ε, ορισμένες εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα και πρέπει κάπως να αντιμετωπιστούν. Ο κύριος Ντόρφμαν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, καταρχήν που ήρθατε και καλή σας μέρα. Ε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για το γεγονός ότι επισημάνατε ποιοι είναι οι στόχοι μας κατά τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πράγματι πρέπει να σκεφτούμε ε, ποιος πρέπει να είναι ο στόχος αυτής της πολιτικής. Και μερικές φορές έχω την εντύπωση ε, μετά τα 10 χρόνια η αποκομμένες ε, άμεσες ενισχύσεις. Αυτό θα σημαίνει ανακατανομή των κονδυλίων ε, που σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορεί να παίρνουν όλοι οι κονδύλια, γιατί σε μια πολιτική πρέπει κανείς να σκέπτεται τι ακριβώς επιθυμεί να προωθήσει και να φέρεται ορισμένα θέματα. Παραδείγματο χάνει το ερώτημα, θέλουμε να ενισχύσουμε οικογενειακέ εκμεταλλεύσεις ε, αυτού που πραγματικά καλλιεργούν τη γη. Και επισημάνατε ότι, και έχετε δίκιο, ότι η αρμοδιότητα για την ε, θέσπιση διατάξεων ε, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά μπορώ επίσης να σε εγγυηθώ ότι αν τελικά ε, δεν χρηματοδοτήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις, τότε απλά δεν θα υπάρχουν. Άρα δηλαδή, σε τελική ανάλυση, η γεωργική πολιτική είναι εκείνη που προκάλεσε τα προβλήματα και που οδήγησε στο να υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα. Οφείλουμε λοιπόν να προωθήσουμε περισσότερο στο επίκεντρο των ενδιαφέροντός μας, τους νέους ανθρώπους, τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και να προάγουμε τη γεωργία και την υπεθρό. Νομίζω αυτό λιγάκι το ξεχάσαμε, ότι η γεωργία Ήπεθρος χρειάζεται επιχειρήσεις, χρειάζεται γεωργούς, άρα δηλαδή η γεωργική ζωή πρέπει να είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας και με μέσα της πολιτικής συνοχής. Αναφέρατε σημαντικά θέματα, την πράσινη συμφωνία. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως γεωργοί, να μην είμαστε απλά θεατές ε, και εδώ στο Κοινοβούλιο και νομίζω και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχω λιγάκι την εντύπωση ότι άλλοι ε, θέλουν θέλουν να αναλάβουν αρμοδιότητες ε, και να μην αφήσουν τους γεωργούς να συναποφασίζουν. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, όσον αφορά στη στρατηγική που θα ακολουθηθεί. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο, είναι και θέμα της γεωργίας. Και αν δεν συμπεριλάβουμε και τους γεωργούς στην Πράσινη Συμφωνία, αυτή δεν θα επιτύχει. Γι' αυτό κάνω έκκληση σε εσά ε, να εκπροσωπήσετε πραγματικά τα συμφέροντα των γεωργών. Ο κύριος Παύλο Ντικάστρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας καλωσορίζουμε κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε επίσης για την παρέμβασή σας, η οποία παρέμβασή σας ε, κατ' ουσίαν ε, αναφέρεται και σε αυτά που είχαμε ήδη πει, είχατε ήδη πει στην ακρόαση στο Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό το Eco Scheme, αυτό το πολύ σημαντικό στόχο της κοινή γεωργικής πολιτικής, αυτό δηλαδή που είναι οι μεγάλες περιβαλλοντικές ε, προκλήσεις που καλύτερα να αντιμετωπίσει και αυτή η Επιτροπή με, με την Πράσινη Συμφωνία. Είναι φιλόδοξα μέτρα, τα οποία όμω πρέπει να την χάνουν διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η διαχείριση να μην είναι μόνο θέμα κρατών μελών. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι που και εσεί επιβεβαιώσατε αυτή την προσέγγιση. Όπω είπε όμω και συνάδελφο κύριος Ντόρφμαν, είναι σημαντικό τη στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο να τη συνδέσουμε με τη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική. Δεν πρέπει να ε, λέμε δίθεν στου γεωργού ότι ε, θα υπάρξουν περισσότερε δεσμεύσει ε, με την κοινή πολιτική, με τη στρατηγική ε, από το χωράφι στο πιάτο και αυτά να τα λέμε ότι θα τα κάνουμε, αλλά κατ' ουσίαν κόβουμε κονδύλια από τον ένα τομέα για να τα περάσουμε στον άλλο. Ε, μην ξεχνάμε, οι Γεωργοί είναι πραγματικά οι πρωταγωνιστές. Και αυτό που είπατε κι εσείς, ότι μια πολιτική των κινήτρων, αυτό πρέπει να υπάρχει, όχι πολιτική τιμωρία. Εμείς θέλουμε να ε, κινητροδοτήσουμε, να πούμε στους Γεωργούς να κάνουν περισσότερα, να τους δώσουμε ευκαιρίες, όχι να επιβάλλουμε τιμωρίες. Κύριε Επίτροπε, ε, αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. βεβαίω και δεν είναι εύκολο, γιατί και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε δυσκολίες. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα έχετε αντίστοιχε δυσκολίες ε, στο σώμα των Επιτρόπων. Αλλά κύριε Επίτροπε, αν έχουμε μια κοινή στρατηγική, νομίζω ότι θα πετύχουμε το στόχο μας. Καλή δουλειά σας εύχομαι συνάδελφος Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας στην Πράσινη Εβδομάδα και για αυτά τα λόγια στα γερμανικά που είπατε κατά την εισαγωγή σας. Η ατμόσφαιρα που ήταν ε, κατά τη διάρκεια της Πράσινη Εβδομάδα στους Γεωργού ήταν πάρα πολύ Ποτέ δεν ήταν έτσι. Οι Γεωργοί ε, φοβούνται ότι ε, θα αναγκαστούν να υπαχθούν στη γερμανική νομοθεσία και αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή χάνουμε τους νέους γεωργούς, δεν θέλουν αυτοί να συνεχίσουν τις εκμεταλλεύσεις. Εγώ έχω πάρα πολλά ερωτήματα για το τι ακριβώς ε, μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, μέχρι ποιου βαθμού μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η κοινή πολιτική μπορεί να αντιταχθεί σε αυτή την πράσινη συμφωνία που είναι καλή, όλοι οι γεωργοί γνωρίζουν ότι πρέπει να προστατεύουμε καλύτερα το περιβάλλον και θα χαρούμε όταν θα εκταμιευθούν τα κονδύλια, αλλά εξακολουθούμε να ανησυχούμε ότι παρόλα αυτά οι γεωργοί δεν θα πάρουν τα κονδύλια και απλά θα αναγκαστούν να κατακλειστούν με χιλιάδες διατάξεις. Μιλήσατε κύριε Επίτροπε για αξιολόγηση των επιπτώσεων εκτίμηση αντικτύπου. Αν γίνει αυτό από πλευρά επιτρική Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σα παρακαλώ να τα συνεπολογίσετε όλα, όπως τη διαγραφή τη προστασία των φυτών, μείωση των λοιπασμάτων, ε, προποθέσει για την ευημερία των ζώων. Αυτά όλα είναι δαπάνε που σε τελική ανάλυση επιβαρύνουν το γεωργό και αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε εκτίμηση αντικτύπου όμως ε, ξεχνάμε το επιπλέον κόστος που επιβαρύνει τη γεωργία, αυτό δεν είναι σωστό. <clears throat> Το τρίτο που θέλω να πω αφορά στα βιολογικά προγράμματα. Γνωρίζετε ότι εμείς στη Γερμανία αυτή τη στιγμή ε, υπάρχουν περιορισμοί για το βιολογικό γάλα. Το βιολογικό γάλα δεν μπορεί να πουληθεί πια στην αγορά σε υψηλότερη τιμή και ε, εάν θέλουμε λοιπόν να περάσουμε όλα τα προϊόντα στις βιολογικές καλλιέργειες, ε, για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε και τα απαραίτητα κονδύλια. Κύριε Πίτροπε, ευχαριστούμε που ήρθατε. Από την προηγούμενη εβδομάδα ξέρω ότι έχουμε και ένα κοινό όραμα όσον αφορά στις βιολογικές καλλιέργειες. Παρόλα αυτά, όσον αφορά το θέμα της επικείμενης γεωργικής μεταρρύθμισης, έχει αναφερθεί επανειλημμένα Τώρα διαπραγματευόμαστε αυτά που είπε ο προκάτοχός σας. Μέχρι το τέλος του έτους θα προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά. Ε, παράλληλα έρχεται και η Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο και σκέφτομαι πώς θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Ακούμε ότι οι τριμερείς διάλογοι θα τα λύσουν όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή να πούμε ότι αυτά θα επιβαρύνουν τους γεωργούς ε, και αυτά πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στη νέα κοινή γεωργική πολιτική. Παρακαλώ λοιπόν η Κομισιόν να επιταχύνει λιγάκι. Ε, με εκπλήσει το ότι αυτή η πολιτική χωράφη στο πιάτο έχει μεταφερθεί για τον Μάιο ε, και εκπλήσαμε που δεν θα τα κάνετε εσείς όλα αυτά, αλλά ε, κάποιος άλλος επίτροπος. Εγώ θα το έβρισκα καλύτερα αυτά να παραμείνουν σε δική σας αρμοδιότητα. Μιλήσατε για βιολογικές καλλιέργειες. Ε, πράγματι έχουμε δυσκολίες. Ευχαριστούμε που ασχοληθήκατε με την Αυστρία, αλλά ε, μην ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη θέλαμε τον κανονισμό για τις βιολογικές ε, καλλιέργειες. Αυτά όλα πρέπει να εφαρμοστούν ε, σωστά για τους γεωργούς, να μην δημιουργούν ε, νέα εμπόδια. Η κυρία Μίλλορ είπε ότι χρειαζόμαστε στρατηγική για να πληρω... πουλάμε καλύτερα τα προϊόντα, τα βιολογικά στην αγορά. Όχι μόνο εκτάσεις, αλλά και καλύτερες αγορές. Γι' αυτό λοιπόν έχω να αποθέσει τις ελπίδες μου σε εσά στο να έχουμε στόχους να ενισχύσουμε αυτά τα θέματα. Κάπου διαφωνώ με τον κύριο Ντόρφμαν Ξέρετε, ε, τον στόχο της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής κάπου τον έχουμε χάσει. Γιατί δίνουμε πάρα πολλά κονδύλια, αλλά τα τελευταία 26 χρόνια χάσαμε τους μισούς γεωργούς. Κάτι πάει καλά στο σύστημα. Πρέπει λοιπόν να ε, επιβραβεύουμε τους γεωργούς και όχι να παίρνουμε την έκταση ως κριτήριο και να κατανείμουμε τα κονδύλια με βάση αυτό το κριτήριο. Υπάρχουν και άλλα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφος και κύριε Τάβιντ. Zemědělci jsou stále popisováni jako největší eh, škůdci přírody. Eh, je pravda, že lidé... Η πράσινη συμφωνία παρουσιάστηκε και η, η γεωργία συχνά παρουσιάζεται ως εχθρός της φύσης. Πού λοιπόν θεωρείτε ότι θα προκύψουν ενδεχομένω τριβέ. Πού θεωρείτε ότι θα προκύψουν ενδεχομένω τριβέ λοιπόν. και δυσκολευόμαστε να φανταστούμε τρακτέρια παράδειγμα τα οποία κινούνται με την ενέργεια μπαταρία. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν γενικοί στόχοι επί των οποίων όλοι συμφωνούμε. Θέλουμε να αντικαταστήσουμε για παράδειγμα ε, τα ρηκτά καύσιμα. Με τι όμω θα τα αντικαταστήσουμε. Οι βιολογικέ καλλιέργειε είναι ιδιαίτερω ε, κοστοφόρε και οι γεωργοί χρειάζονται περαιτέρω πόρους. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι ολοένα και συρρυκνώνει το πληθυσμό των ε, γεωργών. Ένα άλλο θέμα, οι εισαγωγέ από τρίτες χώρες. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι και εκεί θα γίνονται σεβαστά τα πρότυπα τα οποία επιβάλλουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Κούτσμικ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος της ομάδας των Συντερικών και μεταρρυθμιστών για το γεγονό ότι ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας και κατά τη διάρκεια της ακρόασής σας θυμάμαι ότι σχολιάσατε ότι σκοπεύετε να συνεργαστείτε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η επίσκεψή σας το επιβεβαιώνει αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω δύο ζητήματα. Το ένα εξ αυτών το αναφέρετε και εσείς εισαγωγικά. Το σχέδιο προϋπολογισμού. Και το δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 2027 έχει υποβληθεί, υποβλήθηκε τον Μάιο του 2018 από τον προηγούμενο Επίτροπο. Δεν έγινε τότε συζήτηση καμία προφανώς και κανείς δεν είχε ακούσει άλλωστε τότε την Πράσινη Συμφωνία, το Green Deal. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, η καινούργια Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε αυτό το νέο Πράσινο Σύμφωνο, την Πράσινη Συμφωνία. Και να πούμε ότι αυτό το κομμάτι που αφορά την ΚΑΠ δεν ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι Γεωργοί. Υπάρχουν λοιπόν τριβές και εντάσεις στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ε, έγιναν ε, στις δυτικοευρωπαϊκές ε, χώρες, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, βγήκαν στους δρόμους, ξεχύθηκαν οι Γεωργοί. Πιστεύετε λοιπόν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το σχέδιο προϋπολογισμού δεν συνάδει, δεν ε, είναι αντίστοιχο των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι γεωργοί. Αυτό ήταν το πρώτο λοιπόν θέμα. Κατά δεύτερο, είπατε ότι επισκεφτήκατε την Αυστρία και μικρές ε, φάρμες, μικρά αγροκτήματα, οικολογικά και βιολογικά. Στην ακρόασή σας είχατε δηλώσει ότι θα είναι η προτεραιότητά σας ότι θα κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να υποστηρίξετε τη βιολογική γεωργία. Ξέρουμε όλοι ότι στο δεύτερο πυλώνα υπάρχουν πολλοί περιορισμοί. Περιορισμοί που εμποδίζουν τα μικρά αγροκτήματα από το να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Προτίθεστε να τα καταργήσετε αυτά τα εμπόδια. Ο κύριο Φλέντινγκ. Πάνε Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, Επίτροπε, στην πρώτη σημαντική σας συνάντηση ε, ως Επιτροπός Γεωργίας και καλή επιτυχία σας εύχομαι στο έργο σας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η θέση σας. Αν την κάνετε καλά τη δουλειά σας, το μέλλον θα είναι καλός. Είπατε ότι θα προσπιστείτε τον προϋπολογισμό. Πείτε μας όμως, πώς. Πώς. Γιατί. Το ποσοστό του συνολικού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την Γεωργία προτείνεται να πάει από το 39,36% στο 28,5%. Συζητάμε ε, πολύ και επιμακρών πώς θα πετύχουμε την περικοπή αυτή, αλλά γιατί. 2.000% αύξηση και πλέον για τον προπολογισμό της άμυνας. Θα πολεμήσετε για να πετύχουμε μεγαλύτερη μερίδα της πίτας για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό για τη Γεωργία. Γιατί ακούσαμε τον ε, Ιρλανδό Πρωθυπουργό χθε βγήκε και δήλωσε ότι θα κοιτάξτε τι θα γίνει με τον εθνικό προπολογισμό. Αυτό σημαίνει για μένα ότι πολλοί έχουν ήδη καταλήξει την προσπάθεια να αντιτηρήσουν τον προπολογισμό στα ίδια επίπεδα. Θα προασπιστείτε λοιπόν, θα υπερασπιστείτε το ποσοστό το οποίο αναλογεί στην γεωργία. Για το πώ ε, δαπανούμε λοιπόν τα χρήματα αυτά. Η Μερκοσούρ, για παράδειγμα, 100 εκατομμύρια ε, έλαβε η Ιρλανδία το καλοκαίρι, 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 50% από την ε, Ιρλανδία, το ποσοστό χρηματοδότηση ε, για να μειώσει την παραγωγή της. Και παράλληλα εισάγουμε βόλιο κρέα από το Μερκοσούρ. Πώς θα σβήσουμε αυτές τις πυρκαγιέ που μόνοι μας έχουμε ανάψει. Σε ό,τι αφορά τι εγγυημένε πληρωμέ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει το Μάιο. Δικό μα είναι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Γιατί να μπορούν να αρνηθούν τα κράτη-μέλη τέτοιε πληρωμέ που βασίζονται σε κοινωνικό δίκαιο. Υποστηρίζω λοιπόν την ιδέα προάσπιση τη βιοπικιλότητα, αλλά θα πρέπει να το πληρώσουμε όλα αυτά. Θα επιμείνετε όλα αυτά να χρηματοδοτηθούν. Και τέλο, για τι καταναμημένε πληρωμέ. Είχαμε πει 100% η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 60% είπαμε μετά. Ε, θα πολεμήσετε όμως για 100% πληρωμές επανακατανομής. Και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και έτσι ολοκληρώσαμε το γύρο των ε, συντονιστών. Τώρα, να ακούσουμε τις πρώτες απαντήσεις του Επιτρόπου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους Ευχαριστώ και όλους τους συντονιστές. Ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Και αναφερθήκατε και σε πολλά θέματα τα οποία με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Αναφερθήκατε σε θέματα προπολογισμού, αλλά επίσης ε, αναφερθήκατε και στην οτροπία της ΚΑΠ και έχει δίκιο ο κύριος Ντόρφμαν. δεν έχουμε σαφή εικόνα της κοινή γεωργικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές οι οποίες ε, ε οδηγούν σε αύξηση των εκμεταλλεύσεών μας. Υπάρχουν ε, ε μικρές εκμεταλλεύσεις που, που εξαφανίζονται γιατί δεν είναι σε θέση να γίνουν ανταγωνιστικές. Και τώρα έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση και να αναστρέψουμε αυτές τις διαδικασίες. Πρέπει λοιπόν να την εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και να χρησιμοποιήσουμε τον Green Deal για να δώσουμε ένα τέλος σε αυτές τις αρνητικές ε, διαδικασίες. Για να μπορέσουμε όμως να τη χρησιμοποιήσουμε τη συμφωνία θα πρέπει να έχουμε και αντίστοιχη χρηματοδότηση. Χρειάζονται χρήματα. Δεν είναι δυνατόν η γεωργία μας να αναπτυχθεί ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν μειώσεις στον πρώτο πυλώνα και στο δεύτερο πυλώνα ταυτόχρονα. Η Ευρωπαϊκή Γεωργία δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση. Επίσης, ε, λιγότερες ουσίες προστασίας θα οδηγήσουν σε απώλεια εισοδήματος για τους γεωργούς. Υψηλότερα πρότυπα ευημερίας των ζώων σημαίνει και επιπλέον κόστος. Τα καλύτερα εργαλεία για όλα αυτά βρίσκονται στο δεύτερο πυλώνα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη, αλλά έτυχε να βρεθώ στην Αυστρία και διαπίστωσα ότι ο, ο δεύτερος πυλώνας λειτουργεί πολύ καλά και ε, δαπανώνται ε, τα περισσότερα κονδύλια για να υποστηρίζονται τα προγράμματα περιβαλλοντικής ε, ε, υγείας. Υποστηρίζουμε λοιπόν έναν ισχυρό δεύτερο πυλώνα και αν μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και όλες τις βιολογικές εκμεταλλεύσεις θα μπορέσουμε να επιτύχουμε καλούς στόχους και να έχουμε και σωστά αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία γιατί το Green Deal αποτελεί πολύ καλό πρόσχημα ώστε η στήριξη να πάει σε μικρότερες, πιο αδύναμες εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μέχρι τώρα εξαφανίζονταν γιατί δεν ήταν σε θέση να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες. Θα μπορέσουν λοιπόν με αυτή την υποστήριξη να επιβιώσουν. Κύριε Ντεκάστρο, αναφερθήκατε στα 20 games και όπως σας είπα και εγώ, είμαι καθόλου διατεθειμένος να κάτσω γύρω από ένα τραπέζι και να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και να δούμε συγκεκριμένα θέματα, συγκεκριμένες λύσεις. Ε, καταρχήν συμφωνώ και το συζητούν και οι ίδιοι οι Γεωργοί. Δεν είναι απλώς ένα πολιτικό αίτημα. Οι Γεωργοί θέλουν να γνωρίζουν λίγο καλύτερα τι πρέπει να κάνουν προκειμένου να μπορέσει να θεωρηθεί ότι τηρούν τους κανόνες. Θέλουν να γνωρίζουν πώς έχει η κατάσταση, χρειάζονται σαφείς κανόνες και επομένως είμαι ε, έτοιμος για συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε αυτό το θέμα. Η κυρία Μίλλερ αναφέρθηκε και αυτή στα EcoSchemes, ε, στα οικολογικά αυτά προγράμματα και όπως ε, είπα, αυτό το μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη βιολογική γεωργία είναι στα σκαριά αυτή τη στιγμή. Ε, και το είπε και ο κύριος ε, Χόλμερ. Δεν είναι μόνο θέμα της αύξησης της επιφάνειας αυτών των βιολογικών εκμεταλλεύσεων. Θέλουμε να αυξήσουμε τη βιολογική παραγωγή και τη βιολογική κατανάλωση. Είναι πολύ διαφοροποιημένη η κατανάλωση στα κράτη-μέλη και αν χρησιμοποιήσω και πάλι το παράδειγμα της Αυστρίας, το κάνω γιατί πήγα πρόσφατα, ε, σχεδόν το 25% της γης είναι ε, βιολογικές εκμεταλλεύσεις όπου γίνεται βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και η κατανάλωση είναι περίπου 200 ευρώ κατά κεφαλήν στην Αυστρία. Και πρέπει να πω ότι στην Πολωνία, για να κάνω σύγκριση εδώ με την Αυστρία, έχουμε μόνο 4 ευρώ κατά κεφαλήν κατανάλωση βιολογικών προϊόντων. Οι διαφορές αυτές λοιπόν είναι τεράστιες. Πρέπει να αναπτύξουμε τη βιολογική γεωργία, αλλά δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο ε, μεγαλύτερη επιφάνεια καλλιέργειας εκτινοτροφίας. Θα πρέπει αυτό ε, να γίνεται και με αναλογικό τρόπο. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλο ζευγάρι, να προωθήσουμε ε, και τα βιολογικά προϊόντα και αυτό είναι τμήμα του σχεδίου δράσης που θα σας υποβάλουμε σύντομα. Υπήρξαν και κάποιες ερωτήσεις για τη στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο. πολλά γεωργικά ζητήματα είναι αρμοδιότητα άλλων γενικών διευθύνσεων. Για παράδειγμα, ε, το κατά πόσο θα επιτρέπονται ε, φυτοφάρμακα και ζυσανοκτών. Αυτά είναι αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΤΕ. Σας διαβεβαιώ όμως ότι εγώ συμμετέχω ενεργά σε όλες τις εσωτερικές εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όποια απόφαση ληφθεί επί του θέματος θα πρέπει ε, να βασίζεται και σε αξιολόγηση επιπτώσεων. Και εγώ θα φροντίσω ε, το θέμα αυτό και επίσης θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αν υπάρχει οποιαδήποτε νέα πρόταση για υψηλότερα πρότυπα, υψηλότερες απαιτήσεις, ε, υψηλότερες πιέσεις ε, προς τους γεωργούς, θα πρέπει να τους φροντίσουμε κιόλα. Θα πρέπει να φροντίζουμε τους γεωργούς μας, επομένως εγώ θα ασχοληθώ ιδιαίτερα ενεργά με το θέμα αυτό και δεν θα αλλάξω και στάση. Ο κύριος Ντάβιτ είπε ότι ναι, όντως υπάρχει το πρόβλημα ότι ορισμένες φορές ε, παρουσιάζει κανείς τον Γεωργό ως τον ένοχο. Αυτό ο οποίος ε, είναι υπεύθυνος ε, για τα κλιματικά προβλήματα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Είναι τα πρώτα θύματα. Η ξηρασία και οι φυσικές καταστροφές ε, πλήττουν τους γεωργούς όλο ένα και περισσότερο. Επομένως, οι γεωργοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όλης αυτής της μάχης ε, για το κλίμα. Φυσικά και υπάρχουν και σκέες γεωργικές πρακτικές τις οποίες θα πρέπει να περιορίσουμε ή και να πατάξουμε εάν είναι επιζήμιες για το περιβάλλον. Για παράδειγμα, μου έρχεται τώρα στο νου η γεωργία που είναι τόσο εντατική που είναι πλέον βιομηχανία. Και φυσικά αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Ε, οι, οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις, οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι υπεύθυνοι για αυτή την καταστροφή και μπορεί να υπάρξει και θετικός αντίκτυπος ε, χάρη στη συμβολή τους. Ρωτήσατε και για τις ε, διαδηλώσεις των γεωργών στην Ευρώπη. Ναι, φυσικά και το γνωρίζω. Υπάρχουν ε, γεωργοί οι οποίοι διαμαρτύρονται. Εγώ μίλησα και στους διοργανωτές ε, του κινήματος και φυσικά ο κόσμος ανησυχεί. Ο βασικός φόβος απορρέει από αυτές τις νέες υποχρεώσεις, τις νέες απαιτήσει. και δεν υπάρχουν επαρκή κονδύλια, γι' αυτό και ε, θα πρέπει να προσέξουμε γιατί μπορεί αυτό να είναι εις βάρος και όλου του Green Deal. Πρέπει να επαγρυπνούμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου το Green Deal να είναι επιτυχές. Το Green Deal δεν θα πρέπει να συνοδεύεται από διαδηλώσεις, συγκρούσεις και εντάσεις. Ε, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να το αποφύγουμε οι γεωργοί έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν, ε, υπάρχουν ε, και αιτήματα ε, και τα απίφθηναν και προς τις εθνικές κυβερνήσεις και οι γεωργοί ανησυχούν. Όσον αφορά τις μικρές εκμεταλλεύσεις που ανέφερε ο κύριος Κούσνικ, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Εγώ αναλύω τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ρήτρε που ε, ε, αποκλείουν τελικά τους ε, μικρούς ε, γεωργούς. Υπάρχει ένα ανώτατο όριο, ένα κατόφλι αποκοπής και τελικά αυτοί αποκλείονται από τη χρηματοδότηση και τα κονδύλια πηγαίνουν στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις και οι μικροί γεωργοί αποκλείονται. Εξαρτάται βέβαια από το πρόγραμμα, δεν είναι συνολικός αυτός ο κανόνας, αλλά τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ, τα οποία και είναι η αρμοδιότητά μου και θα τα υποπτεύω, είναι κάτι επί το οποίο θα ήθελα να επικεντρωθώ θα πρέπει άλλωστε να θυμόμαστε και τους μικρούς γεωργούς. Πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και αυτοί στη χρηματοδότηση του δεύτερου πυλώνα. Αυτή θα είναι μία από τις προτεραιότητές μου. Πρέπει ο δεύτερος πυλώνας να γίνει πιο δημοκρατικός, διότι σε κάποια προγράμματα υπήρξε μια στενή ομάδα δικαιούχων και θα πρέπει να φροντίσουμε να διευρύνουμε αυτή την ομάδα και κάθε γεωργός ο οποίος είναι πρόθυμος και θέλει να συμμετέχει σε αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να έχει και τη δυνατότητα να συμμετέχει. Κύριε Φλάναγκαν, οι ερωτήσεις σας αναφέρονται στον προϋπολογισμό, ε, πώς ε, θα υπερασπιστώ τον προϋπολογισμό. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό θα γίνει βάσει και της εντολής που μου έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, μετέχω σε πολιτικές συζητήσεις και προσπαθώ να πείσω τα κράτη-μέλη, γιατί αυτό είναι στα χέρια τους. Προσπαθώ λοιπόν να πείσω τα κράτη-μέλη να είναι πιο τολμηρά ε, για τον προϋπολογισμό. Έκανα πολλές συναντήσεις, πολλές συζητήσεις ε, με κράτη-μέλη και ελπίζω ότι θα υπάρξει μια θετική αλλαγή και θα αλλάξει στάση των κρατών μελών και θα υπάρξουν αυξήσεις. Είναι τεράστιες οι προκλήσεις και για να αντιμετωπίσουμε αυτές τι προκλήσεις πρέπει να έχουμε κατάλληλα μέσα και κονδύλια. Ιδάλω, η ωραία ιδέα του Green Deal δεν θα υλοποιηθεί. Ιδιαίτερα στη Γεωργία. Είναι λοιπόν προ το κοινό μα συμφέρον να μην επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για τον πρώτο γύρο απαντήσεων και τώρα θα λάβουν το λόγο και άλλοι συνάδελφοι. Να σας πω ότι έχουμε περίπου 30 συναδέλφους που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός ε, στην τήρηση του ενός λεπτού. Συνάδελφος Αγγιλάρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, καλώς ορίσατε. Είπατε ότι στην επίσκεψή σας στην Αυστρία είδατε την επιτυχία του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ. Ελπίζω στην επόμενη επίσκεψή σας στην Ισπανία και ελπίζω να έρθετε το συντομότερο θα μπορέσετε να διαπιστώσετε και την επιτυχία του πρώτου πυλώνα της ΚΑΠ που δημιουργεί πλούτο, ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα. Στη σημερινή σας παρέμβαση αναφερθήκατε στο Green Deal και στην ε, μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι βραχυπρόθεσμες συνέπειες της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και η νέα συμφωνία αυτή ανησυχούν τους γεωργούς. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, όπως ε, ρώτησε και κάποιος άλλος συνάδελφος, να σας ζητήσω μάλλον να είστε εσείς αυτός ο οποίος θα καθοδηγήσει αυτές τις συζητήσεις και τα όσα διακυβεύονται. Οι συνάδελφοι του περιβάλλοντος και της υγείας θέλουν να έχουν τον τελευταίο λόγο, αλλά εσείς είστε ο μόνος αρμόδιος και ο πλέον αρμόδιος να αναλάβετε τις ευθύνες για τον κτηνοτροφικό και γεωργικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους ε, δασμούς ε, των ε, Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει κατεπηγόντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει τις ε, πληγήσεις χώρες. Ευχαριστώ και επαναλαμβάνω, ελπίζω να σας δούμε πολύ σύντομα στην Ισπανία. Χαίρομαι που ήρθατε κύριε Επίτροπε. Εμένα αυτό που με σοκάρισε περισσότερο σε αυτά που είπατε ήταν το γεγονός ότι περίπου 3% όλων των ε, ιδιοκτητών ε, έχουν το σύνολο των εκτάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό μοιάζει να μην ενοχλεί κανένα. Μιλάμε όλοι για μικρούς γεωργούς, αλλά το 3% των γεωργών έχει στην ιδιοκτησία του το σύνολο των εκτάσεων. Και διερωτώ που υπάρχει κανείς ε, να στηρίζει την, τις ενισχύσεις κατέκταση στον πρώτο κανόνα. Αυτό δηλαδή σημαίνει κατ' ουσίαν στηρίζεται την τελείως λανθασμένη γεωργία. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και εγώ Παρά τις ε, κομματικές διαφορές ε, θα ήθελα να βρούμε νέες ε, καινοτόμες προσεγγίσεις για να αλλάξουμε τη γεωργία. Γιατί ξέρουμε ότι είμαστε στρεμωγμένοι στον τοίχο. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η πράσινη συμφωνία γιατί έχουμε τεράστια προβλήματα. Και ως γεωργοί δεν χρειάζεται να βρούμε ένα οχυρό για να μπούμε από πίσω και να πυροβολούμε. Είναι πολύ σημαντικό να προστατευτεί ο δεύτερος πυλώνας. Και επειδή θα υπάρξουν περικοπές Ευρωπαίες διαιρωτώ με κατά πόσο θα μπορούσαμε να υποχρώσουμε τα κράτη-μέλη να προβλέψουν ε, ελάχιστα κονδύλια, δεσμευτικά κονδύλια για τις βιοκαλλιέργειες, γιατί αλλιώς θα εξαφανιστούν τελείως οι βιοκαλλιέργειες. Ε, παρακαλώ να τηρείτε τον χρόνο αγόρευσης που προβλέπετε για κάθε έναν από εσάς. Η συνάδελφος κυρία Τόμασιτς έχει το λόγο. πολύ σύντομα, ε, κύριε Επίτροπε. Ορισμένα κρατημέλη συμπεριλαμβανομένης και της ε, Κροατίας πολύ συχνά έχουν ε, εκτάσεις που δεν καλλιεργούνται. Υπάρχουν γεωργοί που μπορεί να έχουν θαυμάσια ιδέες αλλά δεν έχουν αρκετή έκταση στη διάθεσή τους. Θέλω λοιπόν να κατανοήσω με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Τροπή θα προσπαθήσει να πείσει τα κράτη-μέλη να αναδιανύμει τις εκτάσεις, να προβεί σε ανακατανομή γης. Συνάλφος Φριτσάνοβα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, ομιλία σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει αναφερθεί. Πρόκειται για τη χρήση νέων τεχνολογιών στη Γεωργία. Αναφέρομαι στην ε, τεχνική των ε, γονιδίων ε, κατά πόσον προτίθεστε να μειώσετε τη χρήση φυτοφαρμάκων και παράλληλα όμως να μπορούν και οι γεωργοί να βιοπορίζονται. Είναι ένα αρκετά δύσκολο θέμα, γραφειοκρατικά, από γραφειοκρατική πλευρά για να εισαχθεί. Ποια είναι η δική σας άποψη από αυτού. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη εφαρμογή αυτή του θέματος. Συνάδελφος Αμάρο. Κύριε Επίτροπε, Υπάρχει το θέμα της κοινή γεωρικής πολιτικής και της πράσινης συμφωνίας. Και όλα αυτά πρέπει κάπως να συμβιώσουν και να λειτουργήσουν. Ακούσαμε διάφορες απόψεις και ε, από ό,τι καταλάβαμε, οι γεωργοί επικρίνονται επανειλημμένα, δεν υπάρχει ε, βιοπικιλότητα, αλλά ε, το θέμα, η Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει να στηρίζουμε τους γεωργούς. Κύριε Επίτροπε, αν έχουμε αρκετά κονδύλια για την κοινή γεωργική πολιτική θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, αλλιώς θα έχουμε τεράστια προβλήματα στους ε, γεωργούς της Πορτογαλίας αλλά και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να μας μιλήσετε για μικρές γεωργίες, για την ισορροπία που πρέπει να βρούμε ανάμεσα σε μεγάλες και μικρές μονάδες. Επίσης, ε, να μας πείτε πώς μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ισότητα στις πληρωμές, κυρίως στον πρώτο, αλλά και στον δεύτερο πυλώνα. Και πώς μπορούμε όλα αυτά να τα συνδέσουμε και με την πολιτική ε, συνοχή. Συνάδελφος Κρίστενσεν. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ε, χαίρομαι που είναι εδώ ο και ε, προσβλέπω σε επικοδομητική συνεργασία κατά επόμενα πέντε έτη. Έχω ένα ερώτημα. Ε, ποια είναι η στάση σας απέναντι στις νέες τεχνικές έγινε λόγος για τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Η τεχνολογία έχει πάρα πολλές δυνατότητες να δημιουργήσει νέα προϊόντα που θα είναι προσαρμοσμένα στο κλίμα. Και αυτή τη νέα τεχνολογία πρέπει να την εκμεταλλευτούμε στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Ε, θέλω να μερμηνήσετε έτσι ώστε η τεχνολογία κρίσπα να αφαιρεθεί από τον κανονισμό για τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Συνάλληφος κύριος Μπούσμαν. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που βρίσκεστε σήμερα εδώ Έχω μια ερώτηση για την προστασία των ζώων. Όταν έχουμε μεταφορές ζώων, πολύ συχνά βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, τραγικές ε, ε, μεταφορές, τραγικές καταστάσεις, κυρίως όταν τα ζώα μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μεταφέρονται με ευρωπαϊκά πρότυπα. Παραδείγματος χάνουν όταν πάνε στην Ασία, δεν υπάρχει κανένα διάλειμμα. Και όταν ε, μεταφέρει τα ζώα στη Μέση Ανατολή, παραδείγματο εκεί πεθαίνουν πάρα πολλά ζώα. Αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν υπάρχουν επαρκεί έλεγχοι. Παραβιάζονται οι κανόνε. Και εγώ ερωτώ ποια στρατηγική στηρίζετε εσεί έτσι ώστε να μην υπάρχουν τραγωδίε ε, κατά τη διάρκεια τη μεταφορά ζώων. Συνάδελφος Γιούργκελ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό και θα είμαι και σύντομος. Ε, καταρχήν, ε, θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα προς εσάς, κύριε Επίτροπε. Δεν πρέπει να κάνετε αξιολόγηση επιπτώσεων όσον αφορά στην Πράσινη Συμφωνία και καταρχήν ίσως να μας πείτε κατά πόσον οι στόχοι αυτοί ταιριάζουν με τις συμβάσεις μας ή μήπως θα πρέπει να τροποποιηθούν. Και ακόμα ένα ερώτημα. Πολλοί βουλευτές ε, έθιξαν αυτό το σημαντικό θέμα της γης, των εκτάσεων και υπάρχει μία διαδικασία που αφορά στην ε, Πολωνία και στις διατάξεις ε, για την καλλιεργήσιμη γη ε, στην Πολωνία. Ε, μήπως θα έπρεπε να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Έχει τελειώσει το λεπτό μου και εδώ σταματώ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφος Ρούσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω για τον Επίτροπο για το γεγονό ότι ήρθε εδώ σήμερα και πραγματικά ανυπομονούμε μαζί να εργαστούμε ε, μαζί αυτή την Επιτροπή. Χαιρόμαστε που υποστηρίζετε τη διατήρηση του προπολογισμού για τη Γεωργία και θα ήθελα να πω ότι ανησυχώ ιδιαίτερω σε ό,τι αφορά την Πράσινη Συμφωνία. Κυρίω επειδή θεωρώ ότι επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε πολύ υψηλέ ε, φιλοδοξίες, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς θα χρησιμοποιηθούν και ποια εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν. Αυτό χρειάζονται οι Γεωργοί. Εργαλεία ε, για τις ε, νέες ε, σοδιές, για τα νέες τρόπους, ε, προστασίας των σοδιών και το καθεξής. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο τα χρήματα. Ερωτώ λοιπόν τα εξή. Επίτροπε, πώς μπορούμε να φροντίσουμε οι εμπειρία αιώνων των γεωργών ε, στον τομέα αυτό να συμπεριληφθεί στην Πράσινη Συμφωνία. Και τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να δετεθούν τα απαραίτητα εργαλεία και η τεχνολογία που χρειάζεται για τους γεωργούς. Και αν κάποια στιγμή θέλετε να έρθετε και στην Ολλανδία, φυσικά θα σας καλοδεχτούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος η κυρία Κατάινεν. Ευχαριστώ, Επίτροπε, και χαίρομαι ιδιαίτερω που ήρθατε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι στην επιστολή αποστολή σας είπατε με σαφήνεια ότι η μελλοντική μεταρρυθμίση της ΚΑΠ θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με την πρόταση που έκανε και η προηγούμενη Επιτροπή το 2018. Ελπίζω δε ότι θα βρείτε σαφεί λύσει ε, στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περιβαλλοντική πτυχή της Νέας τη Συμφωνία και όλα αυτά θα συνδεθούν και με τα στρατηγικό σχέδιο. Προκειμένου να μην υπάρχουν επιπλέον αμα, επιπτώσεις στο εισόδημα των ε, γεωργών. Χρειάζονται πιο πολύ κίνητρο και λιγότερα αντικίνητρα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς θα εξασφαλίσετε στην Επιτροπή ότι η γεωργία και οι γεωργοί θα θεωρηθούν τμήμα της επίλυσης της ε, κλιματικής κρίσης και όχι οι αποδιοπομπέοι τράγοι. Πώς θα αποτελέσουν λύση. Η κυρία Λία Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Συνέργειες μεταξύ των διάφορων δυνατοτήτων ε, χρηματοδότησης, πώς θα εξασφαλιστούν. Ε, πράσινη συμφωνία, βιοπικιλότητα, οργανική γεωργία, βιολογική γεωργία. Ξέρουμε ότι όλα αυτά ε, έχουν διαφορετικές προθεσμίες. Είπατε ότι θα πρέπει να αλλάξει ο προπολογισμό, αλλά στο εσωτερικό της ε, ΚΑΠ προωθούνται οικονομικές αλλά και μη οικονομικές δραστηριότητες και ακριβώς ε, Γι' αυτό μιλάμε για καλύτερη ποιότητα ζωής, ε, ψηφιοποίηση, καλύτερη εφαρμογή των ε, κανόνων. Και τέλος, δεν προβλέπεται κάποια μεταβατική φάση για την μετάβαση στις ε, εθνικές επιδοτήσεις. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, κάποιες ερωτήσεις. Έρευνα το New York Times για το γεγονός ότι οι πόροι της ΚΑΠ ε, χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν λαϊκιστικά κινήματα και στην Πράσινη Συμφωνία και το θέμα της αλλαγής του κλίματος. Μας μιλήσατε ιδιαίτερως για τις Αζόρες. Ξέρουμε ότι εκεί υπήρξε μεγάλος αντίκτυπος σε ό,τι αφορά την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, αλλά και στον τομέα της γεωργίας ήταν μεγάλες οι επιπτώσεις. Έχετε κάποιες λύσεις λοιπόν να προτείνετε για να βοηθήσουμε όσους καλλιεργούν ε, φρούτα και λαχανικά στις Αζόρες γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη λειψιδρία και είναι και μεγάλη αντικτύπωση, μάλλον αντικτύπωση της αλλαγής του κλίματος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε κύριε πίτροπε. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα διότι έχουμε πολλά πράγματα στους επόμενους μήνες, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, μεταρρυθμίση της ΚΑΠ, νέο Green Deal, πρόβλημα, ε, πρόγραμμα από το χωράφι στο πιάτο ε, ποιος είναι ο ετήσιος προπολογισμός, γιατί δεν μπορούμε να αναθεωρήσουμε την ΚΑΠ χωρίς να γνωρίζουμε τι θα γίνεται με τον προπολογισμό. Το να ζητάμε περισσότερα πράγματα από τους γεωργούς με μικρότερους πόρους θεωρώ ότι δεν είναι θετικό. Και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν πολλούς τομείς οι οποίοι τιμερούνται από τους δασμούς των ΗΠΑ και περιμένουν περισσότερα από την υποστήριξη απλώς της ε, ε περιμένουν κάτι ιδιαίτερα όσοι πλήττονται στη χώρα μου στην Ισπανία και κυρίως για το ελαιόλαδο. Πρέπει και εσείς να στείλετε ένα ε, μήνυμα. Η ιδιωτική αποθήκευση δεν λειτουργεί. Η μείωση των τιμών στο ελαιόλαδο συνεχίζονται και ο συνεργατικός τομέας στην Ισπανία ζήτησε αυτορύθμιση από τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη, η οποία δεν υπάρχει. Και ε, θα πρέπει να πείτε κάτι, διότι ο τομέας του ελαιολάδου στην Ισπανία έχει ε, ο, ενημερώσει για κινητοποίηση στις 30 ε, Ιανουαρίου. Κύριε Καμπριέλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και καλώς ορίσατε, Επίτροπε. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στα καθήκοντά σας. Να έχουμε υπόψη ότι η στρατηγική για το κλίμα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ισχυρή και δυναμική προκειμένου να μπορέσουμε να τονώσουμε και τον κλάδο παραγωγής τροφίμων. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι και στον τομέα της προστασίας του κλίματος θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες καθώς και στο θέμα της ευημερίας των ζώων. Γνωρίζετε, είμαι βέβαιη, κύριε Επίτροπε, ότι θα πρέπει να σεβαστούμε και τις ανάγκες ε, του πληθυσμού που γυράσκει. στη διάσκεψη που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώσατε ότι ένας από τους στόχους σας θα είναι να καταρτήσετε μια μακροπρόθεσμη ε, στρατηγική για την Ήπεθρο. Ρωτώ λοιπόν. Τι μορφή θα λάβει, τι είδους μέτρα θα συμπεριληφθούν. Η στρατηγική αυτή θα συμπεριλάβει και τις ανάγκες των περιοχών αυτών. Αυτή η μακροπρόθεσμη λοιπόν στρατηγική για την Ήπετρο θα πρέπει να αποτελεί παράγοντα που θα λάβει μάλλον υπόψη και τις ανάγκες ε, των, ε, του κομμάτιου αυτού του πληθυσμού. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές σήμερα σε ό,τι αφορά τις άμεσες πληρωμές στα διάφορα κράτη-μέλη, σε ό,τι αφορά και τις διαφορές μεταξύ των ε, γεωργών της Ανατολής και της Δύσης. Η Πράσινη Συμφωνία θα έχει βέβαια αντικτύπο σε όλους τους ε, γεωργούς ε, σε ό,τι αφορά τη φτώχεια, σε ό,τι αφορά το διοικητικό άχθος. Αυτά θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Μιλάμε για τη μείωση των παραστακτών των και άλλων ουσιών. Αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε και μια επιτυχημένη διαδικασία μεταρρύθμισης για διάφορα κράτη-μέλη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως ε, για τους γεωργούς ε, κάποιων χωρών να μείνουν στους ίδιους ρυθμούς όταν οι άλλοι έχουν πιο πολλά χρήματα, έχουν πιο πολλούς πόρους. Θέλουμε να κάνουμε δηλαδή πιο πολλά με πιο λίγους πόρους. Αυτό ε, είναι αδύνατον. Είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη. Πείτε μας την άποψή σας. Και αυτό το θέμα της επιταχυμένης μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά την Πράσινη Συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χάζενκαμπ. Καλώ ορίσατε, Επίτροπε. Μετά τα κοτόπουλα, τα κουνέλια είναι αυτά τα οποία ε, υπόκεινται σε εντατική ε, εκτροφή και παρόλα αυτά δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία. Αν και το έχουμε ζητήσει το 2017. Θέλουμε να επιμείνουμε λοιπόν στην ε, ασφάλεια των μου, Αλλά θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σα στι άθλιε συνθήκε στι οποίε ζουν τα κουνέλια. Δεν υπάρχουν καμία επαφή με τα άλλα ζώα. Όλοι του τη ζωή την περνάνε ε, σε κλουβιά, χωρί να έχουν τρόφιμα, χωρί να έχουν νερό και στο τέλο τα θανατώνουν με πόδινο τρόπο. Στην Ολλανδία τα κουνέλια δεν ζουν τόσο άσχημα όσο στι άλλε χώρε, αλλά επιβεβαιώνουμε με εικόνε ότι ακόμα και εκεί έχουν ε, φρικτά προβλήματα ε, έχουν ε, πληγές στο σώμα τους, στα αυτιά τους και αναγκάζονται να ζουν ε, με νεκρά κουνέλια μέσα στα κλουβιά. Θα πρέπει να καταρχάς ε, να σταματήσουμε, να σταματήσουμε λοιπόν τις πρακτικές αυτές και να ξεκινήσουμε σταματώντας να τα κλείνουμε σε κλουβιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπόκοβιτς. Επιτρέπε. Ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ σήμερα Μιλάμε για μια πράσινη συμφωνία για την ψηφιοποίηση, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς και για τη μεταρρύθμιση ΚΑΠ. Έχουμε λοιπόν πιο περιορισμένους πόρους για την γεωργία και για την υπεθρό. Ενώ αυξάνονται τα οι δαπάνε για το περιβάλλον και για τη γεωργία. Ανησυχούν λοιπόν οι γεωργικοί εκτροφεί και δικαίω. Θα πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να παρακολουθήσουμε αυτή την εξυγχρονισμό σε ό,τι αφορά την ε, θέση εργασίας, ε, τον τουρισμό. Πολλοί στρέφονται σε εναλλακτικέ πηγές ε, εισοδημάτων, ενέργεια, αμα, υγεία. Το, η Πράσινη Συμφωνία περιλαμβάνει και αυτούς τους τομείς. Πώς λοιπόν θα εξασφαλίσετε ότι οι πόροι από τα άλλα ταμεία συνοχής θα φτάσουν τελικά στην Ήπετρο, θα έχουν αποτέλεσμα. Γιατί η Ήπετρος και η Γεωργία είναι τμήμα της λύσης και όχι πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι επόμενος. Η κυρία Σάντερ. ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και καλημέρα, κυρία Πετροπέ. Θα ήθελα να σα εκφράσω την ανησυχία μα όλος ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του Ταμείου για Δική Μετάβαση. Αυτό το Ταμείο το οποίο ε, ουσιαστικά πρέπει να φροντίσει τις ε, περιοχές που εξαρτώνται πιο πολύ από τα αρνητικά καύσιμα είναι σήμερα στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και βρίσκεται στην ίδια στήλη με την ε, ε, χρηματοδότηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτό το Ταμείο όντω θα βοηθήσει τα κράτη που έχουν πιο πολύ ανάγκη να υλοποιήσουν το Ταμείο αυτό για να υλοποιήσουν την Πράσινη Συμφωνία. Τι θα γίνει με τη δεύτερη στήλη. Ε, μήπως θα πρέπει να μπει στη δεύτερη στήλη με την πολιτική συνοχής. Μιλάμε για 7,5 δις ευρώ λοιπόν εδώ σε ό,τι αφορά το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στα πλαίσια της ΕΦΠ θα μπορούσατε να σχολιάσετε πώς θα γίνει δηλαδή αυτή η πράσινη συμφωνία τελικά να μην αποβεί εις βάρος της, ε, α, της Γεωργίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε διατεθειμένοι να συνεργαστείτε με το Κοινοβούλιο και σας εύχομαι καλή τύχη. Λόγω των δασμών των ΗΠΑ, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί και κυρίως οι Ισπανοί παραγωγοί συνεχίζουν να βιώνουν μια πολύ κρίσιμη κατάσταση, ε, εκατομμύρια απώλειες οικονομικές και απώλειες θέσεων εργασίας. Ε, πρέπει να υπάρχει κάποια ευελιξία για την προώθηση του ίνου και την ε, ιδιωτική αποθήκευση του ελαιολάδου που δεν ε, λειτουργήσαν. Ήταν αργή η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πότε θα δουν η παραγωγή το τέλος των δασμών. Πώς διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις ΗΠΑ. Και δεύτερον, πώς ε, θα αποζημιώσετε για τις ζημίες ε, που ε, υπέστησαν κάποιοι γεωργοί, όπως ε, η παραγωγή ελαιολάδου, που ε, προσέφηκαν στα δικαστήρια για να μπορέσουν να βρουν δικαίωση για τους δασμούς αυτούς. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή την εβδομάδα το Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απεφάφει ότι είναι παράνομη αυτή η δασμή. Ο κύριος Σοπε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Επίτροπο για την ανάλυση των καθηκόντων του. Σας εύχομαι καλή τύχη. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Ποια είναι η θέση σας όσον αφορά την πλήρη σύγκριση η κοινή αγροτική πολιτική είναι κοινή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνες και απαιτήσει είναι ίδιες για τα κράτη-μέλη, αλλά η στήριξη μπορεί να είναι και τρεις φορές διαφορετική, τριπλάσια στη διαφορά τη όταν συζητάμε κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, η στήριξη στα κράτη της Βαλτικής δεν φτάνει στο 70% τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά οι Γεωργοί έχουν προβλήματα για να επιτύχουν του στόχου και να ε, τηρήσουν τις απαιτήσει και όταν αυξάνονται οι απαιτήσει και δεν επιλύονται τέτοια προβλήματα, δεν θα μπορέσουμε να εργαζόμαστε όπως θα έπρεπε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίσατε κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ που αφιερώνετε το χρόνο σας εδώ σε εμά. Στη διάρκεια της ακρόασής σας μιλήσατε για μια κοινή γεωργική και διατροφική πολιτική και τώρα έχουμε το σχέδιο από το χωράφι στο πιάτο που είναι επιτάπητος και ε, πρόκειται ακριβώ λίγο πολύ για το ίδιο περιεχόμενο. Να προσπαθήσουμε να έχουμε μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη της και περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανησυχίες ε, στη διατροφή. Ε, οι γεωργοί αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα διότι ε, η κοινωνία αντιλαμβάνεται λίγο, ολοένα και λιγότερο τι συμβαίνει με τους γεωργούς. Ε, αυτή η πολιτική το, από το χωράφι στο πιάτο ίσως είναι μία λύση για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα σύνδεσμο με τη γεωργική πολιτική. Και πώς βλέπετε την ε, ε συμβολή της κοινή γεωργικής πολιτικής στη στρατηγική αυτή. Επίσης, ε, δεν έχουμε παροχή τροφίμων στο τραπέζι μας μόνο από τους Ευρωπαίους γεωργούς. Πώς μπορούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε τους πολίτες αλλά και τους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζωέντροβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε πίτροπε. Σας καταλαβαίνω όχι μόνο γιατί μιλάμε αντίστοιχες γλώσσες, αλλά καταλαβαίνω και τη διάθεσή σας να υποστηρίξετε τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε και την ε, οδό της ε, από συγκέντρωσης της γης από τους λίγους. Ε, και νομίζω ότι η Γεωργία είναι η πλέον εκτεθειμένη στην κλιματική αλλαγή και επομένως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε. Στις 14 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το, ε, ε, την ανακοίνωση για τα επενδυτικά της σχέδια και διαβάζουμε ότι η ΚΑΠ θα δώσει 40% των κονδυλίων του για την κλιματική αλλαγή. Μετά υπάρχει το LIFE ε, και άλλα προγράμματα, 35%. 72% του προγράμματος LIFE θα είναι αφιερωμένο στην κλιματική αλλαγή. Αλλά δεν βλέπω κάτι συγκεκριμένο για τους γεωργούς μας, για να τους βοηθήσουμε να μετριάσουν τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής ε, για τους ίδιους. Θα ήθελα λοιπόν να συμπεριληφθεί και κάτι τέτοιο. Παραδείγματο χάρη, ε, υποκατάστατα φαρμάκων ε, και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ε, υποστήριξη. Ο συνάδελφος κ. Γιάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, να, να ρωτήσω, θα συνεχίσετε έτσι σε ό,τι αφορά τις διοικητικό άγχος που θα επιβαρυνθούν ε, η εκμεταλλεύσεις. Ε, επίσης, να μην μιλάτε μόνο με τους ε, Υπουργούς Γεωργών. Το πρόβλημα είναι λίγο παρακάτω. Οι Υπουργοί Οικονομικών κλείνουν τις τσέπες τους και δεν δίνουν τίποτε. Εκεί θα πρέπει να σχέσετε πιέσεις. Κατά τρίτον, χαίρομαι με την κυνηγιαργική πολιτική που λέτε ότι θα πρέπει να καταρτήσουμε κατάλογο με μέτρα από τις Βρυξέλλες. Μια ιδέα η οποία συχνά έχει συζητηθεί εδώ στην Επιτροπή και πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί αυτή η ιδέα ω στοιχείο για τις επόμενες διαβουλεύσεις. Ε, συγκέντρωση τώρα των γεών. Να πούμε ότι θα πρέπει όλα αυτά να τα συζητήσουμε αντικειμενικά γιατί αποτελούν πρόβλημα. Σε αυτή τη στατιστική λοιπόν αναρωτιόμαστε το 3% είναι το πρόβλημα. Όταν μετράμε και τις μικρές εκμεταλλεύσεις θα φτάσουμε στο 3% και όχι στο 9%. Εδώ θα πρέπει να τα κοιτάξουμε λοιπόν όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και σας κύριε Επίτροπε. Προκειμένου να πείσουμε το Σώμα των Επιτρόπων και τα κράτη-μέλη ότι η γεωργία μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο, και μάλιστα μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην Πράσινη Συμφωνία και να υπάρχει και κατάλληλος υπολογισμός, μήπως θα έπρεπε να ε, δείξουμε και την εδαφική διάσταση κυρίως της ΚΑΠ, να συμπεριληφθεί στη βιοοικονομία για να μπορέσουμε να έχουμε και τη μετάβαση του γεωργικού κόσμου. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη δημόσια υγεία και την ανθρώπινη υγεία κυρίως. Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, ε, την οποία έχουμε ξεκινήσει από τα 2018, αντανακλά πλήρως το, η Πράσινη Συμφωνία. Και θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με την ε, αλλαγή γεών. Ε, τι σκοπεύετε να κάνετε για τη συγκεκριμένη νομοθεσία και τους κανονισμούς σχετικά. Η κυρία Μακίνες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Εγώ ανησυχώ λίγο ε, για τη διάκριση που κάνετε για τους γεωργούς μεταξύ της βιομηχανικής κλίμακας ε, γεωργίας και των οικογενειακών γεωργών. Θεωρείτε ότι είναι η ε, μεν κακή και η άλλη καλή και ξεχνάτε τους περισσότερους που είναι μεσαίας κατηγορίας που προσπαθούν να βγάλουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Αν ε, αναφέρεστε μόνο στα δύο άκρα, κάνετε διάκριση εναντίον αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται σε ενδιάμεσο. Επίσης, ε, δεν αναφέρεστε και τι λιανοϊκέ πωλήσει και στην ε, μεταποίηση. Είναι πολύ σημαντική αυτή η τομή και θα πρέπει να λάβετε υπόψη και τις πιέσει που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί λόγω της μεγάλη κλίμακας μεταποίηση. Γι' αυτό έχουμε του γεωργού στους δρόμου κυρίως για τις τιμές της αγοράς και τα χαμηλά εισοδήματα. Και εδώ δεν άκουσα να αναφέρεστε στα συγκεκριμένα θέματα. Η δεύτερη ανησυχία μου είναι η εξουσία του Επιτρόπου Γεωργίας. Φαίνεται ότι τα περισσότερα από τα καθήκοντά σας τα έχουν αναλάβει άλλοι επίτροποι. Παραδείγματο χάρη, η στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο, ναι μεν είσαστε στο τραπέζι, αλλά μάλλον δεν θα πάρετε και μεγάλη μερίδα. Και επομένως ε, ε, θα ήθελα να ξέρω και τι θα κάνετε. Θα δείτε και τα θέματα ΠΟΕ για τα φυτοφάρμακα και τρόφιμα τα οποία εισάγονται ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν απαγορευμένες ουσίες. Ο κύριο Λεμπρετό. Καλημέρα κύριε Επίτροπε. Εκτίμησα ιδιαίτερα την παρουσίασή σα και κυρίως το να ενισχύσετε την ΚΑΠ και να υπάρχουν συνέργειε μεταξύ ΚΑΠ και πολιτικής συνοχής. Υπάρχει ένα μείζον πρόβλημα που είναι η συγκέντρωση γεών και μας δώσετε ένα φρικτό ποσοστό. 3% των ε, ιδιοκτητών ε, έχουν το 50% των ε, γεωργικών γεών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα κάνετε για να αντιστρέψετε αυτή την τάση, πέραν του να ζητάτε από τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν καλύτερα το δεύτερο πυλώνα και να τον αξιοποιήσουν περισσότερο. Υπάρχουν δύο δύο πολύ μεγάλες απειλές για τους γεωργούς μας. Το πρώτο είναι η πράσινη συμφωνία που ε, σημαίνει ότι θα τους επιβάλλουν και νέες πιέσεις και αν αυτό δεν συμπεριλαμβάνει και νέα κονδύλια θα είναι φρικτές οι συνέπειες. Σημειώνω βεβαίω ότι γίνεται μια ανάλυση επιπτώσεων, αλλά δεν αναφερθήκατε στη δεύτερη απειλή, που είναι οι συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου. Και εδώ ε, έχουμε και τη δεύτερη ερώτησή μου. Τι σχέση βλέπετε εσύ μεταξύ τη ΚΑΠ και των συμφωνιών ελευθέρου εμποριών, που ε, θεωρούν ότι η γεωργία μα είναι απλώ ένα συντελεστή προσαρμογή. Πολύ ωραία. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι ερωτήσεις και τώρα ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο για να μας ε, δώσει τις απαντήσεις. Ε, τα πάμε πολύ καλά από πλευράς χρόνου. Νομίζω ότι και 20 λεπτά μπορείτε να έχετε για να δώσετε τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για αυτές τις πολλές ερωτήσεις. Ε, προσπάθησα να σημειώσω όλες αυτές τις ερωτήσεις για να μην τις ξεχάσω, αλλά ε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη αυτή εξ αρχής ε, αν κάτι μου ξεφύγει, γιατί ήταν πάρα πολλές ερωτήσεις. Κυρία Γκυλάρ. Είπατε σχετικά με τον ε, δεύτερο πυλώνα στην Αυστρία ότι αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Πρέπει να έχουμε κατά νου βέβαια και τον πρώτο πυλώνα. Έχετε δίκιο και οι δύο πυλώνε τη ε, κοινή γεωργική πολιτική είναι πολύ σημαντικοί ε, και γι' αυτό θεωρώ ότι οι γεωργοί πράγματι θα πρέπει να ασχολούνται με τη γεωργία, δηλαδή θα πρέπει να είναι και οικονομικά συμφέρον να ασχολείται κανείς με τη γεωργία και για να γίνεται αυτό χρειάζεται κάποια υποστήριξη. Ε, το θέμα είναι ότι δεν ε, μπορεί κανείς να επιβραβέσει εκείνους ε, που εφαρμόζουν τα σωστά μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Κατά τα άλλα, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και άλλες χώρες όπως η Ισπανία. Εγώ προτίθεμαι να κάνω και άλλα ταξίδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. κυρία Βίνα, εσείς αναφερθήκατε στην συγκέντρωση της γης και στα σχετικά στοιχεία. Νομίζω ότι ο κύριος ε, Λεμπρετόν έθιξε το θέμα αυτό και εκείνος το έθιξε. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, υπάρχει ένα μέτρο που μπορούμε να λάβουμε δηλαδή το κάπινγκ, το ανώτατο όριο ενισχύσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να συγκεντρωθεί η γη για να ε, να επιτευχθούν καλύτερες ενισχύσεις. Από 60.000 και πάνω υπάρχει μείωση και 100.000 ευρώ είναι το μέγιστο της ενίσχυσης που μπορεί να ε, χορηγηθεί. Και θέλω να σας πω ότι ε, επανειλημμένα εδώ στην Επιτροπή οποίοι ήμουν παρόν όταν συζητήθηκαν οι διάφορε μεταρρυθμίσεις της κοινή γεωρικής πολιτικής και εκεί υπήρξαν πάρα πολλέ προτάσεις για το ανατοτόριο. Ε, αυτό το εργαλείο τελικά δεν πέτυχε το ευκταίο αποτέλεσμα. Ε, εγώ σας στηρίζω σε αυτό το θέμα και πιστεύω βέβαια ότι οι μεγάλες επιχείρησει από ένα μέγεθο και μετά αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως βιομηχανικές και όχι πλέον ως παραδοσιακές γεωργικές επιχειρήσεις ε, και θα πρέπει να περιορίζεται η οικονομική υποστήριξη. Βέβαια υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις γιατί κάθε χώρα έχει τη δική της δομή γεωργίας. Στις περισσότερες χώρες μιλάμε για χώρες που έχουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις κάτω από 10 εκτάρια και άλλες που έχουν 130 30 εκτάρια, όπως παραδείγματος χάνει στην Τσεχία. Όσον αφορά τώρα τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη, επ' αυτού του θέματος υπάρχουν διάφορες λύσεις. Ο κ. Γιούργκελ επισήμανε ότι η Πολωνία έχει σαγάγει αρκετά περιοριστική νομοθεσία, η οποία δεν περιορίζει την αγορά γης από τους γεωργούς. Ε, όλοι οι γεωργοί θα πρέπει να έχουν την ίδια πρόσβαση, ε, δεν θα πρέπει να παίζει καθοριστικό ρόλο η θαγένεια. Ε, αυτό που θα πρέπει να παίζει ρόλο είναι κατά πόσον κάποιος είναι γεωργός ή όχι. Και νομίζω ότι επ' αυτού υπάρχει μια διαδικασία ε, από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι αρμόδια η δική μου γενική διεύθυνση για το θέμα αυτό, αλλά βεβαίως θα κάνουμε έναν απολογισμό μετά από δική σας πρωτοβουλία ε, των κρατών μελών. Για τη τελική ανάλυση αυτό που παίζει ρόλο είναι να προαχθούν μέτρα τα οποία θα μεριμνούν η γη να παραμένει στους ε, πραγματικούς γεωργούς. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για τους ε, νέους γεωργούς εξετάστηκε το θέμα αυτό εξετάστηκε το ε, ποιες ε, είναι οι αντιρρήσεις, οι επιφυλάξεις των νέων ε, που θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία. Και αυτό που προβλήθηκε περισσότερο είναι ότι δεν έχουν αρκετή γη. Βέβαια δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κερδοσκοπία με τη γη για να προσποριστεί κανείς το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Τέτοιου είδους σπέκουλες, κερδοσκοπίες. Εμείς ε, δεν τις εγκρίνουμε και γι' αυτό θέλουμε να θεσπίσουμε και τη σωστή νομοθεσία που να απαγορεύει κάτι τέτοιο. Βεβαίως και αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σαφώς και μπορεί να δει το όλο θέμα, σαφώς και μπορεί να αναφέρει επενετικά ορισμένα παραδείγματα, αλλά στη τελική ανάλυση οι ευρωπαϊκές συνθήκες δεν προβλέπουν τίποτα απολύτως για τις συνθήκες ιδιοκτησίας στα κράτη-μέλη. Ε, υπήρξε και ένα ερώτημα από την κυρία Τόμασιτς, ε, συγκεκριμένα το θέμα με τις ε, κρατικές εκτάσεις στην Κροατία. Εγώ επισκέφτηκα την Κροατία, μπόρεσα να διαπιστώσω επί τόπου το πρόβλημα και εκεί υπάρχουν δοκιμασμένες πρακτικές που μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Παραδείγματο χάρη μπορεί ε, για κρατικές εκτάσεις να προβλέπεται μακροχρόνια εκμίστοση. Αυτό το προβλέπει η Πολωνία. Ένα εκατομμύριο ένα εκατομμύριο εκτάρια κρατικής γης εκμιστώνεται σε γεωργούς γιατί αυτή τη στιγμή ε, οι γεωργοί δεν μπορούν, δεν είναι σε θέση ακόμα να αγοράσουν αυτές τις γης. Άρα δηλαδή η μακροχρόνια εκμίστοση γεών αποτελεί μια κάποια λύση. Κατόπιν ετέθη ένα ερώτημα σχετικά με τις νέες γεωργικές τεχνικές. Ετέθησαν αρκετά ερωτήματα σχετικά με τις σύγχρονες γεωργικές μεθόδους. Βεβαίως, εγώ υποστηρίζω τις νέες καινοτόμες μεθόδους ε, και την ε, δημιουργία ε, νέων καλλιεργειών ε, που να προσαρμόζονται καλύτερα στην ε, κλιματική αλλαγή. Όταν θα κατατεθούν ή αν κατατεθούν τέτοιες προτάσεις από τα κράτη-μέλη, εγώ θα τις στηρίξω, γιατί τέτοιες τεχνολογίες, παραδείγματος χάρη ε, γεωργία ακριβίας. Αυτά είναι θετικά βήματα που μπορούν να βοηθήσουν να χρησιμοποιούνται λιγότερα λιπάσματα χωρίς βεβαίως να επηρεάζεται η ε, δραστικότητα των ε, λιπασμάτων. Και με τον τρόπο αυτό περιορίζεται και η χρήση φυτοφαρμάκων. Ε, θέλω να σας πω λοιπόν ότι εγώ σαφώς και είμαι ανοιχτός απέναντι σε τέτοιες νέες πρακτικές. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να στηρίζονται σε επιστημονικά απορίσματα. Οι νέες τεχνολογίες, κυρίως οι βιολογικές ε, τεχνολογίες και οι βιολογικές καλλιέργειες προκαλούν πολλές φορές φόβο. Αυτά θα πρέπει να ε, συνοδεύονται από τεκμηριωμένη έρευνα. Πριν τελικά αδειοδοτούνται οι μέθοδες αυτοί για την πρακτική εφαρμογή. Και ο κύριος Κρίστενσεν έθεσε ένα ερώτημα προς την ίδια κατεύθυνση. Κύριε Μπούσμαν, εσείς αναφερθήκατε στη μεταφορά των ζώων. Και εγώ θλίβομαι βλέποντας αυτές τις ε, τραγικές εικόνες ε, κατά τη μεταφορά των ζώων. Και γενικότερα η κοινή γνώμη θλίβεται και αγανακτεί. Και πολλοί λένε ότι φταίνει η γεωργή. Μα δεν φταίνε οι ε, για τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται τα ζώα στη Μεσόγειο ή οπουδήποτε αλλού. Αυτές είναι βιομηχανικές μονάδες ε, που δεν διασφαλίζουν καλές συνθήκες. Γι' αυτό λοιπόν προφανώς ε, και χρειαζόμαστε καλύτερους ελέγχους για τις ε, ε, μεταφορές των ζώων. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις. Ένα δεύτερο βήμα που είναι εξίσου σημαντικό για μένα είναι η δημιουργία εναλλακτικών λύσεων έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να υπάρξουν αυτές ε, τέτοιου είδους μεταφορές. Παραδείγματο χάρη ε, υποστήριξη μονάδων που προμηθεύουν τις τοπικές αγορές. Ίσως τον δεύτερο πυλώνα μπορούμε να δώσουμε κίνητρα ο γεωργός, ε, ο κτηνοτρόφος ε, να έχει κίνητρα να προσφέρει τα προϊόντα του στην τοπική αγορά. Και κατόπιν τα ζώα να αγοράζονται στην τοπική αγορά χωρίς να πρέπει να μεταφερθούν. Στην περίπτωση αυτή κάνουμε εξοικονόμηση στις ε, μεταφορές και στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας νομίζω ότι μπορούμε να στηρίξουμε κάτι τέτοιο είναι μια ικανοποιητική εναλλακτική λύση για ε, μεταφορά ζών σε μεγάλες αποστάσεις. Εγώ θα στηρίξω ε, τέτοιου είδους προτάσεις στα νέα εθνικά στρατηγικά προγράμματα. Κύριε Γιούργελ, νομίζω ότι απάντησα ήδη στην ερώτησή σας. Εσείς κάνατε βέβαια και άλλη μία ερώτηση που αφορά στις ε, συμβάσεις, στις συνθήκες και στη μεταβατική περίοδο. Ελπίζουμε βέβαια να τα καταφέρουμε, να εγκρίνουμε τις μεταρρυθμίσεις έγκαιρα. Όλα αυτά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις για το πολιτές σε δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζω όμως ότι θα καταφέρουμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο ε, χρονικό διάστημα, σε ένα χρόνο νομίζω, ε, η κοινή γεωρική πολιτική να ξεκινήσει με τις νέες προϋποθέσεις ο κύριος Ρούσεν και εκείνος έθιξε το θέμα των νέων γεωργικών τεχνολογιών. Απάντησα στο θέμα αυτό. Θέλω βέβαια να προσθέσω κάτι που είπα και κατά διάρκεια των ακροάσεων, κάτι το οποίο επιθυμώ να επαναλάβω. Όταν θα εγκριθεί το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, τότε θα έχουμε και τα απαραίτητα κονδύλια για την γεωργική έρευνα, τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, ε, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ευφυώς, έτσι ώστε να έχουμε έρευνα που πραγματικά να εξυπηρετεί ή να υπηρετεί τη γεωργία και να οδηγεί σε πρακτικές λύσεις. Δηλαδή το θέμα δεν πρέπει να είναι να διεξάγουμε μόνο θεωρητική έρευνα, αλλά και στην πράξη ε, να ελέγχουμε την αποδοτικότητα της γεωργίας κατά πόσο είναι φιλική προς το περιβάλλον. Ε, με τα κονδύλια νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε πάρα πολλά. Κυρία Κατάινεν, πολύ σωστά μας ε, είπατε ότι οι γεωργοί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τμήμα της λύσης και όχι ως τμήμα του προβλήματος. Γιατί πράγματι Πολλές φορές αναφέρεται ότι οι γεωργοί ε, φέρουν την ευθύνη και αν δεν υπήρχαν αυτοί δεν θα υπήρχαν προβλήματα. Όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας πρέπει να ξεκινούν από την πεποίθηση ότι οι ε, γεωργοί πρέπει να έχουν κίνητρα για να εφαρμόζουν τις νέες απαιτήσει. Βεβαίως και η γεωργία πρέπει να γίνει πιο φιλική προς το περιβάλλον, αλλά η γεωργία και αυτή ε, πρέπει να προσαρμοστεί γιατί χωρίς τους γεωργούς ε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε περίπου 10 εκατομμύρια γεωργούς στην Ευρώπη οι οποίοι προσφέρουν τα τρόφιμα σε περίπου 500 εκατομμύρια πολίτες και γι' αυτό το λόγο πρέπει να επιδεικνύουμε σεβασμό απέναντι στους γεωργούς. Είναι μια ομάδα που συνεχίζει να συρρυκνώνεται χρειάζεται την υποστήριξή μας ε, για να μπορούμε να διασφαλίσουμε την ε, ασφάλεια τροφίμων στο μέλλον. Ε, πολλοί συνάδελφοι επισήμαναν, πολλοί ευρωβουλευτές επισήμαναν ότι πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός και εγώ Είπα στην αρχή πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ο κύριος Γιάρ είπε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε με τους Υπουργούς Οικονομικών γιατί οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται πάντα και μόνο από τους Επιτρόπους Γεωργίας. Και εγώ ξέρω πώς γίνονται, πώς λαμβάνονται αποφάσεις ε, στα κράτη ε, και εγώ ε, στο Σώμα των Επιτρόπων είμαι υποστηρικτής της Δεν είναι βέβαια όλοι οπαδοί αυτής της άποψης και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις. Ακόμα βρισκόμαστε σε διαπραγματευτική φάση, υπάρχουν όμως διάφορες προτάσεις τις οποίες μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας για να δούμε πώς θα κατανείμουμε τα κονδύλια δίκαια έτσι ώστε στο τέλος να υποφεληθούν όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ε, μόνο νικητές και ετοιμένοι, να παίρνουμε από τους μεν για να τα δίνουμε στους δε. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται. Και τέλος, νομίζω ότι θα πρέπει ε, να συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη. Ε, βέβαια, σημείο πρέπει να είναι η αύξηση του προϋπολογισμού. Και βεβαίως αυτό που ενδιαφέρει επίση είναι και η δίκαιη ε, κατανομή. Κύριε Γκερέιρο, εσείς ε, αναφερθήκατε στους ε, New York Times, στα άρθρα που διαβάζει κανείς την εφημερίδα αυτή και εγώ πρέπει να σας πω ότι στενοχωρήθηκα πάρα πολύ για την κριτική στην κοινή γεωργική πολιτική. Εκεί αναφέρονται καταχρήσεις Πολύ συχνά αναφέρεται ότι τα γεωργικά κονδύλια διασπαθίζονται Έχουμε όμως την Όλαφ ένα θεσμό ο οποίος παρεμβαίνει οποτεδήποτε εντοπίζονται απάτες με κοινωτικά ή ενωσιακά κονδύλια. Εμείς ε, βέβαια θέλουμε να συστήσουμε και ένα κατάλογο προληπτικών μέτρων έτσι ώστε στα εθνικά στρατηγικά προγράμματα να υπάρχουν σαφείς κανόνες παραδείγματος για την κατανομή των κονδυλίων έτσι ώστε να υπάρχουν τα ίδια κονδύλια για όλους και να μην ε, αναγκαστούμε ε, να εφαρμόσουν αρχή ε, όποιος πρόλαβε. Όχι, εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό ίδιοι οι κανόνες, ίδια κριτήρια να επιλέγονται τα καλύτερα ε, προγράμματα οποτεδήποτε πρόκειται για ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων. Έχω κατά νου ένα κατάλογο με προληπτικά μέτρα έτσι ώστε να προλάβουμε δυνατόν τη διαφθορά και την απάτη. Κυρία Κιλέρα, μιλήσατε για το χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία προτείνονται Για μένα αυτό που είναι καθοριστικό είναι τα εθνικά σχέδια. Και με... μιλάμε για μια παράταση της μεταρρύθμισης και τα στρατηγικά σχέδια λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε να εμπεριέχουν επαρκή σχέδια για την προστασία του κλίματος. Φυσικά μιλάμε για την προστασία επία και της νοσοκομείας και της βιοπικιλότητας. Η νοσοκομεία, λοιπόν θα πρέπει σίγουρα να προετοιμαστεί ως σκέλος της στρατηγικής αυτής. Κατά τα θα υπάρξουν νομοθετικές προτάσεις οι οποίες θα κινηθούν προς άλλες κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, αυτά τα τόνισε και η Επίτροπος για την Υγεία και στο πλαίσιο αυτό να απαντήσω και άλλη μια ερώτηση σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του ε, Επιτρόπου Γεωργίας. Η κυρία Μαγκίνης έκανε την ερώτηση νομίζω και κατά πόσο περικόπηκαν οι αρμοδιότητες. Μία αρμοδιότητα αφαιρέθηκε ε, οι κρατικέ επιβοτήσει που ήταν παλιά στον τομέα τη γεωργία, υπήρχε λοιπόν ένα τμήμα το οποίο ασχολούταν με τι με τις κρατικέ επιβοτήσει. Πλέον έχει μεταφερθεί αυτό στον τομέα αρμοδιότητα τη ανταγωνιστικότητα. Δεν έχουν αλλάξει όμω οι αρμοδιότητε. Ουσιαστικά πάντα τα θέματα ευημερία των ζώων, των φυτοπροστατευτικών ήταν πάντα σε άλλη α, γενική διεύθυνση, όχι στη γεωργία. Και όταν το Ελεκτρικό συνέδριο έκανε του κρατικού ελέγχου, Ακόμα και σε ό,τι αφορά τον τομέα της γεωργίας, ουσιαστικά ο Επίτροπος Υγείας ήταν πάντα ο ομολογός μου για τέτοια ζητήματα σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα. Η πρόεδρος ε, μου λέει να ολοκληρώνω σιγά σιγά, αλλά να απαντήσω και την ερώτηση του κυρίου, της κυρίας Αμάρο σε ό,τι αφορά τις μικρές ε, ε, εκμεταλλεύσεις και την πολιτική συνοχή. Θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα σημαντικό διαχωρισμό από τις ε, πόρους ΚΑΠ δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται ε, μέτρα τα οποία θα καταργούν τη γεωργία. Αυτό υπήρχε και στο παρελθόν σε ό,τι αφορά την ανάληψη νέα, δηλαδή δραστηριότητα οικονομική. Δεν μπορούν να καταβάλλονται πόροι από τα αγροτικά ταμεία. Ασφαλώ είναι σημαντικό να υποστηριχθούν τα άτομα αυτά που επιθυμούν να κάνουν την αλλαγή αυτή, αλλά να στραφούν στην πολιτική συνοχή. Αυτή προβλέπεται για τα μέτρα αυτά. Τότε όταν κάποιος εγκαταλείπει τον τομέα της γεωργίας θα πρέπει να στραφεί στην ε, πολιτική συνοχή, στα ταμεία περιφερειακής ανάπτυξης και όχι στα γεωργικά αυτά μέσα, τα οποία πρέπει να εξυπηρετούν τους σκοπούς της γεωργίας. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε το διαχωρισμό αυτό. Και είμαι βέβαιο ότι θα πετύχουμε μία α, συμφωνία. Σα ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρο που μακρηγόρησα. Να σα ευχαριστήσω όμω για τα πολύ άριθμα και πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα και είμαι διαρκώ ε, στην διάθεσή σα. Σκοπεύουμε να κάνουμε και σχετικές αναλύσεις και εγώ θα έρθω σε επαφή μαζί σας ε, εφόσον έχω επιπρόσθετες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις, για παράδειγμα, της Πράσινης Συμφωνίας ε, στην ΚΑΠΑ όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες και αξιολογήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Θεωρώ ότι ήταν καλή ε, αρχή και σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας πραγματικά έχουμε να σχολιάσουμε ότι κάνατε προσπάθεια όχι να αποφύγετε τις ερωτήσεις αλλά πραγματικά στην ουσία τους να τις απαντήσετε. Γι' αυτό λοιπόν προσβλέπω στη μελλοντική μας συνεργασία και αυτό χρειάζεται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ό,τι αφορά τις ανάγκες των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ και πάλι. Thank you.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 So, dear colleagues, we should continue. Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε παρακαλώ. Yeah. so, dear colleagues, please take your seat. Καθίστε, συνάδελφοι, παρακαλώ. Yeah. my. my... <laughs> Μάλιστα, να προτείνουμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Χάσαμε λίγο χρόνο, αλλά νομίζω ότι καλό ήταν να δώσουμε και στον Επίτροπο το χρόνο που χρειάστηκε για να απαντήσει τα πολύ αριθμά ερωτήματα τα οποία ετέθησαν. Να περάσουμε στο 16 της ημερησίας, εντάξει, σε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε το νέο μοντέλο προμηθειών και όχι μάλιστα επιφανειακά, αλλά λίγο πιο εντελεχώς και να καλέσουμε εδώ εμπειρογνώμονες, γιατί υπάρχουν διάφορα μοντέλα υλοποίησης, κεντρικά μοντέλα, περιφερειακά μοντέλα, υβριδικά έτσι, ανάμεικτα μοντέλα υλοποίησης και έτσι λοιπόν Έχουμε μαζί μας ε, τους προσκεκλημένους μας, οι οποίοι θα έχουν από 10 λεπτά ο καθένας στη διάθεσή του από τα κράτη-μέλη να μας παρουσιάσουν ποιες είναι οι σκέψεις τους και οι ανησυχίες τους. Μετά θα ακούσουμε τους συζητητές και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους ε, συναδέλφους. Ο κ. Μπακόφσκι καταρχάς θα μας παρουσιάσει την ε, πολωνική αρχή πληρωμών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι. Μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα στην Επιτροπή σας και να σας πω δύο λόγια για την υπηρεσία για την επαναδιάρθρωση και την εξυγχρονισμό της γεωργίας. Πρόκειται για μια τριπλή α, δομή Έχουμε καταρχάς την κεντρική υπηρεσία. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό μιλάμε για το 10% του συνόλου της υπηρεσίας. Στη συνέχεια έχουμε τα περιφερειακά γραφεία, τα τοπικά γραφεία. Εδώ σε επίπεδο προσωπικού είμαστε στο 34% του συνόλου και στο χαμηλό, πιο χαμηλό επίπεδο, το τοπικό επίπεδο, έχουμε και τα τοπικά γραφεία που αντιπροσωπούν το 55% του προσωπικού μας. Η υπηρεσία μας λοιπόν για την ε, αναδιάθρωση απασχολεί 11.000 υπαλλήλους στην Πολωνία σε όλα αυτά τα γραφεία όπως σας τα ανέφερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα της υπηρεσίας, να σας πω ότι έχουμε διάφορα καθήκοντα. ό,τι αφορά την υλοποίηση πληρωμών στα πλαίσια της ΚΑΠ και της κοινή αλευτικής πολιτικής και οι δύο πολιτικές λοιπόν υλοποιούνται από το ίδιο προσωπικό το οποίο επιτεκνύει κάποια ευελιξία Μιλάμε λοιπόν κυρίως για τον πρώτο πυλώνα, για τις άμεσες πληρωμές. Έχουμε όμως και ε, προγράμματα υποστήριξης της αλίας και της γεωργίας. Ύστερα έχουμε και το Ίδρυμα το οποίο παρέχει τα, τις υπηρεσίες που παρέχουν ε, εθνικές επιδοτήσεις. Ε. Λαμβάνουμε κάποιες εθνικές επιδοτήσεις για να παρέχουμε υποστήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που πλήττονται από την ξηρασία, για παράδειγμα, ή για την υποστήριξη, για παράδειγμα, των γυναικών γεωργών, προώθηση των παραδοσιακών μορφών γεωργίας. Ε. Έχουμε επίσης ε, συστήματα καταχώρησης των ζώων, το σύστημα RAS ε, για την απερίμωση των χωραφιών, θέματα δορυφορικών απεικονίσεων, μητρό παραγωγών και εκτροφέων, μητρό δηλαδή, που περιέχουν όλους όσους υποβάλλουν αιτήσει στην υπηρεσία μας. Το 2017 ήμασταν η μοναδική υπηρεσία καταβολής τέτοιων πόρων στην Πολωνία που παρήχε πόρους και κονδύλια στους γεωργούς. Είχαμε και την υπηρεσία γεωργίας που ήταν ξεχωριστή υπηρεσία. Πλέον έχουμε ενοποιηθεί και έτσι λειτουργούμε πιο ομαλά. Αυτό ήταν πραγματικά μια μεγάλη επιτυχία για μας. Από οικονομική άποψη. να πούμε τα εξή. Η υπηρεσία μας ε, λειτουργεί εδώ και 25 χρόνια. Πέρσι είχαμε την επέτειό μας αυτή την 25η και έχουμε περίπου δηλαδή καταβάλει 80 δις ευρώ αυτά τα χρόνια. Κοιτώντα το ημερολόγιο από το 1994 μέχρι το 2003 ως τμήμα του Γενικού Προπολογισμού είχαμε καταβάλει 3,6% και όταν φτάσαμε στο επίπεδο αμεσοπληρωμών ξεκινήσαμε να υλοποιούμε και να δίνουμε μεγάλα ποσά 96% αύξηση μέχρι το 2019 Πιστεύω ότι στο σημείο αυτό, ε, στην διαφάνεια αυτή, μπορείτε να δείτε και τις πιο σημαντικές σύμφορες 23% άμεσα, συστήματα άμεσων ενισχύσεων. Αυτό περιλαμβάνει και την ευμερία των ζώων, την προστασία της βιοπικιλότητας. Όλα αυτά μπαίνουν στο κεφάλαιο του συστήματος άμεσων ενισχύσεων. Στους επόμενους δύο πυλώνες βλέπετε τα προγράμματα ανάπτυξης πέθρου και λοιπά προγράμματα. Και προγράμματα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί σε ό,τι αφορά το νέο μοντέλο υλοποίηση και το πώ ε, ε, επηρεάζει την υπηρεσία μας. Το στρατηγικό σχέδιο ε, ζητά να προγραμματιστούν δύο πυλώνες για να υπάρχει συνέχεια στους ε, πόρους και στα κονδύλια. Είναι σωστή αυτή η λύση, γιατί από διοικητική πλευρά θα είχε νόημα να συνενωθούν οι δύο αυτές πτυχές, προκειμένου να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός και να γίνονται πιο σωστά και γρήγορα οι πληρωμές, να υπάρχει επίσης και εισαγωγή πιο ευέλικτων κανόνων για την ε, διαχείριση της ΚΑΠ. Αυτό μας βρήκε σύμφωνος λοιπόν κάποιοι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι έχουν υλοποιηθεί έχουν ε, αφιτερήτρα ε, εθνικών δομών και αυτό ήταν σωστό και είχε σωστά αποτελέσματα στην Πολωνία, γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητε στην ε, Πολωνία. Και έτσι λοιπόν χρειάζεται αυτή η ευελιξία για να έχουμε περιθώριο ελιγμού. Έχουμε τώρα και την αρχή της ε, βιώσιμης και σύγχρονης ε, γεωργίας σύμφωνα και με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Κλιματικής Πολιτικής και της Πράσινης Συμφωνίας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τις διάφορες περιοχές με βιώσιμο τρόπο. Έχουμε λοιπόν ε, τοπικές ιδιαιτερότητες στην Πολωνία. Κάποιες περιοχές χαρακτηρίζονται από μεγάλες εκτάσεις, πολλών εκταρίων, πολλές, μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Στο νότο της Πολωνίας η, τα αγροκτήματα είναι κατακαιρματισμένα και πιο μικρά ε, σε έκταση. Θα πρέπει λοιπόν αυτές τις εκμεταλλεύσεις 4-5 εκταρίων κατά μέσο όρο να τις υποστηρίξουμε με το σωστό τρόπο να υπάρξει μια βιώσιμη προσέγγιση προκειμένου να μπορέσουμε να κατανέμουμε τελικά τα κονδύλια με σωστό και αποτελεσματικό τρόπο και να καλύψουμε όλο το φάσμα των ιδιαιτεροτήτων. Υπάρχει η ψηφιοποίηση, οικολογικέ, οικολογικές όλα αυτά προφανώ αποτελούν σημαντικά ζητήματα τα οποία θα αποτελέσουν προκλήσεις του μέλλοντο. θα πρέπει η ψηφιοποίηση να υλοποιηθεί με σωστό τρόπο, να αλλάξει ο τρόπο λειτουργία μας. Χρειάζεται να αυτοματοποιηθούν πολλές διαδικασίες και διεργασίες και στο νέο πρόγραμμα θα προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα συμπεριλάβουμε και να τα λάβουμε υπόψη μας. Σε ό,τι αφορά τώρα τις προκλήσεις, θα τις αφήσω ίσως στο τέλος. Να περάσουμε καταρχάς στην επόμενη διαφάνεια για να δείτε ποια είναι η ιδέα των δράσεων βάση απόδοσης. Συμφωνούμε, συμφωνούμε με την αντίληψη αυτή, με την ιδέα αυτή. Και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων των δράσεων ε, σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ναι, λέει ο πρόεδρος, αν θέλετε παρακαλά να μιλάτε λίγο πιο αργά, να σας παρακολουθούν και οι δερμηνείς, Βεβαίω. Να εξασφαλίσουμε λοιπόν την σωστή εφαρμογή των μέτρων και τον έλεγχο των δαπανών. Χρειάζεται λοιπόν μια τέτοια φιλόδοξη προσέγγιση. Την καλωσορίζουμε. Και θα θέλαμε να είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τις επενδύσεις. Να υπάρχει αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά τις δαπάνες. Να υπάρξει λοιπόν η προσέγγιση αυτή και με τον τρόπο αυτό θεωρώ ότι θα έχουμε τις δράσεις όπως τις χρειαζόμαστε. Ένα σημείο μας ανησυχεί. Θεωρούμε ότι η δημιουργία δράσεων καλύπτει ένα μοντέλο. Προσπαθούμε λοιπόν να αναπτύξουμε ένα κριτήριο όπου θα προσπαθήσουμε τελικά να πετύχουμε να προσεγγίσουμε τους ε, σωστού δικαιούχους. Δεν ξέρουμε όμως τελική ανάλυση κατά πόσο θα είμαστε σε θέση να πετύχουμε το σωστό αριθμό αιτήσεων. Ενδεχομένω να υπάρχουν κάποιοι νέοι όροι οι οποίοι θα ισχύουν, μα ανησυχούν όλα αυτά στην διαδικασία. Έχουμε κατά νου και τις νέες δράσεις οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν και προσπαθούμε να δούμε πόσες εφαρμογές ενδεχομένω να υφίστανται και πόσα χρήματα ενδεχομένω θα μπορέσουμε να χορηγήσουμε. Είναι σωστό λοιπόν που υπάρχει φιλοδόξη η προσέγγιση. Έχουμε κάποιες ανησυχίε, αλλά εν γέννη μα αρέσει η ιδέα. Τώρα, στα θέματα ευελιξίας. Εδώ έχουμε κάποιες στατικές πτυχές. Δυνατότητα επιλογής τύπων παρέμβασης, για παράδειγμα. Λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες του κρατών μελών. Αυτό θα καταστήσει τις δράσεις μας και πιο αποτελεσματικές. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να οριστούν οι όροι και οι συνθήκες σε τοπικό επίπεδο. μιλώντας για αρτική δράση την ε, γη και όλα αυτά θα πρέπει να οριστούν στο εθνικό επίπεδο γιατί προφανώς στα διάφορα κρατημέλη υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες. Μιλάμε επίσης για τον ορισμό των ε, κριτηρίων νομιμότητα σε επίπεδο κρατών μελών. Όλα αυτά λοιπόν μας βρίσκουν σύμφωνους, τα καλωσορίζουμε. Επίσης το θέμα των ε, κυρώσεων και των ελέγχων. Θεωρούμε ότι η έλεγχοι αυτή στην Πολωνία θα πρέπει να επιλέγονται με σωστό τρόπο. Και τώρα να περάσουμε στην τελευταία διαφάνεια. Και να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η υπηρεσία μας. Ψηφιοποίηση. Εδώ προετοιμαζόμαστε να καταρτήσουμε ένα καινούργιο πρόγραμμα με ψηφιακό τρόπο προκειμένου να υπάρξει πλήρης ψηφιοποίηση στην υπηρεσία μας. Δεν ε, θα ξεφύγουμε από αυτό. Έχουμε προετοιμάσει μια σχετική στρατηγική η οποία και εφαρμόζεται. Στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά τις δορυφορικές εικόνες, ε, συστήματα εξαποστάσεως όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Θέλουμε όμως να προωθηθούν περαιτέρω. Θέλουμε και τέτοιες περιοχές ε, να περιληφθούν και το θέμα της ανάλυσης ε, των περιοχών, ε, τα θέματα της ξηρασίας, οριζόντιες ε, εφαρμογές, συστήματα ενίας εφαρμογής για τους νέους δείκτες. Έχουμε μία βάση δεδομένων, όπως λέγουμε τα δεδομένα από όλη την υπηρεσία. Τα δεδομένα αυτά στη συνέχεια παίρνουν από εξεργασία και μπορούν να διαβιβαστούν και καταρτίζονται ειδικέ εκθέσει. Και επίση ε, ε, παρακολουθούμε τι νέε διαδικασίε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, και να προχωρήσουμε το κύριο. Πολύ ωραία. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ριμπέρο, που είναι πρόεδρο ε, του Οργανισμού Πλεωμών στην Πορτογαλία. Κύριε Ριμπέρο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση είναι ε, αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σημαντική ε, πολύ κρίσιμη η περίοδος στην κοινή γεωργική πολιτική και είμαι σίγουρος ότι αυτή η Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής, άρα δηλαδή θα υπάρξει ε, κάποια μετακίνηση στο σύστημα. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και θετικά ε, στοιχεία του όλου θέματος. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μοντέλο είναι ένα καλό μοντέλο. Είναι ένα μοντέλο που κατά την άποψή μας ε, θα προτείνει νέες λύσεις, διότι αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα υπάρξουν όλο και περισσότερες απαιτήσει σχετικά με το τι αποδίδουν τα χρήματα που επενδύονται. Παλαιότερα ε, ε, επενδύαμε, ήταν σημαντικό το τι επενδύσεις γίνεται, τώρα όμως είναι σημαντικά τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά για τους φορολογούμενους, ε, για τους γεωργούς και γενικότερα για την ευρωπαϊκή στρατηγική. Αυτό το μοντέλο είναι αυτό που σας παρουσιάζουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον ε, άκουσα τις ε, παρατηρήσεις ε, που έγιναν προηγουμένως. Ακούσα τι ελέγχθη για το θέμα των πληρωμών. Αυτό λοιπόν που διαπιστώνουμε είναι ότι μερικές φορές υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν γίνεται απορρόφηση κονδυλίων ή λάθος χρήση των κονδυλίων από την κοινή γεωργική πολιτική. Για μας λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ε, και ίσως και ακόμα πιο σημαντικό να γίνεται κοινή χρήση και καλή χρήση των κονδυλίων. Μερικές φορές το θέμα της κατάχρησης κονδυλίων είναι απλά ε, ένας μύθος που κυκλοφορεί. Πολλές φορές ε, στη χώρα μας διαπιστώνουμε ότι η κοινή γνώμη οι εφημερίδες και οι εξωτερικοί παρατηρητές ε, φύγουν αυτό το θέμα της ε, ε, κακής διαχείρισης των κονδυλίων, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι τελικά δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Δεν προκύπτει αρκετή προστέμενη αξία για τα χρήματα που δαπανώνται. Σε γενικές γραμμές η κοινή γεωργική πολιτική ήταν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην υποστήριξη των γεωργών και των γεωργικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ συχνά όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν καταστάσεις όπου ναι, ε, τηρούνται οι κανόνες, όμως τα αποτελέσματα δεν προκύπτουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Δεν είναι ακριβώς αυτό που επιθυμεί ο φορολογούμενος. Πιστεύουμε λοιπόν αυτό το νέο μοντέλο που βασίζεται στην απόδοση είναι ένα καλό μοντέλο, το στηρίζουμε, αλλά βεβαίως για να είμαστε απόλυτα θετικοί πρέπει και να ε, το συνοδεύσουμε με κάποιες ε, προϋποθέσεις. Και εδώ υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω. Πρώτον, ε, αποτελεσματική απλούστευση. Γνωρίζουμε ότι η απλούστευση είναι σημαντική, διότι πολλές φορές οι δικαιούχοι αγωνίζονται να ε, τηρήσουν τους κανόνες. Και μερικές φορές υπάρχει ε, παρανόηση σε επίπεδο δικαιούχων ή επιβάλλεται ε, επιπρόσθετο και ιδιαίτερο βάρος στους δικαιούχους που προσπαθούν να συμμαρφωθούν. Είπα και προηγουμένως υπάρχει αυτή η άποψη περί ε, κακοδιαχείρισης των κονδυλίων και έτσι αυτη η αποψη περι κακοδιαχειρισης των κονδυλιων και ετσι καταληγουμε στο εξής. Όταν το ελεγκτικό συνέδριο εξετάζει την κατάσταση και μερικές φορές εστιάζουν σε ε, κάποια θέματα που αφορούν στον κεντρικό πυλώνα της κοινή γεωργικής πολιτικής σε θέματα συμμόρφωσης. Αυτό που επισημαίνουν πολύ συχνά είναι ότι όταν ε, τα μέτρα από τον πρώτο πυλώνα είναι σχεδόν ασήμαντα, είναι ότι πολλές φορές τα, πρώτα, τα κονδύλια από τον πρώτο πυλώνα είναι αμεληταία σε σχέση με αυτά του δεύτερου πυλώνα. Στον πρώτο ε, πυλώνα δεν υπάρχει συγχρηματοδότηση, είναι χρηματοδότηση 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο δεύτερο πυλώνα προβλέπεται συγχρηματοδότηση ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη-μέλη. Αυτή είναι η διαφορά, έτσι εξηγείται αυτή η διαφορά. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει συνυπευθυνότητα, ε, προκύπτει και τελείως ε, διαφορετική προσέγγιση. Ε, οι κανόνες είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν για τις εταιρείε και για τους γεωργούς αυτό το δεύτερο πυλώνα όπου προβλέπεται κοινή διαχείριση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτό που πρέπει να εξετάσουμε συχνά είναι ότι υπάρχει η επικουρικότητα και εάν υπάρξει έντονη επικουρικότητα θα επανεθικοποιηθεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επικουρικότητα είναι μια επικουρικότητα η οποία στρατηγικά είναι ε, προσαρμοσμένη, εμπλουτίζεται με σαφείς στόχους ε, που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και επιθυμεί να επιδιώξει. Πρόκειται για συγκεκριμένους στόχους που έχουν καθοριστεί και αυτοί οι στόχοι συμβαδίζουν με την επικουρικότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές δεν πρόκειται μόνο για το πώς κατανοούμε αυτό. Αυτό που εξετάζουμε είναι πώς μπορούμε να προσφέρουμε στόχους σε περιοχές που, είναι, που έχουν παρεμφερεί στόχους, που θέλουν να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των ανθρώπων. Παραδείγματο χάρη στην Πορτογαλία γνωρίζουμε ότι το θέμα δεν είναι οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις αλλά οι μικρές εκμεταλλεύσεις. Και θα σας πω κάτι που νομίζω ότι ε, το γνωρίζετε πολύ καλά. Σε μικρές ε, χώρες ε, έχουμε περίπου 800 δικαιούχους της κοινή γεωργικής πολιτικής 700.000 μάλλον και οι 50.000 ε, έχουν κάποια σχέση με τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δηλαδή ένας τομέας της γεωργίας που είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν που υπάρχει αλλού. Άρα δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει κάποια ευελιξία, ε, τουλάχιστον στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την ε, πραγματικότητα. Και βέβαια ξέρουμε ότι άλλοι οφείλουν να έχουν μια ε, διαφορετική προσέγγιση. Αν δούμε λιγάκι τώρα τη σχέση κόστους-οφέλους ε, και το διοικητικό, τη διοικητική σχέση, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι στο νέο μοντέλο υπάρχει κάτι ε, που είναι σαφές. Η προσέγγιση βασίζεται σε απόδοση, είναι μια προσέγγιση που βασίζεται στην απόδοση απλούστευση της ε, γεωργικής ε, πολιτικής, ε, συγχρηματοδότηση. Αυτά όλα δεν βασίζονται στις δαπάνες, αλλά στα χειροπιαστά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται και που μπορούν πολύ εύκολα να εντοπιστούν, παραδείγματος χάρη, απόδοση της παραγωγής Αυτά λοιπόν βασίζονται στα αποτελέσματα και όχι μόνο στις δαπάνες. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο διευκρινίζουμε την κατάσταση και όλα αυτά είναι και ένα κίνητρο για όσους συμμετέχουν στη διαδικασία. Και γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι όσοι συμμετέχουν ε, θα συμμετέχουν και στο ότι τα χρήματα δαπανώνται σωστά. Άρα δηλαδή όταν τα συστήματα είναι αυτοματοποιημένα Έχουμε πληρωμές που βασίζονται σε κανόνες. Αυτά όλα γίνονται ψηφιακά και νομίζω είναι απόλυτα σαφές ότι η ψηφιοποίηση οδηγεί σε μεικτά αποτελέσματα. Όλα αυτά δεν είναι απλά. Η διαλειτουργικότητα είναι ένα σημαντικό θέμα. Είναι σημαντικό να προστεύεται η ιδιωτικότητα όσων συμμετέχουν στην κοινή γεωργική πολιτική και υπάρχει και βέβαια το θέμα της ε, διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα βρεθούν ε, κάποιες λύσεις σε αυτά τα προβλήματα και όλα αυτά πρέπει να γίνουν ε, Ωστε το δυνατόν νωρίτερα, έτσι ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργική ή διαλειτουργικότητα. Τώρα θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω. Θα ήθελα απλά να πω ότι αυτή η αλλαγή στην προσέγγιση είναι απολύτως απαραίτητη έτσι ώστε να μειώσουμε το διοικητικό κόστος, να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ε, τα χρήματα να κονδύλια, τα κονδύλια να χρησιμοποιούνται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και Επίσης, να μπορούμε να προσφέρουμε κάτι το χειροπιαστό σε αυτούς που ζητούν απλούστευση και ζητούν να έχουν περισσότερο μετρήσιμη στόχη. Με αυτό το σημείο θα ήθελα να ολοκληρώσω με αυτή την παρατήρηση και νομίζω ότι το σημαντικότερο όλων ήταν ότι εγώ θέλησα να πω η ε, προσαρμογή είναι πολύ σημαντική, τουλάχιστον όσον αφορά την Πορτογαλία και πρέπει να ακολουθήσουμε απαρέγκλητα αυτή την κατεύθυνση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη δυνατότητα. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ριμπέρο και περνάμε τώρα στους ε, περιφερειακούς οργανισμούς πληρωμής. Ο κύριος ε, Φαμπρίτσιο Στέλλα, ο οποίος είναι διευθυντής του Οργανισμού Πληρωμής της Βενετίας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους. Είναι τιμή μου να σας παρουσιάζω την υπηρεσία μας ε, εδώ. Θα σας εξηγήσω λίγο το ρόλο μας ε, στο εσωτερικό της περιοχής του Βένετο για να σας εξηγήσω λίγο καλύτερα τα καθήκοντά μας και τη δομή μας. Η περιοχή του Βένετο είναι ιδιαίτερα ετερογενή από πλευρά εδαφική. Έχει μια ορεινή περιοχή. Έχουμε την περιοχή των Δολομητών, θα γνωρίζετε. Έχουμε βοσκότοπους και επίσης υπάρχει και ε, ξυλία, μάλιστα καλή ποιότητα. Έχουμε μόνισμους ε, βοσκοτόπους, ε, μεγάλες ζωοτεχνικές παραγωγές. Υπάρχουν 97.000 εκτάρια μπελώνων επίσης έχουμε πολύ καλή παραγωγή, ηνική παραγωγή, το αμαρόνε, το λόλιο, το βελγάτα και επίσης είναι μια περιοχή ιστορικής σημασίας, πολλές περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και έχουμε και τις παιδινές περιοχές με μεγάλη παραγωγή. Έχουμε αραβοσίτη, σόγια, ρύζι, ε, Abbiamo le specie di maggior rilievo invece... Pazzaria. Eh, και επίσης έχουμε ε, φρούτα, κίβι, ε, ακτινίδιο, ε, ροδάκινα κλπ. Έχουμε επίσης μαρούλια και το πολύ διάσημο μαρούλι του Τρεβίζου, το γνωρίζουν όλοι. Αυτό για να σας δώσω μια εικόνα για το που βρισκόμαστε. Η περιοχή του Βένετο για τις άμεσες πληρωμές η υπηρεσία μας ε, ε, ασχολείται με την περιοχή του Βένετο και έχουμε περιφερειακή δραστηριότητα. Είμαστε ε, δημοσίου δικαίου, έχουμε λογιστικές αρμοδιότητες, ε, αρμοδιότητες διαχείρισης της περιοχής και το καθεξής. Και επίσης ε, ελεγχόμαστε και από την ε, Περιφερειακή Αρχή βάση και των αρχών αυτονομίας. Ο οργανισμός ξεκίνησε τις εργασίες του το 2002 και ταυτόχρονα έλαβε και την πρώτη αναγνώριση ως οργανισμός πληρωμών από το Υπουργείο Γεωργικής Πολιτικής. Το 2011 ο οργανισμός πήρε και τις ε, πρώην επιθεωρήσεις γεωργίας και επομένω είναι το σημείο αναφοράς σε περιφερειακό επίπεδο για τις δημόσιες υπηρεσίες ε, που είναι αφιερωμένες στο γεωργικό κόσμο. Ουσιαστικά, οτιδήποτε αφορά τη διαχείριση και την πρακτική συμβολή γίνεται από το δικό μας τον οργανισμό. Από το 2017 επίσης έχουμε και καθήκοντα ενδιάμεσου οργανισμού, διαμεσολαβητή αν θέλετε, πρόκειται για μια καινοτομία και για μας ως οργανισμό, και διαχειριζόμαστε επίσης και το ε, περιφερειακό ε, επιχειρησιακό πρόγραμμα και ασχολούμαστε επίσης και με ε, όλη την περιοχή, βιοτεχνία, εμπόρια, επιστημονική έρευνα, κοινωνική στέγαση, αστικές μεταφορές κλπ. Πρόκειται λοιπόν για έναν οργανισμό ο οποίος είναι ιδιαίτερα σύνθετος και έχει και πολύ σημαντικές αρμοδιότητες που το έχουν ανατεθεί πολλά άλλα στοιχεία που έχουμε σε θέματα ε, γεωργίας. Έχουμε και όλα τα εινολογικά θέματα που όπως σας είπα στην περιοχή του Βένετο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε και το είδατε επίσης ε, και πρόσφατα με την ε, καταιγίδα που είχαμε πριν από 2,5 χρόνια και την πλημμύρα στην περιοχή της Βενετίας και τις ενδιάμεσες περιοχές και έχουμε να κάνουμε και με την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και για το γεωργικό τομέα, αλλά και για τους άλλους παραγωγικούς τομείς. και έχουμε φυσικά και εξουσιοδότηση για τις ε, περιβόητες ε, ε ποσοστώσεις ή πρώην ποσοστώσεις. Έχουμε περίπου 150 άτομα προσωπικό, έχουμε έδρα σε διάφορες πόλεις, έχουμε έδρα σε 7 πόλεις και έχουμε παρουσία σε όλες τις επαρχίες της περιφερειάς μας έχουμε 112.000 εκμεταλλεύσεις και έναν όγκο άμεσων και έμεσων ενισχύσεων περίπου 800 εκατομμυρίων και θα αυξηθεί ε, αυτό ετησίως. Έχουμε εξαιρετικές επιδόσεις εδώ και χρόνια όσον αφορά τη χρήση του προγράμματος ανάπτυξης της υπαίθρου. Έχουμε περίπου 30.000 ε, επιχειρήσεις οι οποίες ε, μας έχουν εξουσιοδοτήσει τη διαχείριση του εινολογικού τους κλάδου και έχουμε και ε, πολύ μεγάλο αριθμό εκταρίων διαχείρισης. Αυτό για να έχετε μια εικόνα του ποιο είμαστε. Τώρα, η άποψή μας για τη μεταρρύθμιση. Είμαστε διατεθειμένοι να διαχειριστούμε ένα ε, σύστημα το οποίο βασίζεται στις ε, παροχές. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα από ό,τι μας ε, έδωσαν να καταλάβουμε αυτοί που μας παρουσίασαν τις μεταρρυθμίσεις. Από την εμπειρία που έχουμε, ε, το παρόν σύστημα είναι αποτελεσματικό. Έχουμε ένα ποσοστό σφάλματος κάτω από το 3% και έχουμε και ισότιμη μεταχείριση στην ε, Ευρώπη. Ενώ το νέο μοντέλο φαίνεται να είναι μια πολύ σύνθετη πρόκληση, που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν και πολύ σημαντικές προσαρμογές και σε διοικητικό επίπεδο ε, και σε ανθρωπίνους πόρους και ίσως και αύξηση κόστους τουλάχιστον για το αρχικό στάδιο και για τους οργανισμούς πληρωμών και για τους δικαιούχους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, πολύ πιο αυστηρούς κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας και που έχουν και κάποιο κόστος για να μπορέσει κάποιος να το διατηρήσει. Σημαίνει ότι αλλάζουμε και συμπεριφορά που σημαίνει ότι χρειάζεται και χρόνος για να το αντιληφθεί κάποιο είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι δύσκολο να υλοποιηθεί και αρκετά περίπλοκο, κυρίως όσον αφορά την ε, προσαρμογή των μέσων για να το επιτύχουμε. Και ένα ε, σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν είναι μόνο το κατά πόσο θα μπορέσουμε να λάβουμε τις ενισχύσεις, αλλά να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης. Επομένως, κατά την άποψή μας, θα είναι στρατηγική σημασία να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα και νέες τεχνολογίες στους ελέγχους, που θα χρειαστεί και πολύ σημαντικές ε, αρχικές επενδύσεις για να έχουμε ένα σύστημα πληροφορικής για την ε, ανταλλαγή και διαβούλευση των δεδομένων για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τους ελέγχους οι οποίοι θα γίνονται απευθεία στο σύστημα και όχι τόσο επιτόπου. Εδώ και χρόνια εμείς κάνουμε παλήθευση με προηγμένα τεχνολογικά συστήματα και ε, αυτό προσπαθούσα να σας εξηγήσω ότι έχουμε και αρκετά σημαντική ψηφιοποίηση. Ε, όσον αφορά τα περιβαλλοντικά στοιχεία, στην περιοχή του Βένετο έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης το οποίο θα πρέπει να το προσαρμόσουμε βάσει και του νέου μοντέλου τώρα. Ε, πέραν ε, της χρήσης του συστήματος ε, τύπου GIS, που είναι το σύστημα που χρησιμοποιούν σχεδόν όλοι, το Geographical Information System, έχουμε και διάφορα άλλα στοιχεία, για παράδειγμα κινητούς χάρτες και ένα εγχειρίδιο για την ερωσιμότητα, το οποίο μας επιτρέπει να μειώσουμε το χρόνο εκτέλεσης των ελέγχων επιτόπου. Αυτό ε, για να υποστηρίξουμε και τις δραστηριότητες επιτόπου. Υπάρχουν και τάμπλετ και συγκεκριμένες εφαρμογές ε, οι οποίες μας επιτρέπουν να κάνουμε σωστή διαχείριση. Στο μέλλον θα κάνουμε και διαχείριση και των ελέγχων ε, όπως καθορίζονται από το σχέδιο της ανάπτυξης της υπαίθρου. Έχουμε επίση ε, συγκεκριμένε διαδικασίε για τι γεωργικέ εκμεταλλεύσεις ε, και με ε, ε φωτογραφίε, δορυφορικέ φωτογραφίε. Συνήθω τι φωτογραφίε τι κάνει ο ίδιο ο δικαιούχο και εμείς από εκεί και πέρα τι χρησιμοποιούμε και ενημερώνουμε το αρχείο μας και το μητρό μας. Επίσης χρησιμοποιούμε και drone τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μια εσωτερική ομάδα πιλότων ε, που έχουν και κατάλληλες πιστοποιήσεις από την ε, Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και εγώ για παράδειγμα έχω τέτοια άδεια. Ε, η χρήση αυτών των μη επανδρομένων ε, σκαφών είναι πολύ σημαντικό για να λάβουμε κατάλληλες φωτογραφίες για την περιοχή, να κάνουμε κατάλληλους ελέγχους και να δούμε αν υπάρχουν αλλαγές σε χρήση γεών ε, σε περιφερειακό επίπεδο και να επικαιροποιούμε το ολοκληρωμένο σύστημά μας. Από το 2017 χρησιμοποιούμε και ε, πειραματικά το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικος για να δούμε αν έχουμε πρόβλημα στις, σε κάποιες εκμεταλλεύσεις. Από το 2018 και μετά επίσης πειραματιζόμαστε και με τη χρήση δεδομένων από αισθητήρε ραντάρ και πάλι του συστήματος Κοπέρνικος. Εγώ μετά από την ε, καταιγίδα Βάια ε, διορίστηκα ως αρμόδιος για τη διαχείριση της επίγουσας αυτής της κατάστασης. Σε αυτή την περίπτωση ο οργανισμός μας χρησιμοποίησε μία ε, εφαρμογή GIS ε, που λέγεται Skianti και ε, Προσπαθήσαμε να δούμε τις πληγήσεις περιοχές από την καταιγίδα αυτή και ε, από εκεί και πέρα να πάρουμε μία σειρά ε, εδαφικών προ, ε, στοιχείων, φωτογραφίες, πληροφορίες για τους κινδύνους, δασικούς χάρτες και το καθεξής και επομένω μπορούμε να πούμε ότι ήμασταν και προπομπή πολλών θεμάτων που αφορούν την τεχνολογία που παρουσιάζονται στο νέο μοντέλο εφαρμογής της ΚΑΠ. Πολλά από αυτά τα προγράμματα παρουσιάστηκαν από τον οργανισμό μας από το 2015 και μετά και σε μία διάσκεψη που έγινε στη Θεσσαλονίκη το είπαμε στις βέλτιστες πρακτικές με οργανισμούς πληρωμών ε, αρκετών κρατών, χάρη στα προγράμματα τα οποία χρηματοδότησε η Όλαφ. Επίση μπορέσαμε να συμβάλλουμε και σε άλλους οργανισμούς πληρωμών και αναφέρομαι ότι υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερου διαλόγου και υποστήριξης και σε τεχνικό και σε ερευνητικό επίπεδο. Αυτή η ιδιαίτερα προσοχή και η καινοτομία στην ΑΒΕΠΑ είναι γιατί θεωρούμε ότι ε, οι νέες διαδικασίες ε, θα είναι πολύ σημαντικές ε, για τη νέα ΚΑΠ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πλήρως αποδοτικό το σύστημα. Χρειαζόμαστε να έχουμε προσπάθειες και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μπορέσουμε να διαθέτουμε και κατάλληλα εργαλεία ελέγχου. Πέραν από την ε, κατάρτιση των χρηστών, βλέπετε να δούμε και το πόσο σύνθετο είναι το θέμα αυτό. Τα συστήματα, για παράδειγμα, παρατήρησης είναι επίγειας είναι πάρα πολύ ε, περίπλοκα συστήματα, ιδίω όταν κάποιο σκοπεύει να τα χρησιμοποιεί αυτομάτω και όχι όταν τα χρειάζεται. Να πω επίση ότι τα δεδομένα είναι τόσο περίπλοκα ότι είναι, ε, που είναι πολύ δύσκολο να δούμε ποιοι είναι οι κατάλληλοι αλγόριθμοι για να επεξεργαστούμε τι πληροφορίε αυτέ και να τι εφαρμόσουμε σωστά. Ολοκληρώνω λέγοντα ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να απλοποιήσουμε αποτελεσματικά. Μία πιθανότητα θα μπορούσε να είναι να δίνονται ενισχύσεις χωρίς αίτηση, εάν η εκμετάλλευση δεν αλλάζει τα αιτήματά της. Θα μπορούσαμε να αυξήσουμε επίσης το απλοποιημένο κόστος και ένα άλλο στοιχείο είναι να βελτιώσουμε τα συστήματα ελέγχου GIS. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν για να διευκολύνουμε το πέρασμα στην ΚΑΠ και θέλουμε να βολτιώσουμε τι δυνατότητε τη εκμετάλλευση με λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη τεχνολογία, αλλά ο ε, παραγωγός θα πρέπει να είναι ε, και όλες οι διαδικασίες φιλικές προς το χρήστη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να παρακαλέσω τους συζητητές ε, να μιλούν παρακαλώ λίγο πιο αργά. Γιατί ξέρω ότι έχετε πολλές πληροφορίες τι οποίε θέλετε να μας δώσετε, αλλά με παρακαλώ διερμηνήσει να ε, σα ζητήσω να μιλάτε πιο αργά. Να ζητήσω τον... Ε, να δώσω το λόγο στον επόμενο ε, ομιλητή, ο οποίο είναι από τη Βάρδη Βιτεμβέργη. Έχει δυστυχώς λοιπόν την ίδια προφορά όπως και εγώ. Προσπαθεί να τα λέει σε καλά γερμανικά. Έχετε το λόγο. Κύριε Νόρμπερτ, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κυρίε και κύριοι, Αξιότιμε συνάδελφοι, από τις ε, υπηρεσίες ε, πληρωμών. Από τους οργανισμούς πληρωμών. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το γεγονός ότι παίρνω το λόγο για τον τοπικό αυτοοργανισμό πληρωμών της Βάτες Βιτεμβέργης, όπως και οι συναδελφοί μου Έχω να πω ότι σε επίπεδο α, ομοσπονδιακό έχουμε 13 τέτοιου οργανισμούς πληρωμών και υπάρχει κεντρική διαμόρφωση του. Εκτιμούμε το γεγονός ότι θέλετε να ακούσετε σήμερα την απόψή μας λοιπόν και τις δικές μας ε, σκέψεις προκειμένου να ρευθούν υπόψη. Γιατί βάτε Βιτεμβέργη, ο οργανισμός πληρωμών όπως σας είπα είναι μία από του 13 ε, οργανισμούς όπως σας είπα. Ε, έχουμε 60.000 Τέτοιε επιχειρήσει στην ε, Βατεμβέργη, δύο τρίτα εξ αυτών είναι γεωργικέ. Και ε, ε λόγω τη τοπογραφία μα πρέπει να πούμε ότι είναι διαφορετικέ οι απαιτήσει και τα χαρακτηριστικά. Και στην Βατεμβέργη βλέπουμε ότι και σε ομοσπονδιακό επίπεδο στη, στα βόρεια κρατήρια τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι στη Βατεμβέργη ή στην Βαβαρία. Και σε ομοσπονδιακό επίπεδο την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την Πράσινη Εβδομάδα και συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή με τον τρόπο και διαπιστώνουμε λοιπόν ότι τα στοιχεία τα οποία τους απασχολούν είναι αυτά που απασχολούν και εμάς. Και αυτό που ήταν θετικό είναι ότι και η εφαρμογή, η αρμοσιμότητα αυτών που έχουν αποφασιστεί στη νέα ε, αγροτική πολιτική είναι εφικτή. Γιατί χρειάζεται ένα σωστό ε, υλοποιήσιμο σχέδιο. Γιατί μόνο αν είναι υλοποιήσιμα τα σχέδια μπορούν σε τελική ανάλυση να γίνουν αποδεκτά. Και προ αυτή την κατεύθυνση πρέπει να λειτουργήσουν όλοι οι τομεί, όλοι οι παράγοντε. Χρειαζόμαστε λοιπόν καλέ προσεγγίσει. Αυτό το είπαν και οι συνάδελφοι από τι Ιταλικέ περιφέρειε. Είναι αρκετά κοντινέ οι σκέψει και ανησυχίε σα με τι δικέ μα και αυτά που είπαν οι άλλοι συνάδελφοι. Αλλά και αυτό θέλω να το πω εδώ σήμερα, είναι ότι η βασική πρόκληση, οι βασικές πρόκλησει μας προκαλούν και κάποιες ανησυχίες. Έχουμε λοιπόν ένα σημείο το οποίο που συζητιέται έντονα στη Γερμανία, αν λαμβάνονται επαρκώ υπόψη τα τοπικά και περιφερειακά χαρακτηριστικά. Όπω ξέρετε, είμαστε ομοσπονδιακό κράτο και αυτό σημαίνει ότι ο δεύτερο πυλώνα, για παράδειγμα, είναι στα χέρια της, των κρατηδίων και σε ό,τι αφορά την νομοθεσία και την υλοποίηση. Στον πρώτο πυλώνα είναι διαφορετικά τα πράγματα προφανώς και στον πρώτο πυλώνα προφανώς έχουμε την υλοποίηση στα χέρια των κρατηδίων. Αν υπάρχει λοιπόν μια εθνική στρατηγική η οποία εφαρμόζεται και σε περιφερειακό επίπεδο, διαπιστώνουμε ποιε είναι οι δυσκολίε όταν υπάρχει αυτό ο περιφερειακό χαρακτήρα και όλε αυτέ οι διαφορέ οι οποίε στη τελική ανάλυση θα πρέπει να καταλήξουν σε ένα κοινό πρόγραμμα, σε μια κοινή εικόνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μεγάλη πίεση συντονισμού αλλά σε άλλες τομείς μπορούν να είναι πιο έντονες οι περιφερειακές διαφορές. Αυτή η περιφερειοποίηση λοιπόν της εθνικής στρατηγικής δεν είναι κάτι μονομερές και ομοιογενές. Όπως σας είπα, είναι ε, προκαθορισμένο το τοπίο αυτό, ιδιαίτερο στο δεύτερο πυλώνα. Καταλαβαίνουμε τι άχθος συνεπάγεται αυτό για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σε ό,τι αφορά το συντονισμό των κρατηδίων μεταξύ του για τι κοινέ ε, δομέ. Ε, IT, αλλά σε τελική ανάλυση το σύστημα αυτό που προκύπτει θα πρέπει να ταιριάζει, να λειτουργεί από κοινού με το εθνικό σύστημα. Και γι' αυτό λοιπόν απαιτούνται προσπάθειες και όλοι οι παράγοντες πρέπει να έχουν υπόψη τους το πόσο δύσκολο είναι το θέμα και να δείχνουν κατανόηση. Γι' αυτό είναι η Γερμανία το μοναδικό κράτος μέλος που κάνει τέτοιες, προωθ... κάνει ενισχύσεις για δύο έτη. Γιατί αυτό αποτυπώνει τις δυσκολίες μας σε ό,τι αφορά τις σωστές διόδους χορήγησης των πόρων ε, προς τους δικαιούχους και την περιφερειοποίηση, όπως σας ανέφερα. Γι' αυτό λοιπόν, ε, σε ό,τι αφορά την ε, παρακολούθηση, είναι το μοντέλο του μέλλοντος, αλλά θεωρούμε ότι στην παρούσα φάση έχουμε κάποια σημεία κριτικής για αυτό το monitoring. Αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτή η υποχρεωτική παρακολούθηση να μπορέσει να συνδεθεί με το σύστημα διοίκησης και ελέγχου από το οποίο θέλουμε και μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να απομακρυνόμαστε. Γιατί στην τελική ανάλυση αυτό το monitoring θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια της περιφερειακής διαμόρφωσης της χώρας μας. Αυτή η περιφερειακή λοιπόν διαμόρφωση σε ό,τι αφορά το monitoring, την παρακολούθηση, σημαίνει ότι ένα σύστημα παρακολούθηση τέτοιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων περιφερειών. κοιτώντα, για παράδειγμα, βλέπουμε στο Μαρεναδρυμό τις ε, δορυφορικές εικόνες και εκεί διαπιστώνουμε τις πρώτες δυσκολίες. Ε, δεν είναι όλα τα ίδια όπως για παράδειγμα στις Άλπες, στη Βαβαρία. Εκεί που χρειαζόμαστε λοιπόν ε, παρακολούθηση να είναι και εφικτό και χρήσιμο το αποτέλεσμα. Ωστόσο, θεωρούμε κάποια στοιχεία δεν έχουν ακόμα ε, αποκρισταλωθεί όπω θα έπρεπε και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου εκ των υστέρων σε ό,τι αφορά τον έλεγχο κυρίω ε, των όρων των οικολογικών ε, προγραμμάτων. Γι' αυτό λοιπόν ζητήσαμε ω τώρα το εξή. Λέγαμε ναι στο monitoring, στην παρακολούθηση, αλλά σε θελούσια βάση, ως μία μόνο δυνατότητα ελέγχου σε ό,τι αφορά τα συστήματα, τα διοικητικά και τα συστήματα ελέγχου του μέλλοντος. Η διενέργεια ενός ελέγχου compliance to performance, η μόρφωση ε, απόδοσης. Είναι κάτι το οποίο ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές, είπαν πόσο σημαντικά είναι τα στοιχεία και πόσο θετικά είναι πολλά στοιχεία που περιλαμβάνονται, αλλά για μας ως ε, οργανισμός πληρωμών αυτό έχει και κάποιες συνέπειες και θα ήθελα πραγματικά να σας τις επισημάνω σήμερα. Έχουμε την υποχρέωση να παρουσιάσουμε αποτελέσματα και επιδόσεις στο μέλλον. Τα αποτελέσματα που πρέπει να πετύχουμε λοιπόν, γιατί αυτά είναι που θα καθορίσουν την επιτυχία της αγροτικής πολιτικής. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι και εδώ, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση, τα, οι έλεγχοι αποτελεσμάτων θα πρέπει να εντετηθούν στις περιφερειακές εργασίες μας. Στη συνέχεια έχουμε και σε σχέση με τη βασική νομική ε, βάση κάποιες νομικές ε, προδιαγραφές για τον ε, πώς θα πρέπει να διαμορφώνονται οι έλεγχοι στα, κρατη, στα κρατηδία. Και σε ό,τι αφορά αυτή την απλοποίηση την οποία διακηρύσουμε για τα προγράμματα υλοποίηση στα κρατήδια, πρέπει να σας πούμε ότι είμαστε αρκετά διστακτικοί, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μπορούν να γίνουν διάφορες προσαρμογές και έχουμε και διάφορες εθνικές διατάξεις οι οποίες ε, προφανώς μας είναι εξίσου γνωστές όπως και οι ευρωπαϊκές ε, διατάξεις. Αλλά, αλλά σε επίπεδο ελέγχου θέλουμε να διατηρήσουμε αυτά ε, που είχαμε ως τώρα. Να διατηρήσουμε λοιπόν το επίπεδο ελέγχου το οποίο να είναι σωστό σε εθνικό επίπεδο και να μην υπάρχει ε, ανταγωνισμός για την πιο ε, μεγάλη ε, απλοποίηση και αυτό να αποβεί προς εις βάρος του σωστού ελέγχου. Θα πρέπει στη τελική ανάλυση δηλαδή να υπάρξει μια συσσόρευση των συστημάτων που θα επιτρέπει τον σωστό έλεγχο των διατάξεων ελέγχου. Να υπάρχει ένα σωστό επίπεδο δηλαδή ελέγχου και τελικά να είναι σωστό το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά σημαντικό και θα μας επιβάρυνε ιδιαίτερα κάτι τέτοιο στην υλοποίηση. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν και συστήματα τα οποία ανταποκρίνονται και στους πόρους. Γι' αυτό λοιπόν εδώ θα θέλουμε να παίξουμε για μια άλλη φορά το χαρτί της επικουρικότητας για την τελική ανάλυση. Ε, δεν θα θέλαμε να έχουμε ένα τεράστιο γραφειοκρατικό άκθος στη Μιτεμβέρκη για ένα ε, μικρό, πραγματικά μικρό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι ε, εδώ θα πρέπει να υπάρχει το επίπεδο ποιότητα και θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε πραγματικά η επικουρικότητα, πώ μπορεί να διαμορφωθεί με σωστό τρόπο και πώ θα λεφθεί πιο πολύ υπόψη. τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω το θέμα ε, των μοναδιών ε, ποσών. Ξέρουμε ότι αυτό ως σημείο αναφοράς είναι σημαντικό. Αυτό να γνωρίζετε. Και ομολογώ ότι το θέμα των, ποσών, των μοναδιών ποσών για μας ως οργανισμός πληρωμών είναι κάτι το οποίο το κατανοούμε. Και φυσικά τα θέματα περιεχομένου θα πρέπει να τα εξετάσουμε. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, έτσι όπως ορίζεται η μοναδία ποσό, θεωρώ ότι υπάρχει υπερβολικά μεγάλο άγχος για μια ομοσπονδιακή δομή όπως η δική μας. Μιλήσαμε για την περιφερειακή διάσταση. Ε, θα πρέπει να λεφθεί υπόψη σε ό,τι αφορά ε, τα μοναδιάποσα θα πρέπει να λεφθεί υπόψη και θα πρέπει να υπάρχει σύγκριση ανάλογα με τις θέσεις, ε, τις δομές των πληρωμών και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη λοιπόν όλες οι παράμετροι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θεωρούμε ότι είναι τεράστιο το άχθος αν μείνουν τα πράγματα ως έχουν σε ό,τι αφορά τα άνατοτα ποσά ή τα μέσα ποσά, μοναδιά ποσά. Εδώ θα κλείσω. Όπως σας είπα, τα μοναδιά ποσά θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τελικά να ανατρέψουν ε, την περιφερειακή αυτή διάθεση, η οποία συμπεριλαμβάνεται και στο εθνικό πρόγραμμα στρατηγικής. Αυτό δεν θα ωφελούσε, θεωρώ, την περιφερειακή διάσταση. Θα κλείσω στο σημείο αυτό. Σας ευχαριστώ και ελπίζω ότι σας παρουσίασα τα θέματα τα οποία ε, μας απασχολούν, τα οποία θεωρούμε ότι αποτελούν προκλήσεις και προφανώ προσβλέπω στην συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ακούσουμε τους εισηγητέ. Ο Πάλο Ντεκάστρο είχε ζητήσει το λόγο, όμω να πάρει πρώτο ε, το λόγο. Να του δώσω το λόγο για Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη. Πρέπει να πάρω το αεροπλάνο και δεν θα μπορέσω να κάτσω για να ακούσω τι απαντήσει. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω όλου του ομιλητέ, κυρίω την τελευταία αναφορά. Ε, το θέμα αυτής της ε, πρώτης μεταρρύθμισης, ε, αυτό το οποίο όπως ξέρετε εξετάζουμε, το συζητάμε, προτείνουμε κάποιε αλλαγέ σε όλε αυτέ τι νομοθετικέ πράξει. και με το να υπάρχει ένας ενιαίος οργανισμός πληρωμών, ε, αυτό ε, κατ' ουσίαν αποκόπτει τις σχέσεις με τις Βρυξέλλες. Γι' αυτό ε, το σκεπτόμαστε, εγώ είμαι λιγάκι αρνητικός, αυτό το θέμα της επανεθνικοποίησης που κατά κάποιον τρόπο συμπίπτει με συγκεντρωτικοποίηση. Γιατί από τη μια δίνει κανείς την αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη, από την άλλη όμως μέσα στα ίδια τα κράτη-μέλη αφαιρούνται αρμοδιότητες από τις περιφέρειες και μεταφέρονται σε κεντρικό επίπεδο. Άρα αυτό είναι αυτό που αφορά τον νέο οργανισμό πληρωμών. Ένα ερώτημα. Αν προχωρήσει αυτό το σχέδιο, τότε όλη αυτή η δουλειά που έχετε κάνει, ε, σε τελική ανάλυση τι θα γίνει με αυτή τη δουλειά τι νόημα θα έχει να υπάρχουν περιφερειακοί οργανισμοί πληρωμών, εάν τελικά υπάρχει ένα ενιαίο και οι αποφάσει ε, λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο. Ακόμα και αν υπάρχει κάποια σχέση με τα κρατήδια ή με τι ε, περιοχέ, αυτή είναι η ερώτησή μου. Ε, εάν τελικά προχωρήσει η κατάσταση ω και και τι θα γίνει με αυτό την κατάσταση που υπάρχει τώρα με τα κέντρα πληρωμών. Ζητώ συγγνώμη που θα αναγκαστώ να φύγω. Ο κύριος Απέτα Γιά Σαπέτα για δύο λεπτά. Επειδή είναι μόνο ε, δύο λεπτά, ε, ξεκινάω με την αξιολόγηση ε, και τα συμπεράσματα. Κοιτάξτε, σήμερα βρισκόμαστε σε μία κέρια στιγμή της ε, Γεωργίας. Το κατά πόσον θα είναι καλή ή κακή η μεταρρύθμιση, το πρόσωπο της Γεωργίας είναι οι οργανισμοί πληρωμών. Εάν δηλαδή πετύχει μεταρρύθμιση, πρέπει εκείνοι να πετύχουν. Ε, μπορούμε να φτιάξουμε τις επικεφαλίδες, αλλά αν δεν ισχύει η βάση, τίποτα δεν θα έχουμε καταφέρει. Ε, αυτή τη στιγμή ε, αυτό που θα κάνουμε είναι να διαμορφώσουμε το κείμενο και αν τα καταφέρουμε θα είμαστε και ευγνώμονες ως ευρωβουλευτές. Υπάρχει το θέμα της περιφερειοποίησης. Από, όλους τους, ε, από όλες τις πολιτικές ομάδες λένε ότι ναι το θέλουμε αρκεί το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που όλοι οι οργανισμοί πλωμών είπαν ότι βλέπουμε ε, σε αυτό το κοινό μοντέλο να υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες. Ε, παρ' όλα αυτά όμω, είναι σημαντικό να διεκδικήσουμε την απλούστευση. Η ε, απόδοση από την κατάρριξη γραφειοκρατίας πρέπει να φτάσει στους γεωργού και γι' αυτό είπαμε όλοι να προβλέψουμε μία μεταβατική περίοδο. Τώρα αν θα είναι ένα ή δύο χρόνια, αλλά να έχετε την ευκαιρία ευκαιρία να ε, προσαρμόσετε το σύστημα. Ακριβώς όπως κάθεστε εδώ, ε, θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων. Επιθυμούμε όλοι οι γεωργοί να έχουν το απλούστερο μη γραφειοκρατικό σύστημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ε, ε, η Ιταλία τα καταφέρνει καλά, η Γερμανία, η Πορτογαλία. Αυτό είναι θαυμάσιο. Χρειαζόμαστε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Και είπατε ότι χρειαζόμαστε ανεκτικότητα, ε, να διαχωρίζουμε ανάμεσα σε λάθη και κακή διαχείριση. Α πούμε, έχω μια περίπτωση όπου ένα γεωργό ανέφερε τρία εκτάρια λιγότερα και τιμωρείται. Αυτό δεν το κατανοεί. Αυτό ήταν απλά ένα παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμάς, Συνάδελφο Μίλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας ε, για όλα αυτά που μας ε, είπατε. Δεν θέλω ε, να επαναλάβω αυτά που είπε ο συνάδελφος, αλλά θέλω να σας πω ότι δουλεύουμε πάνω σε μία θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Πιστεύουμε μέχρι τα, μέση του, μέχρι τα μέσα του έτους ε, να έχουμε επεξεργαστεί μια θέση και να ξεκινήσει ο τριμερής ε, διάλογος. Είχαμε μια συνεδρία των συντονιστών. Έχουμε τώρα συμπεριλάβει όλες τις απόψεις και ε, πολύ συγκεκριμένα έχουμε να σας υποβάλουμε ερωτήσεις. Για μας λοιπόν η ανταλλαγή απόψεων είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί έχουμε συγκεκριμένα άρθρα 14, 15, το 87 και άλλα συναφή άρθρα που που είναι ε, καθοριστική σημασία. Ίσως μπορούμε να τα πούμε και σε γραπτή μορφή με περισσότερες λεπτομέρειες. Για μένα λοιπόν είναι σημαντικό να μας πείτε ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες των οργανισμών πληρωμών. Πραγματικά χρειαζόσαστε μεγαλύτερη ευελιξία ε, όσον αφορά τους στόχους ε, και τους δείκτες των στόχων και την απόδοση και πιστεύετε ότι οι οργανισμοί πληρωμών πράγματι είναι πρόθυμοι να δουλέψουν με το μοντέλο της απόδοσης, γιατί μιλάμε για μια μεταβατική περίοδο δύο ετών. Και κατά την άποψή σας, ε, πόσο απαραίτητο είναι να υπάρχουν υποδομές και πόροι. Γιατί τώρα έχουμε το προσωπικό, αλλά διερωτώμε κατά πόσον αρκούν όλα αυτά, γιατί αν πρέπει και να κάνετε τη μέτρηση και την αξιολόγηση, νομίζω ότι θα είναι πιο πολύπλοκη η κατάσταση. Πιστεύετε ότι ο στόχος ε, της απλούστευσης, ε, ο στόχος αυτός ε, μπορεί να επιτευχθεί με αυτό το μοντέλο. Σε γενικές γραμμές αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλοι μας δεχόμαστε ότι επιθυμούμε να περάσουμε από τη συμμόρφωση στην απόδοση. Γνωρίζουμε ότι ε, πρέπει ε, να προστατεύσουμε το κλίμα και το περιβάλλον, αλλά ο δρόμος προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ακόμα ακανθώδης. Πολύ ωραία. Ε, περνάμε τώρα στις πρώτες απαντήσεις των τεσσάρων ε, οργανισμών πληρωμών και μετά ε, θα τεθούν και άλλες ερωτήσεις. Θα λοιπόν να ε, ξεκινήσω με τον κύριο Νοβακόφσκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάω με το τρίτο ερώτημα, διότι νομίζω ότι το ερώτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο θέματα που είναι πολύ σημαντικά σε σχέση με το νέο πρόγραμμα. Πρώτον, οι νομοθετικές ε, διατάξεις ε, και μετά η ψηφιοποίηση. Αυτοί είναι οι τομείς οι οποίοι θα είναι οι ε, πιο σημαντικοί όσον αφορά τα αποτελέσματα. Για μας αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε σωστό ορισμό, να έχουμε μετρήσεις έτσι ώστε να μπορούμε όλα αυτά να να τα χρησιμοποιήσουμε στο σύστημα της, ε, ε, στο ψηφιοποιημένο σύστημα και μετά να μπορούμε να καταρτίζουμε τις ε, εκθέσεις. Όσον αφορά τις ανάγκες προσωπικού, μέχρι τώρα δεν κάναμε αξιολόγηση, άρα δηλαδή δεν λέμε ακόμα κατά πόσο χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό. Έχουμε την εντύπωση ότι το προσωπικό που έχουμε αρκεί έτσι ώστε να προετοιμάσουμε τη νέα προοπτική και γι' αυτό ακριβώς προετοιμαζόμαστε. Και πάω τώρα σε μία από τις ε, προηγούμενες ερωτήσεις. Ε, υποστηρίζουμε πλήρως ε, την προσέγγιση της περιφερειοποίησης που είναι πολύ σημαντική για μας. Αυτό που έχει σημασία είναι να λαμβάνουμε καλύτερα υπόψη μας τα δεδομένα των περιφερειών. Και εδώ είναι σημαντική η αιρεσιμότητα. Ε, στις μικρές επιχειρήσεις κάτω από 10 εκτάρια σε εμά ισχύει το εξή. Υπάρχει ο κίνδυνος, ε, ε, μερικοί να μην μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις. Στον τομέα αυτό θέλουμε να ξεφύγουμε από την αιρεσιμότητα. 1.300.000 δικαιούχοι στα στατιστικά δομένα βλέπουμε ότι 600.000 επιχειρήσεις είναι κάτω από 10 εκτάρια. Εδώ λοιπόν η εισαγωγή της ε, αιρεσιμότητας ε, για μας ε, θα σήμαινε αύξηση των δαπανών και επίσης και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για τον προγραμματισμό. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικότερα ερωτήματα όσον αφορά το νέο σχεδιασμό και όσον αφορά στη μεταβατική περίοδο εμείς θα θέλαμε να προτείνουμε δύο χρόνια ή δυνατόν ο κύριος Ριμπέρο. Θα ξεκινήσω με τα πιο απλά ερωτήματα. Είναι σαφές για μας ότι καλύτερα για μεταβατική περίοδο να έχουμε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γιατί αυτό ε, θα μας διευκολύνει στην τεχνολογική, τεχνολογική προσαρμογή. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες ε, που ακόμα υπολείπονται. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω. Θα ήθελα όμως επίσης να πω ότι θα υπάρξει βεβαίως τεχνολογική προσαρμογή αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν και δύο άλλα θέματα που είναι πολύ σημαντικά ε, εμάς, εμείς ε, θέλουμε να μην υπάρχει επικάλυψη των δύο μοντέλων. της ε, απόδοσης με τη συμμόρφωση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτά τα δύο ε, να συμπίπτουν. Και υπάρχει και το θέμα της απλούστευσης. Όσον αφορά την cross-compliance για τους μικρούς οδηγούς, τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να έχετε έτσι μια ιδέα, στην Πορτογαλία και με βάση την αξιολόγηση που έχουμε θα είχαμε αύξηση κατά 50% των ελέγχων για να γίνεται ο πλήρης ελέγχος που χρειαζόμαστε όλων των ε, γεωργών και όλων των συστημάτων. Αυτό είναι τεράστια αύξηση. Κατά... Μέσα από μια ιστορική διαδρομή έχουμε μια cross-compliance που οδηγεί στο έχουμε περίπου 160 ευρώ Άρα δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσον θα είχε νόημα να έχουμε αυτό το διοικητικό βάρος, όλο αυτό το διοικητικό βάρος για άλλα 160 ευρώ. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια βασική πτυχή. Ε, πρέπει να υπάρχει η απλούστευση στη διαδικασία ελέγχου. Κυρίως ε, στις μικρές επιχειρήσεις. Όσον αφορά την περιφερειοποίηση, ε, δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα για μια χώρα όπως είναι η Πορτογαλία. Ε, υπάρχουν άλλες χώρες όπου αυτό είναι ένα θέμα, αλλά σε εμά δεν είναι τόσο σημαντικό το θέμα. Η Πορτογαλία έχει τρεις αυτόνομες ε, περιοχές με κυβερνήσεις και κοινοβούλια, αλλά έχουμε μία αρχή πληρωμών. Άρα δηλαδή το θέμα δεν είναι τόσο σημαντικό κατά την εμπειρία μας αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά ίσως να είναι κάπου αλλού. Ε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, ε, κυρίως ε, τους βουλευτές για τις ερωτήσεις και για το επικριτικό πνεύμα με το οποίο συμφωνώ. Ως οργανισμός πληρωμής, κυρίως από αυτά που ακούσαμε και από το συνάδελφο από τη Γερμανία. Και εμείς, παρά το γεγονό ότι είμαστε ένας πολύ εξελιγμένος ε, και σημαντικός οργανισμός πληρωμών με προηγμένες τεχνολογίες, θεωρούμε ότι το πέρασμα ε, σε αυτά τα δύο διαφορετικά μοντέλα, σε αυτή την αλλαγή νοοτροπίας που θέλω να πω ότι είναι και πολιτιστική αλλαγή, θα έχει σίγουρα κάποιο κόστος. Κόστος ε, και όσον αφορά τον ε, οργανισμό πληρωμής, αλλά και όσον αφορά και τα καθήκοντα ε, για τους γεωργούς και φυσικά θα αυξηθεί και το κόστος. Και μας μας ανησυχεί αυτό και μας ανησυχεί και αυτό που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Δεκάστρο και το ανέφεραν και οι συνάδελφοι, το γεγονός ότι δεν υπάρχει άμεση επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η άμεση σχέση. Αυτό ε, μας απέφερε πολλούς καρπούς, μας έκανε ε, πιο προηγμένος και μας προσέφερε και τη δυνατότητα να είμαστε πιο προηγμένοι. Εμείς ε, αδράξαμε αυτή την ευκαιρία η οποία προσφέρεται σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε δομή που έχει οργανισμό πληρωμής. Ακόμα και αν εμείς ήμασταν διατεθειμένοι πλήρως και έτοιμοι ε, για αυτή την ε, αλλαγή, δεν είμαι βέβαιος ότι είναι έτοιμοι και οι γεωργοί. Εγώ μάλλον είμαι πιο επικριτικό, πιστεύω ότι οι Γεωργοί δεν είναι έτοιμοι να αντιληφθούν γιατί συμβαίνουν τα πράγματα ε, έτσι και γιατί μέχρι σήμερα, μιλά πάντα για τη δική μα την περιοχή, που το σύστημα απέφερε καρπούς, ε, γιατί να πρέπει να αλλάξει τώρα εκ βάθρων. Και γνωρίζουμε ότι όταν υπάρχει μια αλλαγή, ακόμα και αν η αλλαγή αυτή είναι θετική, υπάρχει πάντα ένα κενό. Ξεκινάμε πάντα από πιο χαμηλά. Και δεν ξέρω και αν ε, η Ιταλική χώρα τα αντιλαμβάνεται αυτά, δεν είναι τις αρμοδιότητές μου και έχει ζητήσει αυτά τα δύο χρόνια ε, αναμονής ή αν θέλετε ε, τα μεταβατικά, τα οποία θα μας ε, είναι και ιδιαίτερα σημαντική. Κα, ευχαριστώ πολύ. Ja, ich kann mich, oh, Και εγώ συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Ε, ε, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα του κ. Ντικάστρο, ε, πράγματι το θέμα της περιφερειακής διαμόρφωσης και ε, διαχείρισης είναι πολύ σημαντικό σε ένα ομόσπονδο κράτος. Και εμείς πιστεύουμε ότι όσον αφορά τα κίνητρα που πρέπει να υπάρχουν εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να έχουμε κατά νου το τι ακριβώς προσφέρουν οι οργανισμοί πληρωμών στο σύστημα και αυτό να ενισχυθεί. Εγώ ε, θέλω να σας πω το εξής. Η προσέγγιση για την απόδοση είναι καλή. Γιατί νομίζω με αυτή μπορούμε να επιτύχουμε πάρα πολλά. Και πράγματι όσον αφορά τις ε, αλλαγές θα πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα. Αυτό που επίσης είναι σαφές είναι ότι στο νέο σχέδιο κανονισμού σε τελική ανάλυση αναφέρεται ότι θα πρέπει να έχουμε ένα εύρυθμα λειτουργούν σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Ε, σε τελική ανάλυση ε, θα πρέπει να δούμε λιγάκι και το θέμα της ποιότητας και αυτό που ενδιαφέρει είναι ε, κατά πόσον μπορούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Στην κίτρινη κάρτα εκεί το είδα ε, για να το κάνουμε θα χρειαζόμασταν 1,7 δις ευρώ και η αξία που θα προέκυπτε από τις κυρώσεις είναι 7.500 ευρώ. Άρα δηλαδή δεν αξίζει τον κόπο. Και αυτά είναι τα θέματα όπου σας λέω ότι το εθνικό σύστημα παίζει ρόλο. Τέτοιου είδου θέματα θέλουμε να εξετάσουμε. Όπω σα λέω, η περιφερειοποίηση στο πλαίσιο της, ε, του στρατηγικού σχεδιασμού είναι σημαντική. Ε, νομίζω ότι μπορούμε κάπως να τα καταφέρουμε. Παρ' όλα αυτά, το μοντέλο της απόδοσης, νομίζω το θίξατε κυρία Μούλερ, ε, πράγματι ο στόχος είναι σωστός και θέλουμε να το στηρίξουμε. Όσον αφορά σημαντικά θέματα, το είπε και ο συνάδελφος, υπάρχουν διάφορα θέματα, ε, κυρίως όσον αφορά στις ε, μικρές επιχειρήσεις για τη δέσμευση του άνθρακα, παραδείγματος χάρη, νομίζω ότι εκεί μπορούμε και στον νέο Γεωργό να, δώσουμε, να καταλάβει ότι θέλουμε νέα κίνητρα με την κοινή πολιτική, κοινή, κοινή πολιτική γεωργίας. Αυτό είναι κάτι που σκεφτόμαστε μεταξύ άλλων. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ. Και να περάσουμε στον επόμενο γύρο ερωτήσεων, τις οποίες θα μπορέσουμε να συνοψίσουμε από ένα λεπτό ο καθένας, ε, ο, η συνάδελφος η κυρία Σάντερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους σας για τις παρουσιάσεις σας. Και νομίζω ότι το διακύβευμα είναι πραγματικά μεγάλο στο κείμενο αυτό. Θα ήθελα να επιμείνω σε δύο στοιχεία. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την απλοποίηση. Εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις με αυτά που θα αποφασίσουμε. Έχουμε ήδη δώσει κάποια στοιχεία των απαντήσεων σήμερα. Ακούγοντας αυτά που λέτε, δεν είμαι καθόλου βέβαιη ότι μία απλοποίηση τελικά θα αλλάξει κάτι ουσιαστικό για τους γεωργούς μας, ε, οι οποίοι ήδη δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό με τους ελέγχους και την πληθώρα κανόνων. Δεύτερο στοιχείο, το οποίο ακούσαμε και είναι πολύ σημαντικό, είναι ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας ο οποίος θα πρέπει να διατηρηθεί στο μοντέλο και αυτό δημιουργεί ένα έντονο αν θέλετε, ένα, ένα έντονο σύνδεσμο μεταξύ ευρωπαϊκού, εθνικού, περιφερειακού επίπεδου μπορεί να επιτευχθεί με το σεβασμό των ευρωπαϊκών κανόνων. Και προφανώς συνεπάγεται και έναν έλεγχο των ευρωπαϊκών αυτών ε, διατάξεων. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το θέμα της συμμόρφωσης με απασχολεί, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας ε, με μεγαλύτερη ακρίβεια εδώ. Θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσον το θέμα της ενεμοποίηση των εσόδων ε, σα ικανοποιεί και να ξεφύγουμε από την απόδοση. Όχι πως θα την αφήσουμε εντελώ κατά μέρος την απόδοση. Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά που ζητούν οι πολίτες, αλλά σε μια πιο απλή μορφή. Και οι εθνικές αρχές ε, οργανισμοί πληρωμών, σε τι πιστεύουν σε ό,τι αφορά τη διατήρηση των ε, κανόνων συμμόρφωση, Υπάρχει όφελο, ή πιστεύετε ότι υπάρχει μια χαλάρωση στην κατεύθυνση αυτή. Και να πω ότι μου προκάλεσε ε, έκπληξη αυτή η διαφάνεια του εκπροσώπου της Πορτογαλίας, η οποία ξεκάθαρα δηλώνει ότι θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχουν έλεγχοι συμμόρφωση σε εθνικό επίπεδο. Το λέει ξεκάθαρα. Μα ποιος θα τους κάνει λοιπόν αυτούς τους έλεγχους συμμόρφωσης αν όχι αυτή που προβλέπετε. Ευχαριστώ. Έχετε λίγο χρόνο παραπάνω γιατί είμαστε και πιο λίγοι. Ε, κύριε Ντόρφμαν, ευχαριστώ πολύ και για την γενναία δωρεά. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι έχουμε απέναντι μας τους υπεύθυνους οι οποίοι θα κληθούν να τα υλοποιήσουν όλα αυτά που θα αποφασίσουμε. Είναι όλο ένα και πιο περίπλοκο το θέμα όταν συζητάμε υπηρεσίες πληρωμές. Απ' τη μια υπάρχει ε, ένας οργανισμός ο οποίος εξυπηρετεί κάποιες περιοχές ε, ε, και υπάρχει μια περιφέρεια όπως η δική σας, ε, η οποία ίσως υποθέτω ότι είναι και πιο μεγάλη, έχει περιφερειακό σύστημα. Εξετάζοντας εκ τα δύο συστήματα, υπάρχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα κατά την άποψή σας και επίση αυτό το νέο μοντέλο το οποίο ετοιμάζουμε εμείς εδώ, το οποίο είναι όλο ένα και πιο επικεντρωμένο σε εθνικό επίπεδο, εθνικά στρατηγικά σχέδια, θα μπορούσε ίσως να δημιουργήσει πιέσεις για τους ε, περιφερειακούς οργανισμούς πληρωμών. Διότι θα μπορούσε να υπάρξει και μία όθηση προς ε, μία εθνική υπηρεσία ή κατά την άποψή σας αυτό το ευηρετικό σύστημα της Ιταλίας θα μείνει έχει. Ευχαριστώ κύριε Φλάνακαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία ερώτηση που έχω να κάνω προς όλους τους ομιλητές. Ελπίζω να μπορέσετε να την απαντήσετε. Πιστεύετε ότι το μονοπάτι που έχουμε επιλέξει θα μας δώσει την ε, επιθυμητή ευκταία απλοποίηση, γιατί αυτό το επαναλάμβανε ο Επιτροπός διαρκώς, το είπε χιλιάδες φορές πώς θα είναι το σύστημα αυτό πιο απλό τελικά. Δεν ξέρω αν θα είναι πιο απλό, αν θα λειτουργήσει καλύτερα, αλλά θεωρώ ότι η απλοποίηση επί του παρόντος είναι θα μένει 50 ε, μέτρα κάτω στο χώμα. Ο Πολωνός εκπρόσωπος ε, ανέφερε ότι υπάρχουν 11.000 υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται για τη μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική. Αναρωτιέμαι λοιπόν για πιο μικρέ χώρε όπω η Ιρλανδία, Φερρυπίν. Το Υπουργείο Γεωργία ε, έχει σε όλη την Ιρλανδία 3.000 υπαλλήλου όλου και όλου. Προφανώ η Πολωνία έχει πιο, πολλές, ε, πιο μεγάλες εκτάσεις να καλύψει. Θα πρέπει να συνενωθούν πολιτικές όμως μαζικά και αυτό θα ε, περιορίσει τους ανθρώπινους πόρους από όλες τις χώρες. Πιστεύετε ότι πιο μικρές χώρες θα χρειάζονταν πιο πολύ υποστήριξη, γιατί αν έχετε 11.000 άτομα που εργάζονται μόνο στον τομέα της μεταρρύθμισης και εμείς έχουμε 3.000 σε όλο το Υπουργείο Γεωργίας, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Ο Ιταλός επίσης εκπρόσωπος είπε ότι θα κοστίσει πιο πολύ η υλοποίηση των ε, περιβαλλοντικών μέτρων. Πόσο παραπάνω θεωρείτε, ποσοστία, πόσο παραπάνω θα κοστίσει σε σχέση με το τρέχον κόστο και από πού θα έρθουν αυτά τα κονδύλια. Ευχαριστώ πολύ. Ρούσα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και χαίρομαι ιδιαίτερω που γίνεται αυτή η ανταλλαγή απόψεων με του οργανισμού πληρωμών. Γιατί εδώ πέρα στι Βρυξέλλε καταρτίζουμε ε, κανόνε, αλλά στην τελική ανάλυση εσεί τα κληθείτε να τα αντιμετωπίσετε αυτά στην καθημερινή σα δουλειά. Και είναι καλό λοιπόν που σε αυτή τη φάση ήδη συζητάμε την ε, εφαρμοσιμότητα, την υλοποίηση των κανόνων αυτών, κατά πόσο μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε. Ανησυχώ σε ό,τι αφορά το κόστος υλοποίησης, όπως και άλλοι μιλητές. Αυτό το κόστος υλοποίησης και ελέγχου πόσο θα είναι. Και κοιτώντα στο δεύτερο πυλώνα βλέπουμε υψηλά ποσοστά και για την υλοποίηση και για τον έλεγχο Όσο πιο πολλέ προδιαγραφέ θέτουμε προφανώ, τόσο πιο πολύ έλεγχο θα χρειαστεί και τόσο πιο πολύ πιο υψηλά θα είναι τα, το κόστος ε, ελέγχου. Σε ό,τι αφορά τους επιτόπου ελέγχου τώρα, φυσικά είναι και επίπονοι και για τους ελεγκτές και για τους ε, γεωργούς και προφανώς πολύ βόρεια διαδικασία. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να τους περιορίσουμε στο βαθμό το δυνατό τους ελέγχους επιτόπου. Όπως είπαν και κάποιοι μιλητές, ε, θεωρώ ότι οι νέες τεχνολογίες, ε, η έλεγχη μέσω δορυφόρου για παράδειγμα, θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα λύση. Θα πρέπει λοιπόν ε, σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές μας να λάβουμε υπόψη ακριβώς και αυτό το σκέλος της εφαρμοσιμότητας και κυρίως να μην καταλήξουμε να έχουμε διατάξει τις οποίες θα, θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητε ε, ελέγχου, για παράδειγμα, μέσα στον δορυφόρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, τον κύριο Στέλλα θα ήθελα να ρωτήσω. Εσείς αναφερθήκατε σε ένα πολύ ε, καλό παράδειγμα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς πιστεύετε, των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, συγγνώμη, πιστεύετε ότι αυτό το μοντέλο θα πρέπει να επαναληφθεί και σε άλλες περιφέρειες. Ε, το λέω και εν ώψη και πολύ σοβαρών ε, περιστατικών απάτης για ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία προέκυψαν προσφάτως στη Σικελία αλλά και σε άλλες περιοχές. Επίσης, επειδή στην Ιταλία ε, απορρεφώνται με λιγότερη αποτελεσματικότητα οι ε, επιδοτήσεις για την αλία. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε ε, σε περιοχές μεγάλης γεωργικής και λευτικής παραγωγής όπως είναι η Σικελία να συσταθεί ένας οργανισμός ο οποίος θα μπορούσε να διαχειριστεί τα κονδύλια όπως κάνετε εσείς στην περιοχή του Βένετο για την Αλία και τη Γεωργία όπως γίνεται τώρα στην Πορτογαλία, για παράδειγμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, ε, συνάδελφος Νάπατσεκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πολύτιμη συνεισφορά σας ε, ε, στην κατεύθυνση του, της πιο απλουστευμένης κοινή γεωρικής πολιτικής. Και εδώ έχω να κάνω δύο ερωτήσεις. Ε, κάτι που ενδεχομένως να έχετε ήδη βιώσει, αυτό που λέμε ενεργός ε, γεωργός, ε, ε, γνήσιος γεωργός. Τώρα παίζουμε με αυτή την ιδέα του πώς θα τον χαρακτηρίσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, στα κριτήρια που εξετάζεται είναι και το θέμα των δειγματοληψιών, αλλά βασικά θα πρέπει να ελεγχθεί όλος ο πληθυσμός, δεν ξέρω, ο κ. Νοβακόφσκι ίσως ε, να έχει κάποια εμπειρία επί του θέματος. Το ίδιο ισχύει και για μια άλλη ιδέα. Συζητάμε εδώ για, τις, τα χαρακτηριστικά των ε, εδαφών του τοπίου. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα κριτήριο επιλεξιμότητας. Θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο στο θέμα της απλούστευσης του κόστους. Συνάδελφος Τολερέ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ εργάζομαι στον τομέα τη γεωργία εδώ και πάρα πολύ καιρό και μου εξηγούν εδώ και καιρό ότι αυτή η μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ θα απλοποιήσει τη ζωή των αγροτών. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη να σα πω την αλήθεια. Αυτή η απλοποίηση που προτείνεται, η οποία φαίνεται ότι σα προκαλεί μεγάλο ενθουσιασμό θα απλοποιήσει όντω την ε, ζωή των κρατών μελών, αλλά και των ε, γεωργών που συμμετέχουν, για παράδειγμα, μέσω τη ψηφιοποίηση. Σε κάποιε περιπτώσει ε, όλα αυτά δεν λειτουργούν. Για παράδειγμα, δεν λειτουργούν τα τηλέφωνα, δεν λειτουργούν οι τεχνολογικέ αυτέ διατάξει. Τι γίνεται λοιπόν με τον γεωργό, ο οποίο καλείται να εφαρμόσει αυτά τα καινούργια στοιχεία, αλλά τίποτα δεν λειτουργεί. Αυτή η μεταρρύθμιση δεν θα πρέπει να προβλέψει και μια περίοδο προσαρμογής. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφο η κυρία Μέτσα. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ε, με ε, το εξής. Ε, υπάρχει ένας μύθος ότι πρέπει να υπάρχει απλούστευση. Εάν λοιπόν θέλουμε περισσότερα δεδομένα και αν θέλουμε να ελέγχουμε περισσότερο την απόδοση, νομίζω ότι δεν είμαστε στη λογική της ε, απλούστευσης και αυτό είναι σωστό, γιατί ακούω ότι χρησιμοποιείτε την ε, τεχνολογική πρόοδο και ότι ανταλλάσσετε απόψεις ε, για να μπορέσετε να βρείτε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν ας μην μιλάμε πια για την απλούστευση, γιατί δεν είναι αυτός ο στόχος. Και από την άλλη, αν κατάλαβα καλά, ε, η βασική περισσότερη δουλειά δεν προέρχεται από τους γεωργούς, αλλά θα αφορά στα, στους οργανισμούς πληρωμών και στα Υπουργεία των κρατών μελών. Θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσον υπάρχει προϋπολογισμός για το θέμα της ε, τεχνολογικής ανταλλαγής, κατά πόσον αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και κατά πόσον η Κομισιόν στηρίζει τα κοινά κέντρα ερευνών. Αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει είχα να επιλέξω πάρα πολλά και το θέμα είναι ότι ε, πώς μπορούμε να δούμε λιγάκι το θέμα της ε, διάβρωσης του εδάφους. Και το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι κάτι το οποίο μας ε, απασχολεί και πρόκειται για το εξή. Μπορείτε εσείς ε, να μετρήσετε τη συγκέντρωση της γης και αν ναι, ε, πώς και αν όχι, τι είναι εκείνο που λείπει. Και από τον κανονισμό για ολοκληρωμένα δεδομένα του 2018, εκεί μπορεί κανείς να δει τον ε, βαθμό της ιδιοκτησία και τι ανήκει σε μητρικέ εταιρείε. Αυτά τα δεδομένα μπορείτε να τα συνδυάσετε με το IEX. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Ε, την πρώτη προς τον ε, κύριο Στέλλα. Ε, στην ομιλία σας μιλήσατε για ένα σημαντικό κίνδυνο που αφορά στην αύξηση του κόστους που θα συνεπάγεται αυτός ο κανονισμός, αύξηση κόστους για τους οργανισμούς πληρωμών αλλά και για τους δικαιούχους. Και αυτό μας ανησυχά πάρα πολύ γιατί έχουμε επιλέξει να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση της απλούστευσης. Ε, πιστεύετε ότι ε, θα έπρεπε να σκεφτούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε την αύξηση του κόστους που θα επιβάλλει περισσότερο τους ε, δικαιούχους. Και όσον αφορά τις απάτες, ε, στην Ιταλία αποκαλύφθηκε ε, μία μεγάλη απάτη, 50 εκατομμύρια ευρώ απάτη, γιατί κάποιοι έλεγαν ότι είχαν μισθώσει εκτάσεις που κατ' ουσίαν όμως δεν είχαν μισθώσει. Αποκαλύφθηκε αυτή η απάτη, ευχαριστούμε αυτούς που την αποκάλυψαν, αλλά αν περάσουμε σε ένα πιο δύσκολο σύστημα ελέγχου, δεν θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί και ο κίνδυνος των απατών, ε, διότι ε, το προηγούμενο σύστημα μας ε, προσέφερε σημαντικές εγγύησεις, είχαν περιοριστεί πολύ τα ασφάλματα και οι λίγες απάτες αποκαλύφθηκαν. Και θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψη και από αυτού του θέματος. Πολύ ωραία. Τέλειωσαν οι ερωτήσεις. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι μετά ε, να τοποθετηθούν ε, οι οργανισμοί πληρωμών. Κυρία Μπόχμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχά να πω από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θεωρούμε ότι η ανταλλαγή αυτή απόψεων είναι εξαιρετικά ωφέλιμη και προφανώ καθημερινά ε, εργαζόμαστε με του οργανισμού πληρωμών και χαρήκαμε που διαπιστώσαμε ότι και οι ίδιοι οργανισμοί πληρωμών ε, ήρθαν να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για το νέο μοντέλο υλοποίησης. Προφανώς ε, ακούμε και εισακούμε αυτά που λένε οι οργανισμοί πληρωμών και αυτό έχει ξεκινήσει και πριν τη σημερινή διαδικασία. Έχουμε αυτό το δίκτυο των οργανισμών πληρωμής ε, και έχουμε εργαστεί ήδη μαζί με τον οργανισμό αυτό, με τους οργανισμούς αυτούς πριν την υποβολή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περιφερειακή και μη περιφερειακή διάσταση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να διατηρηθούν οι οργανισμοί, οι πιστοποιημένοι οργανισμοί πληρωμή και προφανώς να παραμείνουν και σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτή είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λέμε ότι κοιτάξτε έχουμε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί σωστά και σύμφωνα με το ελεκτικό συνέδριο πραγματικά λειτουργεί σωστά το σύστημα. Θέλουμε οι οργανισμοί πληρωμή αυτοί να συνεχίσουν να αποτελούν παράγοντες κλειδί σε αυτή τη μορφή διακυβέρνηση τη ΚΑΠ όταν κινηθούμε προς την υλοποίηση. Και γιατί, γιατί αυτό το σύστημα είναι σε εφαρμογή εδώ και 20 χρόνια και πραγματικά πετυχάνει αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ΚΑΠ. Το νοποιημένο σύστημα λοιπόν διαχείρισης, έχει όλες τις εφαρμογές, όλο το σύστημα πιστοποίησης, όλα αυτά λοιπόν είναι ήδη ρυθμισμένα. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη να δημιουργηθούν νέα συστήματα IT, ενώ τα συστήματα που ήδη έχουμε λειτουργούν σωστά. Όλα αυτά λοιπόν λειτουργούν άψογα και οι γεωργοί χρησιμοποιούν αυτό το νέο σύστημα IT. Έχουμε λοιπόν εδώ την εξή λογική, να διατηρηθεί η δομή διαχείριση η οποία λειτουργεί χωρί να αλλάξει. Α μην γίνουν αλλαγέ εδώ. Οι αλλαγέ, και αυτό το είπαν και οι πανελίστε μα σήμερα, είναι ότι εφ' θα επικεντρωθούμε στο σκέλος της ε, απόδοση. Αυτό θα αποτελέσει απλοποίηση. Πιστεύουμε ναι από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και γιατί. Γιατί δεν θα έχουμε κανόνε οι οποίοι θα ισχύουν παντού σε όλη την Ευρώπη. Ναι, τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να ορίζουν τα κριτήρια ε, νομιμοποίησης και τα στοιχεία του τοπίου, αλλά δεν θα πρέπει να ορίσουμε τι είναι για παράδειγμα φράχτιζα. Εδώ υπάρχουν οι τοπικέ αυτέ και περιφερειακέ ιδιαιτερότητε, οι οποίε θα μπορέσουν να συνεχίσουν να υφίστανται. Εδώ υπάρχει λοιπόν περιθώριο απλοποίηση γιατί αυτό το one side fits all, η μία ενιαία λύση για όλου. σε κάποιε περιπτώσει σήμερα συνεπάγεται ότι οι αγρότε αναγκάζονται να εφαρμόζουν διατάξει που δεν έχουν νόημα για την περιοχή του, αλλά τι να κάνουμε ισχύουν για όλου στην Ευρώπη. Άρα, για να πετύχουμε αυτή την απλοποίηση, θέλουμε να μπορούμε να ε, προσαρμόζουμε την ε, ε, υποστήριξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχουν λοιπόν διαφορές σε περιφερειακά επίπεδα μέσα στα κράτη-μέλη. Να πω και δύο λόγια τώρα για την ψηφιοποίηση και τον εξυγχρονισμό των συστημάτων, γιατί εδώ προφανώς πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να οδηγήσει σε απλοποίηση, να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που υπάρχουν ήδη. Όταν μιλάμε για δεδομένα από δορυφόρου, αυτά τα δεδομένα ήδη υπάρχουν. Θα θέλαμε λοιπόν να τα χρησιμοποιήσουμε με σωστό τρόπο, προκειμένου να ωφελήσουν τελικά και τον αγρότη και τα συστήματα διαχείρισης συνόρων και ελέγχου των συνόρων για να δούμε και τι γίνεται με τις πληρωμές. Το σύστημα λοιπόν πληρωμής ουσιαστικά θέλει να εξυπηρετήσει τελικά τον ε, Γιώργο για να υπάρξει αυτή η απλοποίηση με τη μείωση των προδιαγραφών. Και τέλος, να πω και δύο κουβέντε για αυτή την, την περιφερειοποίηση και την απλοποίηση. Όταν υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ, προφανώς ε, έχουμε και κράτη-μέλη τα οποία λένε θέλουν ε, να είναι πιο πολύ περιφερειακά τα συστήματα, μα όταν είναι περιφερειακά έχουν μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειε. Και αυτέ οι λεπτομέρειε προφανώ θα πρέπει να ενημερώνονται, να υποβάλλονται εκθέσει ε, όλα αυτά. Και θα πρέπει να υπάρξει μια σύνοψη εθνικό επίπεδο. Αν θέλουμε λοιπόν να προγραμματίζουμε το περιφερειακό επίπεδο, να υπάρχει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικά αναπεριφέρεια, αυτό αποτελεί μια δυνατότητα προφανώ. Και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κληθεί να εξετάσει το επίπεδο προγραμματισμού και σχεδιασμού που έχουν ορίσει τα κράτη-μέλη. Πολλά δεδομένα έχουμε ήδη σε επίπεδο κρατών μελών στους οργανισμούς τον κοιτώντας στους δείκτες για τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις. Τα πιο πολλά δεδομένα ήδη υφίστανται σε επίπεδο κρατών μελών. Προφανώς θα πρέπει να γίνει εξαγωγή από τα συστήματα πληροφορικής IT. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε λάβει υπόψη αυτά που ήδη είναι διαθέσιμα ως δεδομένα και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους τέσσερις εκπροσώπους ε, σήμερα των ε, οργανισμών γιατί πραγματικά μας αποδείξατε ότι έχετε πολύ αποτελεσματικά συστήματα και οργανισμούς πληρωμών και μπορούν να αποδώσουν. Και κάτι τελευταίο, η απόδοση να μην μπει α, καπάκι στις προηγούμενες προδιαγραφές, να αντικαταστήσει τις προηγούμενες προδιαγραφές. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, την πρόεδρο. Ευχαριστούμε την κυρία Μπόχμαν. Και να περάσουμε τώρα στον τελευταίο γύρο απαντήσεων των ε, προσκεκλημένων. Τέσσερα λεπτάκια θα σας δώσω για να απαντήσετε στις ερωτήσεις των συναδέλφων και σε αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θέλετε. Ο κ. Ζαμακόφσκι. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Ε, πάρα πολλές ερωτήσεις ετέθησαν και ελπίζω να μπορέσω να τις απαντήσω όλες. Η κυρία Σαντέρ. Πράγματι, εμείς ε, προσπαθήσουμε να επιτύχουμε την απλούστευση γιατί τη χρειαζόμαστε την απλούστευση εκτός από τον τομέα της πληροφορική που θέλουμε να τον επεκτείνουμε περισσότερο την, τον τηλεεντοπισμό, τον εντοπισμό εξ αλλά και πέρα από αυτό αναζητάμε απλουστεύσεις όσον αφορά την ανάλυση των διαδικασιών. Ο οργανισμός μας είναι αρκετά μεγάλος και τώρα πλέον πρέπει να ορίσουμε εκείνες τις διαδικασίες που υπάρχουν σε διάφορα επίπεδα, δηλαδή από τον δικαιούχο μέχρι την στιγμή της καταβολής των ποσών. Αυτή τη διαδικασία πρέπει να τη χαράξουμε και να την περιορίσουμε ή δυνατόν. Να δούμε κατά πόσον μπορούμε να κάνουμε κάποιες εξοικονομήσεις πρώτων και σε εξοικονόμηση χρόνου. Έτσι μπορούμε να γίνουμε και πιο αποτελεσματικοί σε επίπεδο Όσον αφορά τώρα ε, τον, ε, το θέμα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ενωσιακό παράγοντα, εμείς επιθυμούμε μεγαλύτερη ευελιξία για να μπορούμε την ευελιξία να την επιδείξουμε εκεί που πραγματικά πρέπει να το κάνουμε. Τα εθνικά μας όργανα δουλεύουν συστηματικά και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ε, τα ελεγκτικά αυτά όργανα είναι πολύ πιο περιοριστικά από ό,τι πιστεύουμε και νομίζω ότι έτσι μπορεί να υπάρξει μια καλή εφαρμογή του προγράμματος. Τώρα, πού ακριβώς ε, υπάρχουν ε, οι ουσιαστικές απλουστεύσεις. Ε, σωστά ετέθη αυτό το ερώτημα και θέλω να επισημάνω το εξής. Να επισημάνω κάτι που μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Μέχρι τώρα επεξεργαστήκαμε ένα μέτρο σε κεντρικό επίπεδο και μετά βλέπαμε κατά πόσο αυτό το μέτρο ήταν αποτελεσματικό σε επίπεδο δικαιούχου ή όχι. Δηλαδή, έχουμε εμείς μια λιγάκι διαφορετική κατάσταση, υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες έχουν ιδιαιτερότητες και αν η πολιτική διαμορφώνεται κεντρικά, αυτό οδηγεί στο ότι ορισμένες περιφέρειες επωφελούνται καλύτερα από άλλες. Η περιφερειοποίηση για μας συνεπάγεται και απλούστευση, διότι με τον τρόπο αυτό λαμβάνονται τα σωστά μέτρα ε, σε σωστό σημείο. Δεν θέλουμε κανέναν να αποκλείσουμε ε, και δεν θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ε, θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στις μικρές επιχειρήσεις που συνεπάγονται ε, οικολογική αξία και για τη βιοποικιλότητα και για πολλά άλλα. Τώρα, κατά πόσον αυτές οι διατάξεις μπορούν να εφαρμοστούν, ε, το πρώτο βήμα, η εφαρμογή του προγράμματος. Αυτό είναι δύσκολο, είναι δύσκολη αυτή η πρώτη φάση. Ε, τα προηγούμενα προγράμματα ήταν παρεμφερή. Τώρα όμως έχουμε κάτι το καινούριο, άρα δηλαδή μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά και πρέπει να έχουμε κάποια εμπειρία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Σε τελική ανάλυση αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προσφέρουμε μετρήσιμα αποτελέσματα, γιατί σε τελική ανάλυση αυτό θα μας προσφέρει ικανοποίηση. Ε, τα αποτελέσματα πρέπει να είναι ορατά, ε, πρέπει να μπορούν να εμφανίζονται στις στατιστικές. Όσον αφορά τους ελέγχους, τέθησαν πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Εάν λοιπόν υπήρχε η δυνατότητα να παρατηθούμε από ελέγχου, πολύ, καλά, πολύ ευχαρίστω το κάναμε αυτό. Γιατί πράγματι δεν είναι αλήθεια ότι αν υπάρχουν ε, περισσότεροι έλεγχοι τότε και ε, θα μειωθεί το ποσοστό ε, του σφάλματος. Ε, πρέπει λοιπόν να διορτηθούμε κατά πόσον οι έλεγχοι είναι απαραίτητοι και κατά πόσον ε, μπορούν να αποκαλύψουν παρατυπίες. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια εφαρμογή σε smartphone ε, που προκύπτει τώρα από τους επιτόπου ελέγχους. Όσον αφορά τον ορισμό του ενεργού γεωργού, ξέρετε ένας γεωργός που είναι ασφαλισμένο σε ειδικό ταμείο γεωργών. Αυτό το ταμείο αφορά γεωργούς ε, που έχουν μέχρι και ένα εκτάριο. Αυτός είναι ο ορισμός που δεχόμεθα για τον ενεργό γεωργό. Για το διαδίκτυο δεν έχουμε φόβο ε, για το διαδίκτυο. Ε, Του αντίον έχουμε συστήσει συμβουλευτικές επιχειρήσεις που βοηθούν τους γεωργούς. Αν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, ο γεωργός μπορεί να απευθυνθεί σε μια τέτοια εταιρεία. Και τελειώνοντας, το μοντέλο βεβαίως και πρέπει να τύχει επεξεργασίας. Το μοντέλο ανάλυσης ε, ε, χρειάζεται βελτιώσεων και με αυτό κλείνω την παρέμβασή μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, βλέπετε ότι μπορεί κανείς να μάθει ότι μπορεί να είναι σύντομος, γιατί ξέρετε ότι η καθυστέρησή σας είναι μόνο κατά ένα ή ενάμιση λεπτό. Ο κύριο Ριμπέιρο, ευχαριστώ πολύ για τι ερωτήσει. Ήταν πολλέ. θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ σε αυτέ που δεν απάντησα ακόμα. Η άποψή μα είναι ότι χρειαζόμαστε αποτελεσματική απλοποίηση και εδώ και πολλά χρόνια συζητούμε για την απλοποίηση και φαίνεται ότι πάντα ε, τελικά απλώ περιπλέκουμε τα πράγματα. Σε αυτό το νέο σύστημα όμως θα έχουμε απλοποίηση, αποτελεσματική απλοποίηση για τις εθνικές αρχές και για τους γεωργούς. Δεύτερη ερώτηση. Για τη συμμόρφωση. Είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα αυτό και παραδέχομαι ότι ορισμένες φορές ε, εκπλήσωμαι διότι οι χώρες που έχουν λιγότερη συμμόρφωση ζητούν μεγαλύτερη συμμόρφωση. Όσον αφορά την Πορτογαλία, στο δεύτερο πυλώνα έχουμε 65 με 70% συμμόρφωση στον πρώτο πυλώνα και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ίσως δεν επικεντρωνόμαστε στο σωστό ε, όσον αφορά τη συμμόρφωση, τα πιο αποτελεσματικά πράγματα ε, είναι αυτά τα οποία έχουν συγκεκριμένους στόχους και γίνεται διαχείριση βάσει αυτών. Για παράδειγμα, υπήρχε ένα πρόγραμμα για αμπελώνες, ε, το οποίο εφαρμόστηκε συνολικά στο για το δεύτερο πυλώνα και η διαχείριση γινόταν πλήρως με απλοποιημένο κόστος. Δηλαδή δεν γίνεται κάποιος ε, ειδικό έλεγχος και ξέρουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για τους ελέγχους και ήταν το πιο επιτυχές. Ε, έγινε και έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ιδιαίτερα επιτυχές. Ε, καταφέραμε να απλοποιήσουμε τον έλεγχο αυτό ως προς τη συμμόρφωση. Εμείς ε, υποστηρίζουμε τις πληρωμές και μετά η στήριξη παρέχεται αποτελεσματικά. Όταν ε, γίνονται πληρωμές ε, για στόχους και αποτελέσματα ε, επιτόπου. και όταν αυτοί που εργάζονται στην εκμετάλλευση γνωρίζουν ότι θα πρέπει ε, να έχουν αυτά τα αποτελέσματα για τα οποία έχουν δεσμευτεί, θα πρέπει να φροντίσουν να παρέχουν την υπηρεσία ή το προϊόν με το ε, χαμηλότερο δυνατό κόστος. Επομένως έτσι δεν έχουμε περισσότερες δαπάνες αλλά λιγότερες δαπάνες και ε, καταφέρουν όλοι να έχουν και μία πιο οικονομικά εύρωστη προσέγγιση. οι πιο αποτελεσματική έλεγχοι και τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα είναι αυτά τα οποία δεν βασίζονται σε συμμόρφωση ως προς τις δαπάνες. Ε, δεν ξέρω αν μιλούμε όλοι για το ίδιο πράγμα όταν εξετάζουμε τα θέματα της συμμόρφωσης στην Πορτογαλία και νομίζω ότι και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν θέματα που αφορούν τη συμμόρφωση ως προς τις δαπάνες ε, που δεν έχουν σχέση με τον τρόπο με τον οποίο δαπανούνται τα κονδύλια, αλλά έχουν σχέση με άλλα πράγματα. Ε, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεται ένα πρόγραμμα, για παράδειγμα. Θέλουμε λοιπόν να στηρίξουμε κάποιον για τον εξής απλό λόγο, διότι κατάφεραν να τηρήσουν τις απαιτήσεις ή θέλουμε να έχουμε μια καλή υπηρεσία η οποία να είναι κοινή ωφελία και να πληρώνουμε κάτι τέτοιο και να βασίζεται σε αυτό το σύστημα διαχείρισης. θα πρέπει να γίνεται και μετά στη συνέχεια επαλήθευση και έλεγχο ω προ τη συμμόρφωση. Όσον αφορά το κόστο τώρα, εδώ ισχύει το ίδιο. Νομίζω ότι εδώ και πάλι θέλουμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα. Θα υπάρχουν όμως ε, και κόστη για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, σε νέα συστήματα, επενδύσεις καινοτομία γενικότερα και φυσικά η αλλαγή αυτή θα επιφέρει κάποιο κόστος. Είναι άλλο να έχει κανείς κάποιο σύστημα στο οποίο θα μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τον έλεγχο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν έλεγχοι καθόλου. Απλώς θα γίνονται για συγκεκριμένες πτυχές, για τη χρήση της γης, για το είδος της καλλιέργειας. Δηλαδή, απτές ε, πτυχές, αυτό είναι ένα σκέλος του ελέγχου, το οποίο διαφέρει πλήρως από έναν έλεγχο στον οποίο αναλύουμε ε, άλλα έγγραφα που αφορούν ε, προϋπολογισμό. Είναι δύο διαφορετικά είδη ελέγχων αυτά. Και ε, στον πρώτο πυλώνα δεν εξετάζουμε πλέον τις δαπάνες, αλλά τους στόχους, τη χρήση της γης, τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένη η επιχείρηση κλπ. Αυτά θα έχουν τελείως διαφορετικό κόστος και μπορεί να γίνουν σε πολύ ε, σύντομο χρονικό διάστημα, ε, αντί να έχουμε παρακολούθηση για την κίνηση των ζώων, για παράδειγμα. Ο κύριος Στέλλα. Ευχαριστώ πολύ. Οι ερωτήσεις είναι αρκετές. Ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω σε όλες, κυρίως αυτές οι οποίες ε, απευθύνθηκαν σε μένα ε, από τους Ιταλούς Ευρωβουλευτές. Ε, στην Ιταλία υπάρχουν οι περιφέρειες, υπάρχει η περιοχή του Βένετο, η Τοσκάνη, η Εμίλια Ρωμάνια, το Πιεμόντε, το Τρέντο, το Μπολτζάνο, η, Λομβαρδία, 8 τον αριθμό που έχουν δικό τους οργανισμό πληρωμών. Οι άλλες που δεν έχουν οργανισμό πληρωμών ε, τις διαχειρίζεται ένας ε, οργανισμός ε, για τις ε, περιφέρειες που λέγεται Τζέα. Και υπάρχει και ο συντονισμός του Τζέα. Σε αυτή την περίπτωση απαντώ και στον κύριο Τζανρούσο. Τι γίνεται λοιπόν. Πολλές περιφέρειες που δεν έχουν δικό τους οργανισμό πληρωμών και αυτό είναι στοιχεία, δεν το λέω απλώς ε, για να επικρίνω, έχουν τελείως διαφορετικές επιδόσεις. Οι περιφέρειες που έχουν δικό τους οργανισμό πληρωμών έχει καλύτερες επιδόσεις. Ο τελευταίος οργανισμός πληρωμής που εγκρίθηκε στην Ιταλία είναι της Σαρδινίας και εκεί πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια μεγάλη όφηση ε, και θέλουν να είναι αυτόνομοι σε σχέση με ένα σύστημα το οποίο κατά πάσα πιθανότητα ε, με στοιχεία, με απτά στοιχεία δεν λειτουργεί όπως λειτουργούν οι άλλοι οργανισμοί πληρωμής. Εμείς ε, πράγματι συνεργαζόμαστε πολύ στενά με άλλες ε, περιφέρειες που δεν έχουν δικό τους οργανισμό πληρωμής και μας ζητούν ε, να τους δώσουμε τις δικές μας βέλτιστες πρακτικές και τι κάνουμε, συνεργαζόμαστε πραγματικά με τις περιφέρειες που μας το ζητούν. Δεν ξέρω εάν το εθνικό Ιταλικό σύστημα είναι έτοιμο για να αντιμετωπίσει αυτή την αλλαγή ε, νοοτροπίας. Ε, κατά πάσα πιθανότητα, εμείς ως ε, περιφέρεια του Βένοτο και ως οργανισμός πληρωμής του Βένοτα, από τεχνολογικής πλευράς ίσως θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Διότι εμείς προσπαθήσαμε να προβλέψουμε λίγο και να έχουμε και ένα όραμα για το τι μελγενέστε, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουν να δώσουν την ίδια απάντηση ε, και από πλευράς ε, του κεντρικού οργανισμού. Δεν ελέγχουμε εμείς την αλία ως οργανισμός πληρωμής, ε, λυπάμαι, αλλά η πρότασή σας ε, είναι κάτι που με βρίσκει και με ένα σύμφωνο, διότι σίγουρα θα μπορούσε να αποτελέσει μια επιπλέον ευκαιρία. Όταν συζητούμε απλούστευση όμως, και πρόκειται να γίνει κάτι, αφού έχουν αναλυθεί όλες οι διαδικασίες, πρέπει να γίνει. Και αν υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο πρέπει να το κάνω εγώ και ένα άλλο ποσοστό που πρέπει να το κάνει ο γεωργός, ε, τι πρέπει να κάνει ο οργανισμός πληρωμής. Πρέπει να προσπαθήσει να απλοποιήσει τη δική του τη δουλειά. Για να απλοποιήσει όμως τη δική του τη δουλειά δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρέσει αυτός κάτι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να εξαφανιστεί κάτι. Σημαίνει ότι πρέπει να είναι λιγότερα και αυτά που κάνει ο γεωργός. Εάν όμως ε, ε, επειδή είπαμε ότι υπάρχει το σύστημα το οποίο πρέπει να εφαρμόσουμε και τα πράγματα είναι περίπλοκο, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ο οργανισμός πληρωμής ή ο οργανισμός διαχείριση να αναλαμβάνει τμήμα των όσων θα έπρεπε να κάνει ο Γιώργος Έτσι είναι το σύστημα. Ε, να μειώνει ο άχθος, αλλά τελικά το κάνει κάποιος άλλος και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνει δημόσια διοίκηση. Εμείς έχουμε μία σειρά από εφαρμογές και τάμπλετ και πειραματιζόμαστε με πολύ καλά αποτελέσματα. Να μας δίνουν, για παράδειγμα, στοιχεία, να μας τα στέλνουν χωρίς να χρειάζεται να πάμε επί τόπου, να μας στέλνουν ασφαλείς φωτογραφίες με γεωγραφικές αναφορές για να μπορέσουμε να τα εντάξουμε στο σύστημά μας. Μπορεί ίσως να αυτή είναι η σωστή λύση. Εμείς χρησιμοποιούμε δορυφορικά στοιχεία και χρησιμοποιούμε και ό,τι άλλο υπάρχει διαθέσιμο από τεχνολογικής πλευράς. Αλλά πρέπει οι από μια αναλογική ε, αντίληψη πρέπει να περάσουν σε μια ψηφιακή αντίληψη. Και αυτό φυσικά πρέπει να ε, το υποστηρίζουμε κι εμείς, αλλιώς δεν θα φτάσουμε σε αυτό το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε. Όσον αφορά τώρα τις απάτες, ε, σίγουρα είναι πολύ σημαντικά αυτά. Εμείς κάνουμε πολλά προγράμματα με την Όλαφ, συνεργαζόμαστε, έχουμε ήδη κάνει τρία προγράμματα και είναι πολύ σημαντικά, αλλά αν θέλετε, συμβαίνουν. Δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό. Ορισμένε φορέ μα εκπλήσουν και εμά ε, και μπορεί να πρέπει να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι. Και υπάρχουν και άλλα αρκετά σύνθετα ζητήματα, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο στη διάθεσή μου. Ελπίζω να σα τα πω την επόμενη φορά, αν βρεθεί άλλη ευκαιρία. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη. Και εμεί σα ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο για να κλείσουμε. Ε, σήμερα λοιπόν ε, ακούστηκαν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Είμαι ευγνώμων και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστώ κυρία Σάντερ. Νομίζω ότι αυτά που δείξατε πραγματικά είναι καθοριστική σημασίας, ακόμα και αν ε, από τη δική μου την άποψη ε, ισχύει αυτό που σας είπα ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή από τη συμμόρφωση στην απόδοση. Νομίζω κανένας εκπρόσωπος εδώ ε, από τους οργανισμούς πληρωμών δεν λέει ότι δεν χρειαζόμαστε ελέγχους. Είναι απόλυτα σαφές ότι χρειαζόμαστε τους ελέγχους. Ε, ε κύριε Μπόχμαν, ε, νομίζω και εσείς είπατε ότι έχουμε καλά συστήματα και αυτά θα πρέπει να τα συνεχίσουμε. Έτσι λοιπόν όταν ε, μιλάμε για την ε, ε, απλούστευση, την απλοποίηση. Ε, νομίζω ε, αυτό που εννοούμε είναι να δει κανεί του ελέγχου, δηλαδή να δούμε κατά πόσον σε κάποιου διαπιστώνουμε ότι η έλεγχη αυτή είναι απαραίτητη. Νομίζω σε πολλέ περιπτώσει θα διερωτηθούμε με ποια μέσα είναι απαραίτητο να υπάρξουν αυτοί οι έλεγχοι. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις Ίσως θα πρέπει να αναζητηθούν κάποιες άλλες λύσεις αν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Και έτσι κατανοώ και την έννοια της ε, επικουρικότητας. Για μας ε, είναι εξίσου σημαντικό και νομίζω αυτό είναι σαφές ε, να δούμε λιγάκι τα ποσοστά ελέγχου και μπορούμε να τα περιορίσουμε εκεί όπου πιστεύουμε ότι το σύστημα λειτουργεί και ότι αν το αλλάξουμε δεν θα προκύψει τίποτα καλύτερο. Άρα δηλαδή με λίγα λόγια ευθύ εξ αρχή διαφάνεια σημαίνει ότι πρέπει να είναι απόλυτα σαφές τι και μέχρι ποιου βαθμού θα πρέπει να ελέγχεται και ε, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και το τι επιτυγχάνει ένα εθνικό κράτος. Αυτό όμως που ενδιαφέρει είναι να δούμε και τι ε, προκύπτει για μας, για τους οργανισμούς ε, πληρωμών. Νομίζω ότι πάνω σε αυτό έχουμε τις μεγαλύτερες δυσκολίες μας και εκεί ε, πολλές φορές ε, προβάλλει μια πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορούμε να ε, λειτουργήσουμε με σωστό τρόπο. Αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο. Ε, θα συνεχίσουμε να επισκεπτόμεθα τους ε, γεωργούς. Το θέμα είναι με ποια ένταση. Γιατί νομίζω ότι οι γεωργοί χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες και σε τελική ανάλυση έχουμε τον οργανισμό πληρωμών, ο οποίος έχει αρκετά μεγάλες επιτυχίες, η αντίδραση είναι πολύ θετική και νομίζω ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να τον συνεχίσουμε. Κατά τα άλλα, ε, υπάρχουν πάρα πολλές ε, ερωτήσεις ε, που ελπίζω να απαντήθηκαν όλες. Κάπως τα χάσα λίγο. Το θέμα είναι ε, κατά πόσο θα πρέπει να αλλάξουν το σύστημα. Ε, σε τελική ανάλυση... Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ε, ανάγκη ελέγχων ε, που θα πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί. και τα άλλα θέματα νομίζω ότι ε, άκουσα ότι απαντήθηκαν από τους αντέλφους. Αυτό που έχει σημασία και το είπε η κυρία Μπόχημαν είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά δεδομένα. Αυτό είναι σημαντικό και σωστό. Το θέμα είναι κατά πόσον τα θέματα αυτά είναι τα σωστά, αν θα πρέπει να χρειαζόμαστε άλλα στοιχεία στους ελέγχους. Και το είπατε και μόνοι σας, ε, ε, κύριε Μπόχιμαν, βεβαίω υπάρχει αυτό το τεράστιο υλικό των δεδομένων. Ε, θα πρέπει να το δούμε τι θα κάνουμε με την περιφερειοποίηση και το ερώτημα είναι ε, κατά πόσον μπορούμε να κάνουμε σχετικά με το να ξεκαθαρίζουμε ποια στοιχεία χρειαζόμαστε. Και νομίζω υπάρχουν πολλά θέματα που μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Και έτσι ολοκληρώσαμε την ε, ανταλλαγή απόψεων με τους οργανισμούς πληρωμών. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους εκπροσώπους των Αθηνικών οργανισμών που ήρθαν να μας μιλήσουν και τις επόμενες εβδομάδες που θα έχουμε τις διαπραγματεύσεις. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε τις ε, συζητήσεις μαζί σας ε, μέσω της γραπτής οδού και ενδεχομένω να παραμείνετε σε επαφή με του ε, εισηγητέ και του σκιώδει εισηγητέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μα αφήρασατε το χρόνο σήμερα για να συζητήσουμε τι επιπτώσει του νέου μοντέλου υλοποίηση. Μπορείτε λοιπόν να παραμείνετε στις θέσεις σας για να τελειώσουμε την σημερινή ημερησία διάταξη. Ε, έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών. Αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, θεωρούνται κεκριμένε οι αποφάσει. Στα 18 λοιπόν έχουμε τα διάφορα από πλευρά. Δεν έχω κάτι να σα αναφέρω. Δεν ξέρω αν εσεί κάτι έχετε να υποβάλλετε στα διάφορα. Αν όχι, να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίαση στο 19 είναι στις 17 Φεβρουαρίου στις 3 το απόγευμα. Τα λέμε λοιπόν και στις 18 Φεβρουαρίου θα έχουμε ε, ολόκληρη μέρα. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ ιδιαίτερους όλους όσους έμειναν μέχρι τέλους και σας εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό.